the president. Good evening, colleagues. If I could ask you to please... Καλησπέρα, συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε και Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ο πρόεδρος, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, έχει καθυστερήσει και ζητά συγγνώμη. Πολλοί είχαμε προβλήματα με τις πτήσεις. Η δικιά μου πτήση προσπάθησε δύο φορές να προσγειωθεί στη Βασιλεία και δεν τα κατάφερε, αλλά προσγειώθηκε στο Στρασβούργο. Οπότε είμαι εδώ αλλά προφανώς ε, και οι άλλοι συνάδελφοι δυσκολεύτηκαν και ζητάω την υπομονή σας γιατί μόλις μου έδωσαν τα χαρτιά επαναλαμβάνω τη συνεδρίαση που είχε διακοπεί στις 13 ε, Ιανουαρίου και θέλω να κάνω μια ανακοίνωση επευκαιρία της ημέρας μνήμης σήμερα θα ήθελα να τιμήσουμε τη μνήμη των Ιταλών και λοιπόν ε, θυμάτων ε, της εξόδου ε, των Ιταλών από την Ίστρια και των Δαλματών και των υπολείπων μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η υπεράσπιση της δημοκρατίας και της ανοχής και η καθημερινή μας προσήλαση στις ευρωπαϊκές αξίες είναι ο καλύτερος φόρος τιμής σε αυτά τα θύματα. Η μετάβαση από τα δύο αντιμαχόμενα μπλοκ σε μία ένωση ειρήνης δείχνει πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μία Ευρώπη η οποία θα έχει στην πρώτη θέση τον σεβασμό για τους πολίτες της. Σας παρακαλώ να σηκωθείτε για ένα λεπτό. Thank you. Σας ευχαριστώ. Να κάνω κάποιες ανακοινώσεις πριν περάσουμε στα διαδικαστικά. Ευχαριστώ. Ναι. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 29ης και 30ης Ιανουαρίου είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν σχόλια. Εάν όχι, τα πρακτικά εγκρίνονται. Περνάμε τώρα σε κάποιες άλλες ανακοινώσεις. Ξεκινάμε με την σύνθεση του Κοινοβουλίου μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου. Σύμφωνα και με την σχετική συμφωνία, οι έντολες των βουλευτών του Ηνωμένου Βασιλείου έληξαν στις 31 Ιανουαρίου 2020. Τα ονόματα των βουλευτών θα προσθεθούν στα σημερινά πρακτικά σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28 Ιουνίου 2018 και μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου στις 31 Ιανουαρίου, οι αρμόδιες αρχές 13 κρατών μελών μας κοινοποίησαν ε, την εκλογή 24 νέων βουλευτών από 1η Φεβρουαρίου 2020. Τα ονόματα και αυτών των βουλευτών θα περιληφθούν στα σημερινά πρακτικά. Το Κοινοβούλιο σημειώνει την εκλογή του. Καλωσορίζω του νέου συναδέλφου και επισημαίνω ότι θα καταλάβουν τις ε, έδρε του ε, στο Κοινοβούλιο και θα έχουν τα πλήρη δικαιώματα σύμφωνα με τον κανονισμό. Η επόμενη ανακοίνωση μετά από την ε, σύνθεσή του Κοινοβουλίου και των Επιτροπών που εγκρίθηκε στις 15 Ιανουαρίου έχω λάβει από τις πολιτικές ομάδες και τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές τους διορισμούς της Επιτροπές ε, του Κοινοβουλίου σήμερα με το άρθρο 209. Ο κατάλογος ε, των βουλευτών έχει δημοσιευτεί και θα προσθεθεί στα πρακτικά. Περνάμε τώρα στα διαδικαστικά. Κυρία Ομπρέ. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να επενθυμίσω τον εσωτερικό κανονισμό μετά το, με το, βάση το άρθρο 125 παράρτημα 7. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, βρίσκονται σε καθεστώς ε, μη νομιμότητας. Θα πρέπει κάθε 1η Ιανουαρίου να δημοσιεύουν την ε, δήλωση οικονομικών συμφερόντος. Κανένας όμως δεν το έχει κάνει. Αυτή η παράληψη δεν είναι τυχαία πολλοί ε, επίτροποι θα πρέπει να παρετηθούν από διάφορα διοικητικά συμβούλια αλλά αν κοιτάξουμε τις δηλώσεις οικονομικών συμφερών των διαφόρων ε, επιτρόπων, παραδείγματος χάρη του αρμόδιου επιτρόπου για τα ψηφιακά, έχει, ε, πάνω από, έχει μετοχές πολλές στην Amazon. δεν μπορεί λοιπόν να συνεχίσει να είναι επίτροπος με βάση αυτό. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σέβεται αυτή την υποχρέωση να δημοσιεύει τη, τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων επιτρόπων για να ξέρουμε τι ακριβώς παίζεται με βάση το χρήμα που έχει ο καθένας. Σας ευχαριστώ. Θα διαβαστούν αυτά στον Πρόεδρο. Θέλω να περάσω τώρα. Με συγχωρείτε, υπάρχει κι άλλο διαδικαστικό. Παρακαλώ, κυρία Σνάλφη. especial a El Salvador da delegação. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πρόκειται για την ε, αντιπροσωπεία ε, στο Σαλβαδόρ υπήρξαν πάρα πολλέ προσπάθειες εκφοβισμού, μια προσπάθεια εκβιασμού προς τους βουλευτές, διότι υπονομεύεται η ειρήνη και η σταθερότητα σε αυτή την χώρα ε, πόθηκε ε, η, ε, η απέτηση η Ευρώπη να μην ε, συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Συζητάμε τα διαδικαστικά. Εντάξει, σημαντικό αυτό, αλλά δεν είναι διαδικαστικό, οπότε περνάμε σε αλλαγές ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν αρκετά αιτήματα. Θέλω λοιπόν την υπομονή σας. Έχετε το τελικό σχέδιο μερίσιας διάταξη που ενέκριναν ενέκρινε διάσκεψη των Προέδρων στις 6 Φεβρουαρίου. Περνάμε λοιπόν στην τρίτη ομάδα. ID ζήτησε μια συζήτηση για τη δήλωση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και Κομισιών για ελευθερία λόγου και θρησκευτικό φονταμενταλισμό ως πέμπτο θέμα το απόγευμα της Τρίτης μετά την συζήτηση για τη νέα στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Θα δώσω τον λόγο στον ε, κύριο Ρεβιέ. Έχουμε την υπόθεση Μιλάν στη Γαλλία από το όνομα μιας ε, νεαρής γυναίκας 16 χρονών ε, που καταγγέλει το Ισλάμ και δέχτηκε απειλές θανάτου επειδή δημοσίευσε κάτι στο Instagram της. Κατηγορείται ότι Μίλησα με χιδέα λόγια εναντίον του Ισλάμ. Όμως έχουμε ελευθερία έκφρασης και μπορούμε να κριτικάρουμε ε, μία θρησκεία. Πολλές, πολύ λίγες φωνές ε, εκφράστηκαν στη Γαλλία εναντίον αυτής της, ε, αυτού του διωγμού. Αυτό δείχνει ακόμα περισσότερο την ε, δηλία των ελίτ μας, γιατί υποκύπτουν σε ένα Ισλάμο-κομμουνιστικό Ισλάμ. Δεν θέλουμε να μας επιβάλλουν την ταυτότητά μας και τον τρόπο ζωής μας. Φυσικά κάθε θρησκεία, το Ισλάμ, δεν οδηγεί πάντα στην τρομοκρατία, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπως το Σαρλί Εμπτό που δημιουργούν κάποια ερωτηματικά. Θέλει κάποιος να ε, μιλήσει κατά της πρότασης αυτής. Πρόεδρε. Πρέπει να υπερασπιστούμε την ελευθερία έκφρασης και αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία ε, μιλάει από μόνο του. Η πρότασή μας δεν είναι κατά τη συζήτηση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να θέσουμε τη συζήτηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Την Τετάρτη θα κάνουμε μια συζήτηση για να μιλήσουμε για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και του μίσου στην Ευρώπη. Θα θέλαμε να μιλήσουμε για την ελευθερία έκφρασης που θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ομαδικά. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση στα πλαίσια αυτή τη συζήτηση που είχαμε προβλέψει για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού και του μίσους. So λοιπόν το αίτημα για τροποποίηση για την συνημερήσια διάταξη της Τρίτης. Έχουμε ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πρόκειται για την ε, πρόταση του ID. Ε, Παρακαλώ να γνωρίζετε τι ψηφίζετε. Πρόκειται για την πρόσταση να αλλάξει η μερίσια διάταξη της Τρίτης ε, σε σχέση με, και να έχουμε μια δήλωση επιτροπής όσον αφορά την ελευθερία του λόγου. Είναι σαφές. Ωραία. Νομίζω ότι υπάρχει κάποια σύγχυση στο σώμα. Έχει προταθεί μια τροποποίηση για την ημερήσια διάταξη ε, της Τρίτης. Κύριε Περλαμέ, θέλετε αυτό να ε, συμπεριληφθεί σε ένα ε, σημείο το οποίο βρίσκεται ήδη στην ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ, διευκρινίσετε. Η πρότασή μας είναι εάν όλοι οι συνάδελφοι δεχθούν να ψηφίσουν, να συμπεριληφθεί το θέμα της ελευθερίας του λόγου στην συζήτηση η οποία θα διεξαχθεί την Τετάρτη. Ε, δέχομαι ε, την πρόταση αυτή. Αν είναι σαφές ότι πρόκειται για μια συζήτηση για την ελευθερία της έκφρασης σε σχέση με την ε, άνοδο του φονταμεναλισμού όσον αφορά την, αυτές τις ελευθερίες, δεχόμαστε δεν φαίνεται ότι έχει αποσυρθεί η πρόταση αυτή. Νομίζω ότι υπέρ του αιτήματο του κυρίου Μπελαμέ. Χρειάζεται να ψηφίσουμε για την πρόταση του κυρίου Μπελαμέ. Ωραία. Ε, θα γίνει τότε μια ονομαστική ψηφοφορία ή να ψηφίσουμε δια ανατάσεω τη χειρό. Όσοι είναι υπέρ τη πρόταση του κυρίου Μπελαμέ, παρακαλώ υπέρ. Θα διεξαχθεί η να ψηφισουμε δια ανατασσεω τη χειρο οσοι ειναι υπερ τη προταση ψηφοφορία αν θέλετε. Κατά παρακαλώ. Ε, θα πρέπει να γίνει επαλήθευση. Άρα λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έλεγχος, ηλεκτρονική επαλήθευση για την πρόταση αυτή. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψυχοφορίας, Η πρόταση του κυρίου Μπελαμέ απορρίπτεται. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση με τον κύριο Ριβιέ. Η, δική σας ε, πρόταση και αυτή έχει απορριφθεί μαζί με την πρόταση του κυρίου Μπελαμέ. Ε, θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Εάν η πρόταση του κυρίου Μπελαμέ είχε γίνει δεκτή, εμείς θα αποσύραμε το δικό μας αίτημα. Εφόσον ε, απορρίφθηκε, θα θέλαμε το δικό μας αίτημα να υποβληθεί σε ψηφοφορία. Εντάξει λοιπόν, θα έχουμε την πρόταση ε, τροποποίησης της ημερήσιας διάταξης της τρίτης διονομαστικής κλήσης. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. And the Πέραση ψηφοφορία. Ε, απορρίπτεται λοιπόν. Δεν θα υπάρξει αλλαγή. Υπάρχει μια άλλη πρόταση αλλαγής της ε, ημερήσιας διάταξης ε, την Τρίτη, ε, το Renew, σε σχέση με τη δήλωση του Συμβουλίου όσον αφορά τα περιοριστικά μέτρα εν ώψη της κατάστασης της Βενεζουέλας. Να συμπεριληφθεί ως δεύτερο θέμα στην ημερήσια διάταξη the Group. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Κάνιας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αντικείμενο αυτή τη πρόταση σχετίζεται με τη μία εκπλήρωση εκ μέρου τη Ισπανική κυβέρνηση τη ε, απόφαση 2064 ε, σαν αφορά με την επιβολή κυρώσεων στο καθεστώ του κυρίου Μαδούρα. Στι 19 Ιανουαρίου ε, η νόμιμη κυβέρνηση παρέμεινε 14 ώρες σε ισπανικό έδαφος ε, και τελικά το Κοινοβούλιο ενέκρινε κάποιες ε, κυρώσεις. Ωστόσο υπήρξαν έξι διαφορετικές εκδοχές αυτών των κυρώσεων. Η παραβίαση του διεθνούς δικαίου έγινε αφού ο Χουάν ε, Γκουαϊντό ζήτησε να σκληρινθούν οι κυρώσεις κατά του Μαδούρο. Εμείς ζητούμε να δεξιθεί μια συζήτηση ούτως ώστε να υπάρξουν εξηγήσεις εκ μέρους της πανικής Κυβέρνησης γιατί μόνο οι χώρες ε, μέλη που είναι οι χώρε μέλη επιφορτισμένε να επιβάλλουν αυτέ τι κυρώσει εφόσον έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Δεν είναι δυνατόν ε, να, υπάρχει ατιμορρησία στις περιπτώσεις αυτές. Συγγνώμη, μιλάτε υπερβολικά γρήγορα. Και παρακαλώ να γίνει με ονομαστική ψηφοφορία. Είναι κάποιος κατά αυτής της πρότασης. Ο κύριος Μόρεν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το σώμα για να επιτεθούμε στην Ισπανική κυβέρνηση. Γιατί κύριε Κάνια, το αίτημά σας ανταποκρίνεται μόνο σε μεροπτικά και κομματικά συμφέροντα και δεν ταιριάζει σε αυτό το σώμα. Η Ισπανική κυβέρνηση επανέλαβε εξ αρχής τη δέσμευσή της να συμφωνήσει με τη γραμμή της Ευρώπης όσον αφορά τη Βενεζουέλα. Ε, ε, και θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ότι είναι η Επιτροπή, αυτή η οποία επανέλαβε κατ' επανάληψη ότι οι, τις κυρώσεις θα πρέπει να τις επιβάλλουν οι χώρες μέλη. Δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να συνεισφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην κατάσταση αυτή παρά μόνο να υπερασπιστεί τα δικά του να υπερασπιστούν ορισμένα τα δικά τους κομματικά συμφέροντα. Ευχαριστώ πολύ. Υπέρ της ε, πρότασης να αλλάξει η μερίσια διάταξη, παρακαλώ. Κατά ε, να γίνει έλεγχος. Παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Άρα θα αλλάξει η μερίσια διάταξη ε, σε σχέση με τη δήλωση αυτή του Συμβουλίου και της Επιτροπής θα συμπεριληφθεί ως δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης την Τρίτη. Τώρα θα περάσουμε στην ε, Τετάρτη και έχουμε εδώ δύο ομάδες που υπέβαλαν κάποιες ε, προτάσεις. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι οι πράσινοι ζήτησαν ε, όσον αφορά, ε, να γίνει ψηφοφορία όσον αφορά την ολοκλήρωση της ε, συμφωνίας με το ελεύθερο εμπορίου με το Βιετνάμ. και να συμπεριληφθεί και, το, και η ψηφοφορία για το συνοδευτικό ψήφισμα. να παραλυφθούν αυτά από την ημερήσια διάταξη. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Μορέλ. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητάμε να αναβληθεί η ψηφοφορία, γιατί το κείμενο για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου, αλλά και το ε, κείμενο για την προστασία των επενδύσεων, είναι ενάντιο σε αυτό που ψηφίσαμε πριν από λίγες εβδομάδες για την κλιματική επίγουσα ανάγκη και για τη νέα πράσινη συμφωνία. Ε, είναι μια συμφωνία που δεν μπορεί να εκτελεστεί, δεν είναι ούτε δεσμευτική, έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι προβληματικό. Θα ήθελα όλοι οι συνάδελφοι, πέρα από τις πολιτικές του ευαισθησίες, να καταλάβουν τι μας, λένε, μας λέει η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων και πολλές ε, ΜΚΟ ευρωπαϊκές που μας κρούν τον κόδωνα για την κατάσταση των ε, εργασιακών δικαιωμάτων, συνδικαλιστικές ελευθερίες στο Βιετνάμ, δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε αόριστες ε, υποσχέσεις από την κυβέρνηση του Βιετνάμ. Θέλουμε εγγύησεις, θέλουμε απτά πράγματα. Δεν μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε, γι' αυτό ακριβώς ζητούμε την αναβολή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαμπέρ. Όχι, η κυρία Κέλλερ. Διορθώνω, λέει η πρόεδρος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει στην, στο ψήφισμα για την Πράσινη Συμφωνία φέτος να υπάρχουν δεσμευτικές διατάξεις και κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίσης, το Κοινοβούλιο που πρόσφατα εξελέγει είπε ότι οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης είναι βασικό στοιχείο της σημερισίας διάταξης. Είναι η πρώτη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου η οποία ε, τίθεται σε ισχύ με αυτή την Επιτροπή. Η συμφωνία αυτή όμω ε, διαπραγματεύτηκε χωρί αυτή τη δέσμευση. Πριν ζητήσει κάτι τέτοιο ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πριν ζητήσει δηλαδή τέτοιε δεσμευτικές διατάξει για το κεφάλαιο βιώσιμη ανάπτυξη. Τον Ιανουάριο το Κοινοβούλιο ψήφισε μία έκθεση για την απλούστευση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ένταξη σε όλε τι πολιτικέ. Δυστυχώ δεν έχουν ενταχθεί στην Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου με το Βιετνάμ. Γιατί βλέπουμε όλε τι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπορούμε να φανταστούμε, στο Βιετνάμ. Ε, γι' αυτό ζητάμε μία δέσμευση σαφή από την κυβέρνηση του Βιετνάμ ότι θέλουν πραγματικά να βελτιώσουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει όμω και γι' αυτό ακριβώ πιστεύουμε ότι πρέπει να διορθωθεί η κατάσταση. Χρειαζόμαστε περισσότερε δεσμεύσει και από την Κομισιόν και από την κυβέρνηση του Βιετνάμ. Γι' αυτό ζητούμε λοιπόν την αναβολή τη ε, ψηφοφορία ε, του κειμένου αυτού. Ο κ. Μπουρζουά, ο εισηγητή. μικρόφωνο. Έχω χάσει τη φωνή μου. Θα προσπαθήσω να είμαι ξεκάθαρο όμω. Εγώ σα. Καλό συνάδελφοι, κάνω έκκληση να μην αναβάλουμε ούτε τη συζήτηση ούτε την ψηφοφορία. Υπάρχει πρόταση στην ε, Επιτροπή για αναβολή. Ε, όμως ε, ψηφοφορία ψηφίσαμε και δεν πέρασε κάτι τέτοιο. Αποφασίσαμε να υπάρξει ένα συμβασμό, να παρακολουθήσουμε περισσότερο την εφαρμογή των δύο συμφωνιών, που είναι και η κλασική πρακτική του ILO. Να ζητήσουμε επίση περισσότερε δεσμεύσει από τι βιετναμεζικέ αρχέ. Και έτσι έκαναν. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τη επικύρωση της σύμβασης του ILO, το έκαναν. Και αυτό είναι προηγούμενο. στην κοινή επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Βιετνάμ ε, θα υπάρχει, συμφωνήσαμε ότι θα υπάρχει συμφωνία, συμφωνήσαμε συγγνώμη, θα υπάρχει παρακολούθηση των δύο συμφωνιών. Και το Κοινοβούλιο μας θα εμπλακεί ε, στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με το Βιετνάμ και επίσης τι άλλο έκαναν. Υπάρχει ανεξαρτησία των οργανώσεων που συμμετέχουν στις ε, εσωτερικές συμβουλευτικές ομάδες. Είναι θέμα αξιοπιστίας. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα βέβαια που διακυβεύονται. Συνάδελφοι, θα ψηφίσουμε καταρχάς για την πρόσθεση της ΓΟΕ που σημαίνει αναβολή και θα ψηφίσουμε με ονομαστική ψηφοφορία για την αναβολή που ζητάει η Γκουε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίσουμε τώρα για την πρόταση που σας παρουσίασε η κυρία Κέλλερ. Να αναβάλουμε τις δύο εκθέσεις με ονομαστική κλίση. Ψηφίσουμε πάλι. Κλείνουμε την ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Δεν θα γίνει καμία αλλαγή λοιπόν. Και προνάμε σε ένα άλλο σημείο για την Τετάρτη. Η ομάδα του ΕΛΚ ζήτησε μία συζήτηση σε ένα ε, προφορικό ερώτημα για ίντερνετ για τα παιδιά να προστεθεί το απόγευμα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Όλμπριχτ για να αιτιολογήσει το αίτημα της, ε, του ΕΛΚ. Εκ μέρους του ΕΛΚ θα ήθελα να ζητήσω να προσθέσουμε στην ατζέντα μας το προφορικό ερώτημα το ίντερνετ, ένα καλύτερο ίντερνετ για τα παιδιά. Στις 11 Φεβρουαρίου έχουμε τη μέρα του ασφαλούς ίντερνετ. Ξεκίνησε το 2004 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτή η μέρα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια δραστηριότητα για να προωθήσουμε ασφαλή πρόσβαση των παιδιών στο ίντερνετ. Γι' αυτό μαζί με του συναδέλφου πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Όχι μόνο εμεί οι πολιτικοί, είναι σημαντικό και οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτέ γενικά να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να μιλήσουμε για αυτή την ημερίδα μάλλον της, ε, του ασφαλούς ίντερνετ για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Ποιο θέλει να μιλήσει κατά? Όχι, δεν υπάρχει κανένα. Πρέπει να ψηφίσουμε. Ας το ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση. Ούτως ή άλλως είναι στην ατζέντα, έχει μπει. Πέρας προφορίας. Υιοθετείτε. Αυτό το σημείο θα προσθεθεί ως τελευταίο σημείο στην μερίσια διάταξη της Τετάρτης. Καλύτερο ίντερνετ για τα παιδιά. Ευχαριστώ. Και περνάμε σε ένα άλλο σημείο από τους πράσινους CFA που ζήτησε η, μια δήλωση τη Επιτροπή για την παρέμβαση τεσσάρων κρατών μελών σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση τη πολιτική ανταγωνισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό να προσθεθεί ω έκτο σημείο το απόγευμα. Θα δώσω το λόγο στον Μισελ Λαμπέρ για να αιτιολογήσει το, αυτό που ζητούν οι πράσινοι. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριοι συνάδελφοι, ε, το, στις 4 Φεβρουαρίου ε, τέσσερα μέλη, η Γαλλία, η Πολωνία, η Γερμανία και η Πολωνία ε, υπέγραψαν μία δήλωση ε, καλώντας τον ε, ε, Επίτροπο κ. Βασταγκέρ να αναθεωρήσει την πολιτική του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η πολιτική ανταγωνισμού εμπίπτει αποκλειστικά στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύω ότι είναι απολύτως, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να, το Κοινοβούλιο να αποφανθεί επί του θέματος αυτό, γιατί εμείς ε, θα πρέπει να συνεισφέρουμε εδώ, αλλά θεωρώ ότι το ύφος της ε, επιστολής τελικά δικαιολογεί και μία συζήτηση με τον ε, Επίτροπο. Γι' αυτό θα ήθελα να σας καλέσω να γίνει η συζήτηση αυτή την Τετάρτη. Ποιος είναι κατά της ε, ε, πρότασης. Ποιο θέλει να μιλήσει μάλλον, συγγνώμη, κατά της πρότασης αυτής. Ε, ναι, πιστεύω ότι ο κύριος Λάμπερτ έχει δίκιο. Αυτό το κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφανθεί σε σχέση με την πολιτική ανταγωνισμού. Ε, καθώς και σε άλλες συζητήσεις όσον αφορά την αναθεώρηση των κρατικών ενισχύσεων. Αλλά θα πρέπει αυτό να γίνει μέσα από τα επίσημα κανάλια. Την προσεχή εβδομάδα η Επιτροπή Εμπορικών Υποθέσεων θα κάνει την ψηφοφορία για εμπορικά θέματα και κάνει τις πραγματεύσεις ούτως ώστε η έκθεση αυτή να ψηφιστεί το Μάρτιο. Ε, γι' αυτό δεν βλέπω λόγους ε, να καθυστερεί η συζήτηση αυτή τη βδομάδα. Γιατί το κείμενο του συμβασμού θα μπορέσει, όπως σας είπα, να ψηφιστεί ενδεχομένω ε, την προσεχή εβδομάδα στην Επιτροπή. Ποιοι είναι υπέρ της ε, προταθής τροποποίησης στην ημερήσια διάταξη. Παρακαλώ. Κατά αποχές απορρίπτεται η ημερήσια διάταξη παραμένει ως έχει. Τέλος, ε, όσον αφορά την ε, Πέμπτη, ε, η ΚΟΕ ζήτησε μια δήλωση της Επιτροπής για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών σε εμπορικές σχέσεις να προσθεθεί ως πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Άρα στην περίπτωση αυτή θα ξεκινούσε σε 9 η συνεδρίαση. Σε λίγες εβδομάδες ε, θα υπογράψουμε μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την ε, κυβέρνηση του Τραμπ. Διαπραγματευόμαστε για ελεύθερο εμπόριο, για χλωριωμένα κοτόπουλα, κρέας με ορμόνες, ε, προϊόντα της Μονσάντο κτλ. Υποβαθμίζεται λοιπόν εδώ πέρα το περιβάλλον, η δημόσια υγεία και η υγεία των ζώων. Και είναι εις βάρος των Ευρωπαίων αγροτών. Οι Βρυξέλλες διαπραγματεύονται χωρίς άδεια από τα κράτη-μέλη. Το Συμβούλιο δεν έχει δώσει εντολή για να γίνει διαπραγμάτευση για γεωργικά προϊόντα με τη ΣΥΠΑ και επιπλέον το Κοινοβούλιο αυτό σύμφωνα με την Συμφωνία των Παρισίων έχει θέσει ως απαραίτητη προϋπόθεση να γίνει σεβαστή αυτή η συμφωνία στις μελλοντικέ εμπορικές διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, την στήριξή σας για μια κατεπίγουσα συζήτηση για τις εμπορικές ε, συνομιλίες με τις ΗΠΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Είναι κάποιος κατά αυτής της πρότασης. Παρακαλώ. Να ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όλοι βεβαίως ανησυχούμε για τις σχέσεις ε, με τις ΗΠΑ, πρέπει να τις παρακολουθούμε εκ του σύνεγγης, αλλά με σωστό τρόπο. Γι' αυτό έχουμε προσκαλέσει τον επόμενη εβδομάδα τον Επίτροπο Χόγκαν στην ε, Επιτροπή Ίντα και μετά βεβαίως θα το συζητήσουμε στην Ολομέλεια. Αλλά πρώτα απ' όλα ας κάνουν τη δουλειά τους οι Επιτροπές. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τίθεται σε ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. και πέρασε. Απορρίπτεται. Οπότε η μερική διαταξή παραμένει ως έχει. Η ομάδα του ΕΛΚ ζήτησε να προσθεθεί μια συζήτηση για την προφορική ερώτηση για τη στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο το πρωινό της Πέμπτης. Α, πρέπει να σας πω ότι αυτό σημαίνει ότι θα ξεκινήσει η συνεδρίαση 9 η ώρα το πρωί. Και δίνω τον λόγο στον κύριο Λίντς για να υποβάλει το αίτημα εξ ονόματος του ΕΛΚ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο θα παρουσιαστεί τέλος Μαρτίου από την Κομισιόν. Επηρεάζονται από αυτή η στρατηγική η Γεωργή και η Ήπεθρος. Γι' αυτό το ΕΛΚ θεωρεί απολύτως απαραίτητο να συζητηθεί ο κεντρικός ρόλος της γεωργίας πριν από τη δημοσίευση της στρατηγικής. Μόνο έτσι θα μπορέσει να οριστικοποιηθεί η στάση του Κοινοβουλίου για ζητήματα όπως η χρηματοδότηση, η ανταγωνιστικότητα και η σχέση με την ΚΑΠ. Για τον λόγο αυτό η ομάδα του ΕΛΚ ζητά αλλαγή της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το άρθρο 158. Ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Είναι κάποιο κατά αυτή τη πρότασης. Όχι. Λοιπόν, τι θέση ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Όπως είπα, οι συνεδρίες θα ξεκινήσει στις 9 και προστίθεται το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Τελευταία πρόταση για αλλαγή της ημερήσια διάταξης την Πέμπτη είναι από την ομάδα Renew. Ζήτησαν η συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τον κορονοϊό να αφαιρεθεί από την ημερήσια διάταξη. Δίνω τον λόγο στον κύριο Χάιτεμα για να υποβάλει το αίτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, ο κορονοϊός είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, αλλά για την ομάδα μας ε, δεν είναι το σωστό θέμα για τα κατεπήγοντα. Τα κατεπήγοντα είναι για κάτι το οποίο αφορά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η κατάσταση αυτή εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα, οπότε είναι δύσκολο να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Οπότε κινδυνεύουμε να πατρονάρουμε τους άλλους ενώ θα έπρεπε να συντονιζόμαστε με τις άλλες χώρες για να αποτρέψουμε την διάδοση του ιού. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να βγάλουμε αυτό το θέμα από τα κατεπήγοντα. Σας ευχαριστώ. Κάποιος ε, θέλει να τοποθετηθεί κατά. Παρακαλώ. Ναι, κυρία Πρόεδρε, θα αναφερθώ σε αυτά τα οποία είπε ο κύριος Χάουτεμα ότι υπάρχει ανησυχία ε, δεδομένου του ότι οι εξελίξει είναι πάρα πολύ γρήγορε και οι πολίτε ανησυχούν. σω χρειαστεί μια ευρύτερη συζήτηση για το θέμα αυτό αντί να το βγάλουμε από την ημερήσια διάταξη. Δεδομένου του ότι οι εξελίξει και επί τόπου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι τόσο γρήγορες, προτείνω να γίνει μια συζήτηση χωρίς ψήφισμα για το θέμα του κορονοϊού, τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια συντονισμένη ευρωπαϊκή αντίδραση. Τετάρτη απόγευμα επί τη ευκαιρία. Μάλιστα. Ε, είχαμε φτάσει την Πέμπτη, οπότε θέλετε να ξαναπάει Τετάρτη απόγευμα. Ε, να ρωτήσω τον κύριο Χάλτομα τι άποψη έχει. Εξαιρετική ιδέα. Συμφωνείτε όλοι. Είναι εξαιρετική ιδέα. Πρέπει να... Ωραία τίθεται σε ψηφοφορία. Όσοι είναι υπέρ του να γίνει αυτή η συζήτηση την Τετάρτη. Κατά. Αποχές. Ωραία. Θα γίνει λοιπόν την Τετάρτη όπου θα έχουμε αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Οπότε αυτή είναι η ημερήσια διάταξη. Καλησπέρα σας. Με συγχωρείτε υπάρχει κάποιο διαδικαστικό κύριε Καστάλτο. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Άρθρο 3, 5, 6, 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του άρθρου 158 του δικού μας κανονισμού. Θέλω να ενημερώσω τους συναδέλφους για την σοβαρότατη κατάσταση που υπάρχει ε, για ένα άτομο Αιγύπτιο που, χρησιμο, που χρησιμοποίησε το Erasmus Mundus. Ε, φοιτητή στην Ιταλία που τον απήγαν και τον βασάνισαν. Βρέθηκε 120 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, φάνηκε ότι έχει υποστεί βία, τον, συνέλαβαν και ο Τζούλιο Ρετζένι επίσης ε, είχε την ίδια τύχη. Θα ήθελα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δράσουν και να παρακολουθήσουν τις, καταστάσεις, τις περιπτώσεις αυτές με φοβερή προσοχή και να προσθέσω μια συζήτηση για το θέμα αυτό. Κύριε Καστάλτο, παρακαλώ. Δεν θα πρέπει να σε εξηγήσω τους εσωτερικούς μας κανόνες. Θα μπορούσε αυτό να τεθεί ε, ως σημείο ε, στις ομιλίες ενός λεπτού. Όχι να το θέσετε σαν διαδικαστικό. Δεν είναι σωστό αυτό. Arvoisat kollegat, eh, Συνάδελφοι, θα ήθελα να συνεχίσουμε τώρα. Αφού υιοθετήσαμε την μερίσια διάταξή μας, να περάσουμε στις ε, συζητήσεις. Παρακαλώ, αποχωρήσετε πολύ ήρεμα, ούτως ώστε να συνεχίσουμε τις ε, εργασίες ε, της Ολομέλειας τώρα που καθορίσαμε και την ημερήσια διάταξή μας. Το πρώτο σημείο της μερικής διάταξης είναι η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η διαδικασία Catch the Eye και η διαδικασία της μπλε κάρτας ισχύουν και παρουσιάζονται με τον κλασικό τρόπο εγγραφή ή με το ηλεκτρονικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ζητήσετε να συμμετάσχετε σε αυτέ τι διαδικασίε. Εάν χρειάζεστε οδηγίε, μπορείτε να τι ζητήσετε στην είσοδο τη Ολομέλεια. Και τώρα θα περάσω στα φιλανδικά. Η συζήτηση λοιπόν αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση της οικονομικής διακυβέρνησης. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο Πάολο Τζαντιλόνι, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω την ανακοίνωση που υιοθετήσαμε πριν από πέντε ακριβώς ημέρες. Με αυτόν τον τρόπο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το πρώτο που ξεκινάει τη συζήτηση πάνω στο six-pack και στο two-pack και γενικότερα πάνω στο σύστημα και στους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησής μας. Οι στόχοι της συζήτηση είναι ξεκάθαροι. Από τη μία θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη σταθερότητά μας και θα πρέπει κανένα να το αμφισβητεί αυτό και από την άλλη θα πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη εκ νέου. Η ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνει μια σωστή και ειλικρινή αξιολόγηση της λειτουργίας αυτών των κανόνων τα τελευταία δέκα χρόνια. Οι κανόνες αυτοί δημιουργήθηκαν λόγω της βαθιάς οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Και μετά από 10 χρόνια νομίζω ότι πια πρέπει και μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα για το πώς, για το πώς λειτουργήσαν και τι αποτελέσματα έδωσαν αυτοί οι κανόνες. Έχουμε καλά αποτελέσματα νομίζω, γιατί υπάρχει καλύτερο συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών και σε επίπεδο χρόνου και σε επίπεδο περιεχομένου μεταξύ των κρατών μελών μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της διαδικασίας επιτήρησης. Δεύτερον, μπορέσαμε να μειώσουμε τα ελλείμματά μας σε σχέση με το ΑΕΠ. Το 2011 μόνο τρεις χώρες σέβονταν τους κανόνες για το λόγο ελλείμματος ως προς το ΑΕΠ. Και με βάση την τελευταία αξιολόγηση που κάναμε, δεν υπάρχει καμία χώρα η οποία δεν σέβεται πια αυτόν τον κανόνα. Τρίτον, όλα τα κρατη τα οποία λαμβάνουν οικονομική βοήθεια ή έλαβαν οικονομική βοήθεια, επέστρεψαν στις αγορές. Ακόμα και αν έχουν δυσκολίες και τεράστιες δυσκολίες σε κοινωνικό επίπεδο. Τουλάχιστον όμως είναι πάλι πίσω στις αγορές. Έχουμε και κάποια μεικτά αποτελέσματα μετά από 10 χρόνια λειτουργία αυτών των κανόνων. Καταρχά. έχουμε τη μείωση του χρέους. Ναι, μειώθηκε το χρέος. Από το 90% κατά μέσο όρο στο 80% κατά μέσο όρο. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι αν λάβουμε υπόψη μας και άλλους ε, οικονομικούς παίκτες, ε, όπου ας πούμε οι Αμερικάνοι είναι στο 115% ενώ οι Ιαπωνέοι στο 240%. Σε αυτή τη μέση μείωση όμως δεν λαμβάνουμε υπόψη μας το υψηλό επίπεδο χρέους που έχουν ορισμένες χώρες ακόμα. Μικτά αποτελέσματα και λόγω της περιπλοκότητας των κανόνων αυτών. περιπλοκότητα ίσως είναι και ένας έξυπνος τρόπος για να αντιμετωπίσει κανείς τα προβλήματα. Αλλά αν οι περιπλοκές αυτές είναι υπερβολικές, τελικά δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Και τα κρατημέλη και οι ενδιαφερόμενοι δεν ενδιαφέρονται πια και δεν εμπιστεύονται πια αυτούς τους κανόνες. Ένα τρίτο επίπεδο είναι οι ελλείψεις που έχουμε. Καταρχάς, μειώσαμε τις δημόσιες επενδύσεις μας. Οι δημόσιες επενδύσεις μας δεν είναι πια στο επίπεδο που ήταν πριν από 20 χρόνια. Επίσης, δεν μπορέσαμε να μειώσουμε τα πλεονάσματα σε χώρες που έχουν υψηλά πλεονάσματα. Και τρίτον, γιατί είχαμε προκυκλικές δημοσιονομικές πολιτικές αυτή την περίοδο. Και τώρα με την νομισματική πολιτική είμαστε στο κατώτατο επίπεδο. Αν δεν μπορούμε να έχουμε αντικυκλικές πολιτικές, αυτό δημιουργεί περιορισμούς στη γενική οικονομική μας κατάσταση. Επομένως, έχουμε και καλά αποτελέσματα και μεικτά αποτελέσματα και ελλείψεις και προβλήματα δηλαδή. Τώρα, τι μελιγενέστε. Νομίζω ότι ο κόσμος μας σήμερα είναι πολύ διαφορετικός, οικονομικός πώς, από αυτό 10 χρόνια πριν. Μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τη βαθιά κρίση. Είχαμε διάφορα χρόνια σταθερή ανάπτυξης σε όλα τα κράτη-μέλη. Εδώ και ένα-δύο χρόνια έχει μειωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης. και η εικόνα για τα επόμενα χρόνια χαρακτηρίζεται από βεβαιότητα. Για εσωτερικούς λόγους, το τελευταίο τρίμηνο πέρυσι, του 19 δηλαδή, είδαμε κακά αποτελέσματα σε ορισμένες σημαντικές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχουμε όμως και αβεβαιότητα λόγω εξωτερικών ε, συνθήκων, ε, εμπορικές ε, σχέσεις, προβληματικές, το Brexit που είναι ανοιχτό θέμα ακόμα και τις συνέπειες του κοροναϊού. Αλλά φυσικά είναι πολύ νωρίς να τις αξιολογήσουμε. Αλλά βεβαίως συνεισφέρουν και συνάδουν και επιτείνουν αυτή την αβεβαιότητα. Σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς λοιπόν χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε μία παρατεταμένη ύφεση. Δηλαδή να έχουμε ε, χαμηλή ανάπτυξη, χαμηλό πληθωρισμό, χαμηλά επιτόκια. Αυτό μπορεί να μην συνάδει με τις στρατηγικές που έχουμε στην πράσινη μετάβαση και στην ψηφιακή μετάβαση. Γι' αυτούς τους λόγους ανοίγουμε μία συζήτηση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα καθορίσουμε το πεδίο αυτής της συζήτησης τους επόμενους ε, μήνες. Θέλω να τονίσω δύο βασικά πράγματα. Πρώτη λέξη κλειδί είναι οι επενδύσεις. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να διευκολύνουμε τις επενδύσεις. Κυρίως εκείνες που συνδέονται με τη στρατηγική της πράσινης ε, συμφωνίας που η πρόεδρος Φόντρα Λάιεν λέει ότι είναι η νέα στρατηγική μας για την ανάπτυξη. Και η δεύτερη λέξη κλειδί είναι απλούστευση. Απλούστευση των κανόνων. Όταν προωθούμε την απλούστευση των κανόνων, σημαίνει ότι ο κόσμος πείθεται για αυτούς τους κανόνες. Αν διευκολύνουμε τις επενδύσεις και αν απλουστεύσουμε τους κανόνες, θα μπορέσουμε να σταθούμε ενωμένοι σε αραγές μέτωπο είναι κάτι που πρέπει να μας βρει όλους μαζί προκειμένου να βρούμε λύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Επίτροπε, κύριε Τζεντιλόνι. Τώρα, εκ μέρου του ΕΛΚ, ο κύριο Φέρμπερ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης περιλαμβάνει πολλές ευφύς και σωστές παρατηρήσεις όσον αφορά ε, τα, τα, μη λειτουργικά σημεία του συμφώνου αυτού. Οι κανόνες είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι, δεν είναι διαφανείς. Ε, ε, καμιά φορά είναι προκυκλικές όσον αφορά την επίπτωσή τους και βεβαίω έχουν και θετικέ πτυχές. Τώρα έχουμε μια φάση ανάπτυξης ε, πίσω μας. Αυτό δεν συνέβαλε ούτω ώστε το έλλειμμα να μειωθεί σημαντικά. Τα συμπεράσματα τα οποία, στα οποία καταλήγει η Επιτροπή από τις διαβουλεύσεις σε σχέση με αυτές τις ε, διαπιστώσεις δεν σχετίζονται όμως ιδιαίτερα με τα προβλήματα που περιγράψαμε. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν έχει προβλήματα ευελιξίας. Ήδη η προηγούμενη Επιτροπή ε, όσον αφορά ε, τις ευελιξίες έκανε ότι, ε, την ευελιξία όσον αφορά ό,τι περνούσε από το χέρι της. Οι κανόνες δεν θα πρέπει να γίνουν πιο ευέλικτοι, αλλά θα πρέπει να εφαρμοστούν. Εάν έχουμε το πρόβλημα της υψηλής υπερχρέωσης και θέλουμε να το προσεγγίσουμε αποτελεσματικά, δεν έχει κανένα νόημα ορισμένες ε, δαπάνες να τις, βάζουμε, να τις ε, εξαιρούμε. Αυτό θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Θα ήθελα να πω ξεκάθαρα, ε, το χρέος είναι χρέος. Οποιαδήποτε μορφή νέου χρέους ε, ζημιώνει την, ε, το θέμα του χρέους ε, ανεξάρτητα από το κατά πόσο με τον τρόπο αυτό χρηματοδοτήθηκαν επενδύσεις ή όχι και το ζήτημα της εξυπηρέτησης του χρέους είναι το μόνο θέμα το οποίο αφορά τις χρηματοπιστωτικές αγορές δηλαδή αυτές που δανείζουν τα χρήματα στις χώρες ε, ε, όταν είναι να ανοίξουν στρόφιγγα, δεν θα θέσω το ερώτημα κατά πόσο έγιναν βιώσιμε επενδύσει ή όχι. Γι' αυτό θα ήθελα να σα προειδοποιήσω. Ε, δεν είναι το να ταξινομούμε τι ε, πράσινε δαπάνε ω θετικέ δαπάνε. Με τον τρόπο αυτό θα διολυστήσουμε στην επόμενη παγίδα υπερχρέωση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστούμε. Επόμενο ομιλητή, ο κύριο ε, Φερνάντε, ε, εκ μέρου των Σοσιαλιστών. Ε, Καλώ ήρθατε, κύριε Επίτροπε, στην Ευρωζώνη. Έχουμε 19 διαφορετικές χρηματοπιστωτικέ πολιτικές 19 κυβερνήσεις καταρτίζουν τους δικούς τους προϋπολογισμούς και προσπαθούν να εκπληρώσουν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αλλά εάν ε, μια κυβέρνηση προσπαθεί να εξηγιάνει το προϋπολογισμό και ε, το κατά πόσο υπάρχει μια συνοχή ε, αυτό συναρτάται με τις ε, κυκλικές ε, ανάγκες. Γι' αυτό πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση του συμφώνου. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να βελτιστοποιηθεί η ευελιξία τους ώστε οι να μπορέσουν να προβούν σε αντικυκλικές πολιτικές, αλλά το ζητούμενο εδώ είναι να πρικοδοτηθεί η Ευρωζώνη με μια γη θέση. Και το θέμα αυτό είναι που θα μας απασχολεί στους προσεχείς μήνες. Το εκ μέρους του Renew, κυρία Η αναθεώρηση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, έχει μεγάλη σημασία. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε μια σταθερή οικονομία. Και αυτό βεβαίως είναι καλό για όλες τις ευρωπαϊκές ε, χώρες και για τις χώρες οι οποίες ίσως ε, δεν το αντιλαμβάνονται. Μια Ολλανδική παροιμία λέει ότι ε, το καλύτερο είναι να δίνεις το καλό παράδειγμα. Αλλά περισσότερες ε, χώρες δεν χρησιμοποίησαν ε, τους ε, καιρούς των παχιών αγελάδων για να βάλουν τα οικονομικά τους τάξη. Οπότε τώρα θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα στην αποτελεσματικότητα των κανόνων και την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει μεγάλη σημασία οι κανόνες να είναι διάφανοι. Δεύτερον, οι κανόνες θα πρέπει να είναι απλούστεροι λιγότερο περίπλοκη. Θα πρέπει να ακολουθηθεί επίσης αντικυκλική πολιτική του προπολογισμού. Τρίτον, οι κανόνες δεν πρέπει να ερμηνεύονται με πιο ευέλικτο τρόπο. Η συμφωνία είναι συμφωνία και βλέπουμε με πολύ κακό μάτι την ε, πρόθεση της ε, Κομισιόν να θέσει τις ε, επανεπενδύσεις εκτός ε, του πεδίου εφαρμογή συμφώνου. Νομίζω ότι πρόκειται περί δημιουργικής λογιστικής. Και τέλος, δεν χρειάζεται μια ευρωπαϊκή λειτουργία σταθεροποίησης. Θα πρέπει τα σοκ να τα αντιμετωπίζουν μόνα τους τα κράτη-μέλη και σε αυτό θα βοηθήσουν και ή ε, αγορές. Αυτά λοιπόν θα ήθελα να πω, να είμαστε λοιπόν ειλικρινείς ε, όσον αφορά και την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κεφαλαίων. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σίλβια Σαρντόνε τώρα έχει τον λόγο. Συγχαρητήρια, Επίτροπε Τζοντιγλόνη. Δεν είναι εύκολο να μιλάτε για 10 λεπτά χωρίς να λέτε τίποτα. Όχι και ότι με εκπλήσει βεβαίω, ε, δεδομένη τη κυβέρνηση στην οποία ανήκατε, αλλά δεν φανταζόμουν ε, ότι εσεί ε, ως ω ε, γραφειοκράτη θα έρθετε εδώ πέρα να μα πείτε τίποτα. Έχουμε εδώ πέρα ε, συνενοχή του Τσίνκου Εστέλε με τους χριστιανοδημοκράτες. Παρ' όλα αυτά, η Ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει ε, ξεπουλώντας την κυριαρχία της. Μόνο και μόνο για να σώσει την πολυθρόνα του και το θόκο του ο Πρωθυπουργό. Όταν ε, υπάρχει μια χώρα όπως η Ιταλία με τέτοιο χρέος, δεν έχει κανένα ε, νόημα να λέμε πούμε, ότι θα δώσουμε αίμα. Ε, είναι σαν να λέει κάποιο ο οποίο του έχουν πάρει όλο το αίμα θα, δίνει, ας πούμε, θα, θα γίνει δωρητή αίματος. Μέσα σε τρία χρόνια ε, έχουμε ε, αυξήσει το εμπορικό ισοζύγιο πλωμών κατά 6%. Νομίζω ότι η Ευρώπη λειτουργεί ως Ευρώπη μόνο όταν τη βολεύει. Η Ιταλία έπεσε θύμα ε, επί χρόνια εκβιασμών. Εμείς θα πολεμήσουμε, θα πολεμήσουμε αυτή την επίθεση στην δημοκρατία. Θέλουμε να σώσουμε τους Ιταλούς. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να στηρίξουμε μια τέτοια πολιτική. Σα ευχαριστώ για τους ε, πράσινου. Ο κύριος ε, Ούρτασον έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Οι κανόνες τα τελευταία χρόνια ε, υπήρξαν αναποτελεσματικοί, δογματικοί και τελικά επιδίνωσαν τα πράγματα στην Ευρωζώνη. Και εγώ συμμερίζομαι τους προβληματισμούς που έκανα κάποιοι συνάδελφοι. Επίσης, τα όσα είπατε εσείς, ε, με βρίσκουν σύμφωνο, αλλά θα προσέθετα ότι υπάρχει το λεγόμενο output gap, το οποίο είναι ένα πρόβλημα για την εξυγίανση των εθνικών προπολογισμών. Ωστόσο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη συζήτηση και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα, το... θα προβεί σε αυτή τη συζήτηση. Και θα ήθελα να συζητήσω δύο πράγματα, κύριε Επίτροπε. Πρώτον, δεν, έχουμε... δεν φοβόμαστε να ανοίξουμε τεράστιε συζητήσεις όπως είναι αυτή. Θα πρέπει το Συμβούλιο να σταθεί μπροστά στον καθρέφτη του. Δεύτερον, θα πρέπει να προβείτε σε μια ευφυή εφαρμογή των κανόνων. Ε, εάν θέλουμε να έχουμε Green Deal. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει Green Deal χωρίς την εφαρμογή αυτών των κανόνων και επιμένουμε σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ουρτασούν. Ε, ο επόμενο ομιλητή εκ μέρου του ECR, ο κύριο Γιούρτσικα. Ευχαριστώ πολύ. Τα τελευταία χρόνια γίναμε μάρτυρες μιας ελαφράς βελτίωσης σε δημοσιονομικά ε, θέματα. Όσον αφορά την ε, ευρωπαϊκή κρίση χρέους, είδαμε ότι μειώθηκε τελικά το χρέος. Ορισμένοι οι πολιτικοί ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους ε, χρηματοοικονομικούς κανόνες. Δηλαδή, ίσως θέλουν υψηλότερο έλλειμμα, υψηλότερο χρέος. Ε, προκειμένου να πανεκλεγούν βεβαίως αντί να ε, θεωρήσουν, να προτάξουν το όφελος των πολιτών. Άρα δεν χρειάζονται πλέον εξαιρέσεις από τους κανόνες, αλλά αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι ένα πιο αυστηρό πλαίσιο για την εφαρμογή των κανόνων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει η κυρία Ομπρί για την Εγκούε για δύο λεπτά. Εδώ και τρεις μήνες οι Γάλλοι κατεβαίνουν στους δρόμους με χορεύουν, τραγούδουν εναντίον των μεταρρυθμίσεων των συντάξεων. Επί τρεις μήνες ε, πολεμούν για μια μεταρρυθμίση που θα τους κάνει να δουλεύουν πολύ περισσότερο πολλά, πολύ περισσότερα χρόνια και θα παίρνουν συντάξει πείνα. Ε, αυτή η μεταρρύθμιση εμπνέεται από, την, από το πλαίσιο το ευρωπαϊκό. Και λέει ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος συντάξεων θα μπορούσε να μειώσει το δημόσιο χρέος. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε οικονομίες από τις συντάξεις. Ακριβώς αυτό είναι η φιλοδοξία του, του συστήματος μεταρρύθμισης των συντάξεων. Θα πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε ότι οι συντάξεις ε, κοστίζουν πολύ ακριβά, η δημόσια υγεία ε, κοστίζει πολύ ακριβά. Ε, έχουν, έχουμε δημόσια νοσοκομεία τα οποία κλείνουν. Είναι πολλοί επαγγελματίες της υγείας είναι απογοητευμένοι. Έχουμε κοινωνική προστασία ελάχιστη όλο και περισσότερες οικονομίες. Έχουμε ε, μείωση των ε, φόρων για τους πλούσιους και τις ε, επιχειρήσεις. Αυτό ακριβώς κάνει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Όλη αυτή η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου βασίζεται σε ένα στόχο το ε, ιερό και παραβία στο όριο του 3%. Ένας ε, κανόνας που καθιερώθηκε μία μέρα γύρω από μια στρογγυλή, στρογγυλή τραπεζα και δεν έχει καμία οικονομική βάση και μάλιστα ε, επέκριναν αυτή την ε, αρχή η, τα μεγαλύτερα κεφάλια της οικονομίας. Ε, διερωτώμαστε για την λογική αυτών των κανόνων. Ήγκη και η ώρα, επιτέλους. Ε, θα πρέπει να μην ξεχνάμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ όλη η αρχιτεκτονική της ε, οικονομικής διακυβέρνησης της ε, Ευρώπης πρέπει να τι ξαναδούμε. Θα πρέπει για να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική αλλαγή και τις ανισότητες. Η αναθεώρηση του ε, εξαμήνου ίσως είναι μόνο γίνεται μόνο για ε, διακοσμητικούς λόγους. Γιατί δεν απαντά ούτε στις οικονομικές ούτε στις ιστορικές ανάγκες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάιερ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την ε, δουλειά που έκανε. Να πω ότι θεωρώ ή ότι οι αλλαγές αυτές είναι δικαιολογημένες ε, για να αντιμετωπίσουμε τις μη βιώσιμες πολιτικές πολλών κρατών μελών. Οι αλλαγές που έλαβαν χώρα ανάγκασαν χώρες να αναθεωρήσουν την πολιτική τους και έχουν φέρει την δημοσιονομική πολιτική πιο κοντά στην βιωσιμότητα, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο γιατί είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο. Θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προωθήσουν ε, τις ε, πολιτικές ε, που έχουν προτεραιότητα όπως το Green Deal, αλλά ταυτόχρονα είμαι σίγουρος ότι δεν είναι σωστή η αύξηση του χρέους. Μετά τις διαβουλεύσεις λοιπόν είμαι ανοιχτό σε αλλαγές ανάλογα με το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Νίντερμαϊρ. Τον λόγο έχει η κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πολλοί επικριτές ε, του συστήματος ε, αυτού το περιγράφουν ε, ως ε, έναν ε, φαύλο κύκλο του ευρώ, ο οποίος δεν αφήνει καθόλου περιθώρια στα κράτη-μέλη, γιατί είναι τόσο μεγάλη η λιτότητα, ώστε πνίγεται, καταπνίγεται η οικονομία. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ισορροπημένη πολιτική, προσανατολισμένη στην ευημερία. Θα πρέπει λοιπόν να βασιστούμε πρώτα απ' όλα στην κοινωνική πολιτική, στην ενίσχυση της ε, κοινωνικής και οικολογικής υποδομής. Η καταπολέμηση της ε, κλιματικής αλλαγής, αλλά και η ψηφιακή μετάβαση σημαίνει ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, περισσότερες δημόσιες επενδύσεις από το κράτος. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τον ορισμό του καθαρού ελίματος ε, και να ληφθεί υπόψη εδώ πέρα ο χρυσός κανόνας, δηλαδή δαπάνες χωρίς τις δημόσιες επενδύσεις όμως. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Γκίγκολτ. Κυρία Πρόεδρε, μια, ένα κοινό νόμισμα χρειάζεται και κοινού κανόνε για τον προπολογισμό. Αλλά Ας πούμε την αλήθεια εδώ πέρα, το σύμφωνο αυτό δεν έχει κάνει δεσμευτικό τον συντονισμό, ούτε έχει κάνει τους προϋπολογισμούς πιο ικανούς για το μέλλον. Δεν γίνεται πλέον, δεν γίνονται αντιληπτοί οι κανόνες ούτε από ειδικού όπως εγώ. Και αυτό σημαίνει ότι η Κομισιόν έχει μεγάλο περιθώριο για να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό σημαίνει ότι έχετε κάνει τους κανόνες ένα πολιτικό εργαλείο και ακόμη χειρότερα οι κανόνες αυτοί σημαίνουν ότι υπάρχει υποεπένδυση στα δημόσια αγαθά, εκπαίδευση, σιδηρόδρομοι, ίντερνετ, όλα υποφέρουν. Μεταξύ 2009 και 2018 το ποσοστό δημοσίων επενδύσεων έπεσε από 3,7 σε 2,9%. Χρειαζόμαστε όμως κανόνες που θα ευνοούν τις επενδύσεις. Και όλες τις επενδύσεις μάλιστα. Εξαίρεση για πράσινες ή ψηφιακές επενδύσεις μόνο όπως προτείνετε εσείς δεν λύνει το πρόβλημα γιατί έχουμε τα ίδια προβλήματα στην εκπαίδευση, στην κατοικία, στην υγεία. Γι' αυτό ε, δύο πράγματα λοιπόν είναι σημαντικά να ε, έχουμε έναν προπολισμό ικανό για τον μέλλον και απλοποίηση των κανόνων. Μόνο κατανοητοί κανόνες, είναι ισχυροί κανόνες που μπορούν να εφαρμοστούν. Ο κύριος Παπαδημούλης. Κύριε Τζεντιλόνι, ένας πρώην επίτροπος και πρώην πρωθυπουργός της χώρας σας, της Ιταλίας, ο κύριος Πρόντι, είχε αποκαλέσει το σύμφωνο σταθερότητας ηλίθιο ήσασταν κι εσείς πρωθυπουργό στην Ιταλία πριν γίνετε επίτροπος. Χρειάζεται αλλαγές σοβαρές και όχι απλώς συζήτηση για τις αλλαγές. Γιατί πρέπει να ενισχύσουμε τις επενδύσεις. γιατί μαζί με την απλούστευση που σημειώσατε χρειάζεται και ευελιξία. Πώς θα μειώσουμε τις τεράστιες κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες αν δεν συνδυάσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη με τα ασφαλή δημόσια οικονομικά. Είναι δυνατόν να εφαρμοστεί το Green Deal με αυτόν τον παράλογο θώρακα του Συμφώνου Σταθερότητας όπως εφαρμόστηκε 10 χρόνια. Και γιατί η Κομισιόν ήταν αυστηρή μόνο με τις χώρες που έχουν υπερβολικά ελλείμματα και δεν έκανε τίποτα για τις χώρες που έχουν υπερβολικά πλεονάσματα και παραβιάζουν τους κανόνες. Σε αυτά θέλουμε απαντήσεις. Ευχαριστούμε κύριε Παπαδημούλη. Και τώρα ο κύριος Κίρτσος. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με τον κύριο Τζεντιλόνι ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αυξήσουμε τις δημόσιες επενδύσεις. Ε, θεωρώ ότι είμαστε εφαρμόζουμε τους κανόνες. Ε, για παράδειγμα, συγκρίνεται τα δημόσια οικονομικά των ευρωπαϊκών χωρών είναι πολύ πιο αυστηρά από του ηνωμένου βασιλείου ή από των ηνωμένων πολιτειών γιατί υποθέτω ότι τέτοιου είδους συγκρίσεις πρέπει να κάνουμε σε έναν σύγχρονο και ανταγωνιστικό κόσμο. επίσης θεωρώ ότι έχουμε επιτύχει σε πάρα πολλά. σαν έλληνας μπορώ να σας πω ότι αν λέγαμε ότι το 2012 ή το 2015 η ελλάδα θα δανειζόταν το 2020 ε, με τόσο καλούς όρους και με το δεκαετές ομόλογο στο 11 εκατό ε, ε, δεν θα μας πίστευε κανείς. Επομένως δεν καταλαβαίνω ότι έχουμε χάσει τον έλεγχο, δεν έχουμε χάσει κανέναν έλεγχο, αλλά επειδή ακριβώς έχουμε τον έλεγχο και επειδή έχουμε επιτύχει με μεγάλο κοινωνικό κόστος βέβαια, πρέπει να οργανώσουμε μια επενδυτική εξόρμηση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ευχαριστούμε τον κύριο Κίρτσο. Η κυρία Μάρκες, για ένα λεπτό, η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δίνετε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για το Σύμφωνο ε, Σταθερότητας και Ανάπτυξης που έχει πολλές ε, δυναμίες. Το 2020 οι δημόσιες επενδύσεις είναι κάτω από το επίπεδο των επενδύσεων που περίπου στα μισά κράτη-μέλη ε, σε σχέση με τα προκρίσεις επίπεδα. Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Βιωσιμότητα των οικονομικών μας βέβαια. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις αντικυκλικές πολιτικές. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα σε ένα πιο απλό πλαίσιο και παράλληλα πιο ευέλικτο εκεί που χρειάζεται. Αλλά επαρκέ, βέβαια. Επίσης, θα πρέπει η ευελιξία των κανόνων του προπολογισμού να είναι κανόνας για να είναι πιο πράσινες οι επενδύσεις μας και να καταλάβουμε αν θα πρέπει να τροποποιήσουμε κάποια στοιχεία της στρατηγικής προϋπολογισμού ε, της Ευρωζώνης. Θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια με δείκτες και μεθοδολογίες που εξασφαλίζουν μεγαλύτερη δημοκρατία και μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο, Κύριε Καρέμ. Ε, κύριε Πρόεδρε, 0,5% για την ΑΣΤΑΚ. Ε, κάθε μέρα ακούμε διάφορους αριθμούς που μας, ε, θέλουν να μας παρουσιάσουν ως στοιχεία οικονομικής ευημερίας. θεωρούμε ότι είναι ο χρυσός κανόνας όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλά πότε επιτέλους θα διαφερθούμε για άλλους αριθμούς που είναι πολύ πιο σημαντικοί για το κοινό μας μέλλον το κόστος για παράδειγμα της κλιματικής αλλαγής ή της ε, κοινωνικής πολιτικής. Ε, το, τα, το, ο οίκος μας είναι σε φλόγες. Ε, ε, μια οικονομία υπεύθυνη είναι αυτή η οποία θα ενθάρρυνε τη μετάβαση σε, μια, σε, σε πράσινες επενδύσεις. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε το εξή, ε, συνάδελφοι. Θα πρέπει να εξέλθουμε από το δόγμα της ε, λιτότητας. Είναι προκειμένου να ανταποκριθούμε στην κλιματική αλλαγή. Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση αυτού του αιώνα. Προκειμένου να διαφυλάξουμε την διαβίωση στο κοινό μας ε, σπίτι. Όλα αυτά είναι στα χέρια μας και μόνο. Ε, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καρέμ. Επόμενη κυρία Τινάρη. Όχι, δεν βρίσκεται εδώ. Κυρία Τινάλη. Συγγνώμη, ήταν δικό μου το σφάλμα. Ε, επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Μάρκες. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, αυτή είναι μια σημαντική συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και της Ευρωζώνης ειδικότερα. Ε, καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε την οικονομική κατάσταση και τέσσερις του προπολογισμού στην Ευρώπη στο σύνολό της, αλλά θα έλεγα ότι η τρέχουσα οικονομική διακυβέρνηση είναι, έχει περιορισμένο και όχι πάντοτε θετικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό. Χρειαζόμαστε ένα περιθώριο για επενδύσεις, ιδιαίτερα πράσινες επενδύσεις. Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο το οποίο να ενδιαφέρεται περισσότερο για τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης, όχι μόνο για βραχυπρόθεσμους ε, οικονομικούς δείκτες. Χρειαζόμαστε περισσότερη ευελεξία σε, μια, τόσο δύσκολους καιρούς, ε, ιδιαίτερα αντικεκλικούς κανόνες. Θέλουμε μακροοικονομική ισορροπία για όλους, όχι για τους λίγους. Αλλιώς θα μπούμε σε μια παρατεταμένη, ε, ε, σε τέλμα στην Ευρώπη. Και αυτό θα συνεχιστεί εάν ορισμένε χώρες δεν θέλουν να διορθώσουν τα πλεονάσματά τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Kiitos erittäin paljon edustaja Marques. Sitten huomaan, että seuraavat puhujat eivät... Ευχαριστώ κύριε Μάρκες. Διάφοροι ομιλητές δεν είναι εδώ. μεταξύ των οποίων ο κύριος Γκουσμάου. Η κυρία Ντονάτο δεν ξέρω αν είναι εδώ μπορεί να μην μπόρεσαν να ταξιδέψουν και να φτάσουν λόγω της ε, καταιγίδα. Επομένως, θα περάσουμε στο Catch the Eye. Θέλω να ακούσω ποιος θα μιλήσει στο Catch the Eye. Η κυρία Σπυράκη είναι η πρώτη ομιλήτρια για το Catch the Eye. το σύμφωνο σταθερότητας αποτελεί το πλέγμα εκείνων των κανόνων που εγγυάται την ασφάλεια και την ευημερία του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. ταυτόχρονα όμως πρέπει τώρα να αποτελέσει το εργαλείο εκείνο για την εφαρμογή του green deal και χρειάζεται επιγόντως προσαρμογή. η προσαρμογή ακούει στο όνομα επενδύσεις πράσινες βιώσιμες αδρά χρηματοδοτούμενες επενδύσεις και από εθνικούς προϋπολογισμούς. και στη βάση αυτή θα ήθελα να σας θέσω ευθέως δύο ερωτήματα. το πρώτο ερώτημα σχεδιάζετε να δώσετε στην ελλάδα την ευκαιρία να διαθέσει επιπλέον δημοσιονομικό χώρο σε πράσινες επενδύσεις ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται σε μετάβαση από τον άνθρακα. πώς θα συμβεί αυτό όταν υπάρχει τόσο υψηλό υποχρεωτικό πρωτογενές πλεόνασμα; και το δεύτερο πιστεύετε ότι μπορούν να γίνουν επενδύσεις σε περιοχές σε μετάβαση με ειδικές φορολογικές ζώνες μειώνοντας δηλαδή ειδικά σε εκείνες τις περιοχές το φόρο προστιθέμενης αξίας προκειμένου οι επενδυτές να έχουν επιπλέον ένα ακόμη κίνητρο να κάνουν εκεί πράσινες επενδύσεις και να διατηρήσουν την κοινωνική συνοχή των περιοχών μας όπως είναι η δυτική μακεδονία και η μεγαλόπολη. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λέκας. Είναι εδώ. Ο κύριος Ολέκας δεν είναι εδώ. Ο κύριος Πέκερη. Ο κύριος Ολέκας έχει το λόγο. E, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλεκας λέγομαι. Γι' αυτό δεν αντιδρούσα όταν λέγατε εσείς Λέκας. Όλεκας λέγομαι. Σας ευχαριστώ. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι το σύμφωνο σταθερότητας για την δημοσιονομική μας ασφάλεια. Αυτό που με εξώθησε να ζητήσω το λόγο ήταν όταν σας άκουσα να λέτε ότι η μελλοντική μας ανάπτυξη μπορεί να αντιβαίνει στην Πράσινη Συμφωνία, να αντιβαίνει στο Green Deal. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λιγάκι για ποιο λόγο πιστεύετε ότι η Πράσινη Συμφωνία μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα ε, και να μην είναι ευκαιρία για την οικονομία μας. Γιατί το λέτε αυτό. Εγώ νομίζω ότι η Πράσινη Συμφωνία συμπεριλαμβάνει πολύ σημαντικές επενδύσεις στην ε, έρευνα, ανάπτυξη και επιστήμη, ούτως ώστε οι επιστήμονες να παραμένουν εδώ στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Όλεκας. Επόμενος. Ε, ο μιλητής ο κύριος Πέκκαρινεν. Για ένα λεπτό. Puhemies. ο εσύ τελούστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Teidän viestinne oli aika positiivinen. Σας ευχαριστώ. Το μήνυμά σας ε, ήταν θετικό θα έλεγα. Όμως ε, είπατε ότι το έλλειμμα στον προπολογισμό και ο λόγος του ελλείμματος είναι 80% εμείς αποφασίσαμε ότι πρέπει να είναι 60% σε κάθε χώρα στην ΟΝΕ. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα τελευταία χρόνια έχει ε, ρίξει στην αγορά εκατοντάδες ε, εκατομμύρια. Βλέπετε κάποια απειλή ε, στην αγορά έτσι ώστε η ίδια φούσκα που είδαμε στο παρελθόν να παραμονεύει πάλι ή απλά ήρεμα περιμένετε να επικρατήσει η σταθερότητα. Σας ευχαριστώ, Πέκαρινεν. Και ακολουθεί ο κύριος Ζωάο Φερέιρα. Η um οικονομική διακυβέρνηση δημιουργεί προσκόμματα στην οικονομική ανάπτυξη. Όπως έλεγε και η κυρία Μέρκελ, είναι τίποτα να μην κινείται σε πολιτικό επίπεδο ανεξάρτητα από την κυβέρνηση που υπάρχει. Δημιουργήθηκαν πάρα πολλές ανισορροπίες ε, στην κατανομή του πλούτου. Και εμείς εγκαταληφθήκαμε. Η οικονομική διακυβέρνηση μας εμπόδισε να κάνουμε το παραμικρό, να κουνηθούμε έστω και κατά μία κεραία. Δεν υπάρχουν επενδύσεις δεν υπάρχει παραγωγικό δυναμικό. Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν ξεχαρβαλωθεί. Δεν πρέπει να ξαναδούμε το σύμφωνο απλώς. Θα πρέπει να το καταργήσουμε αυτό το σύμφωνο σταθερότητας καθώς και το ευρωπαϊκό εξάμεινο που εξασφαλίζει το βάλτομα, ελάχιστους μισθούς και καμιά δημοκρατία. Ευτυχώς που ξύπνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά δεν θα πρέπει απλώς αυτά να είναι λόγια και ένα περιεχομένου. Ευχαριστώ. Κύριε Φερέιρα. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Καστάλντο. Δεν είναι εδώ όμως. Άρα, η κυρία Γιούτα Πάουλους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον με τι ζήλο συζητείτε εδώ ότι θέλουμε βιώσιμες, ε, ότι θα πρέπει βιώσιμες επενδύσεις να εξαιρεθούν από τους ε, κανόνες περί των επενδύσεων. Δεν θεωρώ ότι κάτι τέτοιο έχει νόημα, συμφωνώ μαζί σας, αλλά μου φαίνεται εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι κανόνες βιωσιμότητας σε άλλες επενδύσεις δεν παίζουν απολύτως κανένα ρόλο. Ε, γιατί ε, δισεκατομμύρια έχουν ε, χαθεί σε καύσιμα, σε επενδύσεις στον άνθρακα επενδύσεις χαμένες ε, που οδηγούν στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Και μου, φαίν, μου κάνει εντύπωση το γεγονό ότι από τη μία λέτε ότι δεν θα πρέπει να προσεγγίσουμε με τόση αυστερότητα τις βιώσιμες επενδύσεις. Από την άλλη θέλετε να δώσετε τόσα χρήματα σε μη βιώσιμες επενδύσεις. Ja sitten nyt on edustaja Castaldo, varapuhemies, saapunut paikalle ja hän πολύ. Ο Αντιπρόεδρος κ. Καστάλντο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, αγαπητέ Επίτροπε. Διαφορετικό ε, είναι το πλαίσιο από 10 χρόνια πριν. Ε, έχουμε χαμηλή παραγωγή. Φτάσαμε σε μια φάση που πρέπει να ξαναδούμε την προσέγγισή μας ε, αυτούς τους, αυτούς κανόνες και τους περιορισμούς του προπολογισμού που δεν είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της στιγμής. Ε, πρέπει να ελέγχουμε τους κανόνες, αλλά ε, υπάρχει και ένα πρόβλημα ασύμμετρης εφαρμογής και έτσι δημιουργείται μια ταχύτητα δύο ταχυτήτων λόγω ε, της υπερβολικής πίεσης της Κομισιόν απέναντι σε κράτη που έχουν δημόσιο χρέος. Έχουμε μακροοικονομικές ισορροπίε επίση σε κάποιες χώρες. Τελικά λοιπόν η Κομισιόν κατάλαβε βέβαια τη σημασία του τη σημασία που έχει το να ξαναδούμε του κανόνε του προπολογισμού, αλλά είναι σημαντικό να κάνουμε επενδύσει για να καταπολεμήσουμε τα ανεργία, ε, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης ε, αντιμετωπίζοντας κλιματική αλλαγή και να κάνουμε πράσινε επενδύσει και να έχουμε ίσω και πράσινα ομόλογα. Ε, Επίτροπε, ελπίζω να συνεχίσετε σε αυτόν τον δρόμο, γιατί ε, το να αλλάζουμε το ράβεξι, το να αρχίσουμε το ράβεξι είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η Ευρωζώνη. Ευχαριστώ κύριε Καστάλντο. Κύριε κυρία Γκραπίνη. Ε, ευχαριστώ Επίτροπε. Είμαι πεπισμένη ότι θα, με, θα μου απαντήσετε στο εξή ερώτημα. Αν η, προσαρμόσουμε την οικονομική διακυβέρνηση στην πραγματικότητα. Τι θα συνέβαινε με την Ευρώπη, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ε, δύο, μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, Σέγγεν και εκτός Σέγγεν. Έχουμε την Ευρωζώνη και χώρες εκτός της Ευρωζώνης. Έχουμε χώρες διαφορετικής οικονομικής ανάπτυξης. Έχουμε όμως το ίδιο. Όλοι όμως έχουμε τους ίδιους κανόνες ε, και τα ίδια όρια στο διαφορά το έλλειμμα. Και δεν μπορούμε να επενδύσουμε έτσι. Επίσης, τι θα γίνει με τα κονδύλια που χρειάζονται για την Πράσινη Συμφωνία. Αυτά θα μπορούσαν να δοθούν ε, στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Πώ θα εξασφαλίσουμε ότι οι πρώτε αλλαγέ ε, τη οικονομική διακυβέρνηση θα μειώσουν τι περιφερειακέ ανισότητε Τα κονδύλια ε, συγκεντρώνονται σε 4-5 χώρε με βάση το ελεγκτικό συνέδριο. Και αυτό αυξάνει την ε, περιφερειακή ανισότητα. Πώ θα ανταποκριθείτε σε αυτό, ε, προσπαθώντα να αλλάξετε του κανόνε οικονομική διακυβέρνηση. Ευχαριστώ την κυρία Γκραπίνη. Ο επόμενο ομιλητή, κυρία Ντέιλι. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πολλά μας είπε η Κομισιόν για την αναθεώρηση των δημοσιονομικών πολιτικών και των μέτρων που ελήφθησαν μετά το κράχ. Αλλά αυτά είναι λίγα πράγματα σε σχέση με το τι πραγματικά συμβαίνει στους Ευρωπαίους πολίτες. Εδώ πέρα απλά ξεπλένετε την λιτότητα. Είστε περήφανοι που μειώσατε τα υπερβολικά ελλείμματα όπως τα αποκαλείτε. Αλλά δεν μας λέτε τι σήμαινε αυτό για τους πολίτες τα χρέη των τραπεζιτών που πλήρωσαν οι πολίτες και το αποτέλεσμα το είδαμε αυτό στις Ιρλανδικές εκλογές όπου οι πολίτες καταψήφισαν την λιτότητα. Καταψήφισαν τους κανόνες ε, που σταματάνε τις επενδύσεις ε, στις εργατικές ε, κατοικίες και κάνουν τους ανθρώπους άστεγους. Η Κομισιόν λοιπόν μας ρωτάει τι μπορεί να γίνει καλύτερα σε αυτόν τον τομέα. Να σας πω εγώ να αλλάξουν οι κανόνες περί χρέους και ελλείμματος, να μην ισχύουν, παραδείγματος χάρη, για τις εργατικές κατοικίες. Δεν το κάνετε για τα όπλα, δεν μπορείτε να το κάνετε και γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Και τον λόγο έχει ο κύριος Γόλας και είναι ο τελευταίος στο Κετσιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το ξαναδούμε αυτό το σύμφωνο πρέπει να αποκτήσει μια καλύτερη μορφή, αλλά για να είμαι ειλικρινή, πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτε έχουν εγκαταληφθεί λόγω των αυστηρών κανόνων σας. Λέμε ότι ε, ε υπάρχει οικονομική σταθερότητα και ασφάλεια. Α, για ποιον! Δυστυχώς, πάρα πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπονται τα κράτη-μέλη χρειάζονται την ευελιξία για να φροντίσουν καλύτερα αυτούς που χρειάζονται βοήθεια. Και, όπως είπε και η συνάδελφος στην Ιρλανδία, το Σαββατοκύριακο, τα νεοφιλελεύθερα κόμματα που κυβερνούσαν υπέστησαν ήττα δεινή γιατί δεν εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα αυτών που έχουν ανάγκη. Και κάτι τελευταίο για τις υποδομές έχουμε αναγκαστεί να φτιάχνουμε υποδομές με ΣΔΙΤ ενώ μπορούμε να δανειστούμε λεφτά με 1% αν δεν είχαμε τον κανόνα του 3% που μας επιβάλλεται. Σας ευχαριστώ κύριε Γόλας. Οπότε χαίρομαι ιδιαίτερος που τηρήσατε όλο τον χρόνο ομιλίας. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον Επίτροπο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους βουλευτές για τις ε, παρεμβάσεις τους. Ε, νομίζω ότι αυτή είναι απλά η αρχή της ε, συζήτησης που θα έχουμε τους επόμενους 5-6 μήνες. Λοιπόν, αν υπάρχουν κάποιες κοινέ απόψεις σε αυτήν την συζήτηση, αντιλαμβάνομαι ότι ε, υπάρχει μια συμφωνία σε τρία γενικά πράγματα. Πρώτον, ότι πρέπει να αναθεωρηθούν οι κανόνες. Δεύτερον, είναι πολύ κύκλικη. Και τρίτον, πρέπει να γίνουν λιγότερο περίπλοκοι. Ε, είναι μια περιορισμένη βάση, αλλά ε, θα γεφυρώσουμε τις διαφορές μας πρέπει νομίζω να αποφύγουμε το σκεπτικό ότι έχουμε δύο διαφορετικές ιδεολογικές θέσεις ε, υπέρ της σταθερότητας, υπέρ κατά της ανάπτυξης ε, ε, γιατί έτσι δεν θα γίνει μια σωστή αναθεώρηση των κανόνων. Και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να συνεισφέρει σοβαρά στο να γεφυρώσουμε τις ιδεολογικές διαφορές. Μετά Υπάρχουν και άλλες διαφορές τις οποίες αντιλαμβάνομαι ότι δηλαδή εάν θέλουμε να απλοποιήσουμε να μην είναι ε, οι κανόνες αυτοί ε, κύκλικοι ε, νομίζω ότι μπορούμε να ε, πάμε προς σωστή κατεύθυνση. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Όλα αυτά συνδέονται με τον κύριο στόχο της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου δηλαδή την πράσινη μετάβαση. Η απάντησή μου είναι ναι. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθούμε πώς θα μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη μετάβαση χωρίς να υπάρχει μια σοβαρή δέσμευση για τις ε, δημόσιες δαπάνες. Γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του στόχου για την πράσινη μετάβαση και της αναθεώρησης της ε, οικονομικής ε, διακυβέρνησης. Ε, πρόκειται λοιπόν για ένα πρώτο βήμα στις συζητήσεις που θα συνεχιστούν τους επόμενους μήνες. Ευχαριστούμε κύριε Τζεντιλόνη. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Θα αλλάξει και επίτροπος. κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Συνάδελφοι, το επόμενο θέμα είναι δήλωση της Κομισιόν Αξιολόγηση της νέας μεθόδου διεύρυνσης που προτείνει η Κομισιόν. Λόγο έχει ο Επίτροπος ε, Βαρχέλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που βάλετε αυτό το θέμα στη ημερήσια διάταξη αμέσως μετά την υιοθέτηση από την Κομισιόν ε, της πρότασής της για την ε, αναθεωρημένη μεθοδολογία διεύρυνση. Με αυτόν τον τρόπο θα παρουσιάσουμε τι ιδέες μα και θα ενισχύσουμε τη διαδικασία ένταξης, ε, ούτω ώστε να είναι πιο αξιόπιστη η διαδικασία της ένταξης ε, της Ευρωπαϊκή Ένωσης ε, των Δυτικών Βαλκανίων. Εμείς γεωπολιτικά έχουμε επαφή με τους γειτονές μας, είναι πρώτη προτεραιότητα. Θα πρέπει να έχουμε ισχυρή και ενιαία φωνή και να παίξουμε πλήρως το γεωπολιτικό μας ρόλο ειδικά όταν πρόκειται για γειτονέ μα, απέναντι στου γειτονέ μα. Αυτό ισχύει 100%. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία. Προς το συμφέρον μας είναι αυτό, αλλά είναι και θέμα βέβαια αξιοπιστίας μας. Η προτεραιότητα της ε, Επιτροπής αυτής είναι να επιταχύνει την πρόοδο στα Δυτικά Βαλκάνια, να υπάρχει μια αξιόπιστη προοπτική μελλοντική ένταξης, Γι' αυτό ε, δουλεύουμε πάνω σε τρεις άξονες. Ο πρώτο είναι η ανακοίνωση για την αναθεωρημένη μεθοδολογία διεύρυνση, που θα σα εξηγήσω όσον ούπο πιο αναλυτικά. Δεύτερος άξονας είναι να ανοίξουμε ε, διαπραγματεύσεις με την ε, Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και θα παρουσιάσουμε ένα οικονομικό σχέδιο ανάπτυξης για την περιοχή. Θα ενισχύσουμε την προσπάθεια οικοδόμησης ε, στεναρών και ανθεκτικών οικονομιών και θα προσπαθήσουμε να φέρουμε αυτές τις χώρες πιο κοντά στα δικά μας πρότυπα. Σε ό,τι αφορά την αναθεωρημένη μεθοδολογία διεύρυνσης, έχουμε τέσσερις βασικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν και για τις χώρες ε, που είναι υπό ένταξη, αλλά και για τα δικά μα κράτη-μέλη. Καταρχά, θα πρέπει να είναι πιο αξιόπιστη η διαδικασία. Οι χώρε θα πρέπει να κάνουν τι μεταρρυθμίσει που υπόσχονται και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιδράει σε αυτή την πρόοδο για να υπάρχει αξιοπιστία θα πρέπει να εστιάσουμε στις ε, θεμελιώδες, ε, θεμελιώδες ελευθερίες και μεταρρυθμίσεις γιατί αυτή είναι η καρδιά της πραγματικής αλλαγής και μετασχηματισμού. Αυτό σημαίνει κράτος δικαίου, ε, λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, οικονομικά κριτήρια και αξιόπιστη δημόσια διοίκηση. Επίσης, η πολιτική διαδικασία θα πρέπει να μπει στο προσκήνιο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε συμμετοχή υψηλού επίπεδου στι χώρε αυτέ μέσω ε, τακτικών συνόδων κορυφή ε, με τα Δυτικά Βαλκάνια και υπουργικών συνόδων. Θα πρέπει να εμπλέξουμε τα κράτη-μέλη ε, πιο έντονα και να του δώσουμε περισσότερε ευκαιρίε να παρακολουθήσουν και να θεωρήσουν τη διαδικασία για να στηρίξουν ε, τι θεμελιώδει ελευθερίε. Όμω χρειάζονται αυτέ τι θεμελιώδει ελευθερίε. Η τρίτη ελευθερία είναι η ανάγκη η διαδικασία αυτή να γίνει πιο δυναμική με έμφαση σε βασικούς τομείς. Ομαδοποίηση κεφαλαίων τομείς πολιτικής, ούτω ώστε να κάνουμε πιο ενδελεχή πολιτική συζήτηση ανά θέμα. Επίσης θα μας επιτρέψει να εντοπίσουμε ευκαιρίες για γρήγορη ευθυγράμμιση και εμπλοκή των, ε, στις ε, ε, δικές μας πολιτικές, όπως ψηφιακή ατζέντα, τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και ενέργειας. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι όταν γίνονται και εφαρμόζονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις, πριν από την έναρξη, τότε ε, η έναρξη το, της ομάδας κεφαλαίου και το κλείσιμο των επιμέρους κεφαλαίων θα πρέπει να περιοριστεί εντός του χρόνου. Ε, αυτό εξαρτάται βεβαίως από την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων της χώρας. Αυτό είναι σημαντικό, σημαντική πολιτική προσφορά από πλευράς μας προς την περιοχή. Αν κάνουν αυτό που πρέπει, θα είμαστε κι εμεί έτοιμοι να του δώσουμε αυτό που πρέπει. Ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα, ε, οι μεταρρυθμίσει τη δημόσια διοίκηση, τα οικονομικά είναι βασικό στοιχείο. Θα είναι το πρώτο κεφάλαιο που θα ανοίξει και θα είναι το τελευταίο που θα κλείσει. Και επαρκής πρόοδος χρειάζεται σε αυτούς τους τομείς, ούτω ώστε να ανοίξουν άλλες ομάδες κεφαλαίων. Επίσης, θα πρέπει η διαδικασία να είναι πιο προβλέψιμη και για τις δύο πλευρές. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιε χώρε θα πρέπει να έχουν σαφήνεια μεγαλύτερη για τις συνθήκες που θα πρέπει να εκπληρούν και ποιε είναι οι θετικέ επιπτώσεις όταν υπάρχει πραγματικά πρόοδο και ποιε είναι οι αρνητικέ συνέπειες σε περίπτωση που δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Χρειαζόμαστε ε, σαφή, κίνητρα για να υπάρξουν μεταρρυθμίσει. αν οι χώρε προχωρήσουν. Ε, Στι μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνήσει, τότε οι πολίτε θα πρέπει να δουν τα ωφέλη αυτής της ε, ένταξης, της ε, επιταχυμένης ε, αυτής προσπάθειας και θα υπάρχει μεγαλύτερη χρηματοδότηση και επενδύσεις. Παράλληλα, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι σίγουρα ότι υπάρχει δυνατότητα αντιστροφής και διορθωτικών μέτρων όταν οι μεταρρυθμίσεις αυτές ε, εκτροχιάζονται. Αυτό θα γίνεται μέσω πιο αποτελεσματικών μέτρων, ε, επιβολής κυρώσεων, ε, σε περίπτωση που υπάρχει βάλτομα ή οπισθοχώρηση. Επίσης, θα πρέπει να επαναλάβω ότι ενισχύουμε και βελτιώνουμε τη διαδικασία βεβαίως, αλλά ο στόχος είναι παραμένει ο ίδιος, η προσχώρηση και η πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα με αυτό, δεύτερο στοιχείο, δεύτερος άξονας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει συστάσεις για να ανοίξουν ε, οι διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και τη Βόρειο Μακεδονία και ελπίζουμε να μπορέσουν να ξεκινήσουν πριν από την Σύνοδο ε, στο Ζάγκρεπ. Γιατί και οι δύο χώρε έκαναν αυτό που του ζητήσαμε. Στην πρόσφατη, στην πρόσφατη επίσκεψή μου στα Σκόπια και στα Τύρανα, τόνισα τη σημασία των ε, μεταρρυθμίσεων και ζήτησα να συνεχίσει η εφαρμογή του. Και οι δύο χώρε έχουν προχωρήσει και θέλουν να κάνουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Παράλληλα, για να είμαστε αξιόπιστος εταίρος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, κάνει αυτό που υποσχέθηκε. Η Κομισιόν θα δώσει λεπτομέρειε πληροφορίε για την πρόοδο που έκαναν αυτέ οι δύο χώρες ε, το Φεβρουάριο για να προετοιμάσουμε το έδαφο για το Συμβούλιο που θα πάρει την απόφαση. Και είμαστε πεπισμένοι ότι οποιαδήποτε περαιτέρω αναβολή θα οδηγήσει σε κίνδυνο να υποσκάψουμε τη σταθερότητα ολόκληρη περιοχής. Κινδυνεύουμε επίσης ε, χειρισμούς από τρίτες χώρες και άλλα αλότρια αφηγήματα. Επίσης, αυτές οι μετασχηματιστές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνουν οι χώρες των Δυτικών ε, Βαλκανίων θα πρέπει να υποστηριχθούν όταν έχουμε ε, οικονομίες της αγοράς, ε, οικονομίες που λειτουργούν. Ε, Επομένω, εν ώψη τη ε, Συνόδου Κορυφή ε, του Ζάγκρεπ, θα προτείνουμε μια νέα προσέγγιση πολιτική που θα είναι ο κροκονιαίο λίθο για την ατζέντα που θα πρέπει να ακολουθήσει η περιοχή. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την παρουσία μα στα Δυτικά Βαλκάνια, θα πρέπει να αυξήσουμε τι επενδύσει και να βοηθήσουμε για να κλείσουν τα χάσματα τη οικονομική ανάπτυξη μεταξύ ημών και ημών. Θα πρέπει να δούμε τι μέτρα πρέπει να λάβουμε, ούτω ώστε να υπάρξουν επενδύσει στα Δυτικά Βαλκάνια, να ενισχύσουμε την πρόσβαση στην νέα αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση και επιχειρηματικέ ευκαιρίε, να βελτιώσουμε τι επιχειρήσει και το επενδυτικό κλίμα και να σταματήσουμε τη φυγή των εγκεφάλων από την οποία πάσχει η περιοχή. Όπω βλέπετε, είναι μια πολύ φιλόδοξη ατζέντα αυτή για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Χρειαζόμαστε πολιτική στήριξη από το Κοινοβούλιο για να τα καταφέρουμε. Μαζί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αξιοπιστία και εμπιστοσύνη, άρα θα πρέπει να μεταχειριζόμαστε του εταίρου των Δυτικών Βαλκανίων όλο και περισσότερο σε μελλοντικά μέλη. Αυτός είναι ο κοινά αποδεκτός προορισμός μας. Είναι προ όφελο τη Ευρωπαϊκή Ένωση εν το σύνολο Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you, Commissioner. I now open the floor for Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Τώρα το λόγο έχουν οι ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Η κυρία Γκάλ εκ μέρους του ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ε, ε, θα ήθελα να πω ότι χαιρετίζω αυτή τη νέα διαδικασία που προτείνει η Επιτροπή, γιατί μπορούμε με τον τρόπο αυτό να βγούμε από το αδιέξοδο και μπορεί να αποτελέσει μια γέφυρα μεταξύ δύο ομάδων ε, χωρών μελών. Η μεν είναι υπέρ τη διεύρυνσης, οι άλλε πιο επιφυλακτικέ. Ε, θα πρέπει να είμαστε προσανατολισμένοι στο αποτέλεσμα και για το Μαυροβούνιο θα πρέπει να είναι θετική αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει να προχωρήσουμε τις χώρες αυτές ο κύριος Επίτροπος σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα υπέβαλε μια θετική πρόταση και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε ίσως να λύσουμε την κατάσταση αυτή πριν από τη Σύνοδο Κορυφή το Μάρτιο και μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ευρωματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία γιατί και οι δύο χώρες κατέληξαν σε αποτελέσματα και τώρα θα πρέπει οι χώρες μέλη καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουν ένα βήμα προς τα μπρος. Το διακύβευμα εδώ είναι οι χώρες αυτές των Δυτικών Βαλκανίων κατά πόσο θα υπάρξει ειρήνευση και σταθεροποίηση στην περιοχή αυτή. Ο κύριος Πίτσουλα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Επίτροπο για τις προσπάθειες που κατέβαλε και το κείμενο που υπέβαλε η νέα προταθήσα μεθοδολογία ε, έρχεται μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων. Είναι αυτονόητο ότι τα πρωτεία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας. Θέματα που σχετίζονται με τη διαφθορά, τη δικαστική εξουσία και το οργανωμένο έγκλημα, καθώς και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ελευθερία της έκφρασης. Ε, συμφωνώ ότι θα πρέπει να υπάρξουν πιο θετικά στοιχεία προκειμένου οι χώρες αυτές να ολοκληρώσουν το πρόγραμμά τους όσον αφορά το δίκτυο μεταφορών ή το Ευρωπαϊκό Green Deal. Ε, η δική σας προσέγγιση δεν ε, διαφοροποιείται πολύ από το υφιστάμενο πλαίσιο διαπραγμάτευσης που έγινε πιο πολύπλοκο μετά τη τελευταία διεύρυνση. Ε, το θέμα είναι κατά πόσο οι χώρες αυτές προτίθενται να κάνουν τις διαπραγματεύσεις βάσει της νέες μεθοδολογίες. Για παράδειγμα, το Μαυροβούνι διαπραγματεύεται εδώ και 8 χρόνια και μόνο ένα κεφάλαιο παραμένει ανοιχτό. Ε, γι' αυτό ελπίζω ότι ε, τα πιο επιφυλακτικά μέρη θα συμφωνήσουν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Γιατί μια απόφαση μετάθεσης αυτής της διαδικασίας θα καθυστερήσει πάρα πολύ το μέλλον των χωρών αυτών. Η νέα μεθοδολογία μας δίνει ένα βιώσιμο μοντέλο και να εναπόκειται τώρα στις χώρες μέλη να μπορέσουν να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους όσον αφορά την διαδικασία της διεύρυνσης. Ο κύριος Κουτσούκ, εκ του Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσω από το τέλος. Κύριε Επίτροπε, μιλάμε για την αποτυχία του Συμβουλίου του Οκτωβρίου. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλη αποτυχία τον Μάρτιο. Και συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε ότι πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα και να μην κάνουμε υποσχέσεις ε, που δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε. Σήμερα όμως πρέπει να δούμε πώς ε, μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί και να δούμε τι θα κάνουμε για τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες των λαών των Δυτικών Βαλκανίων. Ελπίζω να μην έχουμε πάλι εκπλήξεις στην τελευταία στιγμή. Είναι πάρα πολύ νωρί για να βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς θα λειτουργήσει η νέα μεθοδολογία, αλλά για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου πρέπει να έχει δυναμισμό αντί να περιπλέξει τα πράγματα. Να εστιάσει περισσότερο στις ε, θεματικές δέσμες και να έχει σαφείς όρους Είμαι υπέρ της νέας αυτής διαδικασίας. Αλλά δεν θέλω η νέα αυτή ιδέα να καταλήξει ξανά σε μια κατάσταση όπου η περιοχή θα μείνει πάλι εκτός ε, νυμφώνος. Ε, γι' αυτό στην πολιτική μας ομάδα προσφάτως εγκρίναμε ένα έγγραφο θέσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια με βάση τις αξίες μας. Ε. Θέλουμε οι πολίτες ε, των υποψήφιων χωρών να έρθουν πιο κοντά και να ωφεληθούν από την διαδικασία ένταξης. Να έρθουμε σε επαφή με τους εταίρους μας ε, νωρίτερα στις ε, βασικές πολιτικές όπως το πράσινο deal, ψηφιακές πολιτικές κτλ. για να μπορέσουν να ωφεληθούν πριν από την ένταξη. Η ευρωπαϊκή προοπτική είναι ισχυρό κίνητρο για μεταρρυθμίσεις και εμείς στην ομάδα μας πάντα ήμασταν υπέρ μιας σαφούς τέτοιας πολιτικής. Θεωρούμε ότι οι μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι με τη διαδικασία διεύρυνση. Πρέπει να μεταρρυθμίσουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι λόγω των χωρών αυτών, αλλά για δικούς μας λόγους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δίνω τώρα τον λόγο στην κυρία Μπομφρίσκο για δύο λεπτά. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η προσφορά αυτή που κάνετε βεβαίως αποτελεί και μια παραδοχή αποτυχίας στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα τον μηχανισμό του κράτσου που είναι η μοναδική διασφάλιση. Όμως Έχουμε ανεργία και οικονομική ανισορροπία η οποία εκθέτει την περιοχή σε ασύμετρα σοκ. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια εγγύηση της συνύπαρξης σε ένα διευρυμένο σύστημα μεταξύ ε, αρκεί αυτό ε, για την ιδιαιτερότητα της Αλβανίας η οποία βρίσκεται σε ένα πόλεμο με τον εαυτό της. Ε, υπάρχει διαφθορά, ε, δεν υπάρχει δημοκρατική κουλτούρα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη οργανωμένη εγκληματικότητα. Ε, λοιπόν, συνάδελφοι και κύριοι Επίτροπε, η Κομισιόν προτείνει μία μέθοδο, αλλά δεν μπαίνει στην ουσία των ε, θεμάτων. Λοιπόν, ακριβώς αυτά τα είδαμε πριν από λίγους μήνες για αυτές τις χώρες αλλά θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι μελλοντικέ προοπτικέ ε, ένταξη αυτών των χωρών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τα ζητήματα και τις ε, ασφάλειες τα οποία έχουν ε, χειροτερέψει. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτείτε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες σας έχουν δώσει μια σαφή εντολή να υπερασπιστείτε και να προστατεύσετε την Ευρώπη. Λοιπόν, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις πάρα πολλές αβεβαιότητες ε, των Δυτικών Βαλκανίων. Θα πρέπει λοιπόν να αποτελέσει βασικό κομμάτι της διαδικασίας αυτής το μη αναστρέψιμο του κράτους κέου. Σας ευχαριστώ για τους ε, πράσινους για ένα μισή λεπτό. Η κυρία Φων Κράμον Ταουμπαντέλ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάλφοι, καλωσορίζουμε τη νέα μεθοδολογία για την διεύρυνση. Οι δέσμες αυτές μας δίνουν μια νέα δυναμική, αλλά βεβαίως ε, ιδιαιτέρως ε, μεγάλη σημασία έχουν τα θεμελιώδη, το κράτος δικαίου και η χρηστή διοίκηση. Χωρίς αυτά δεν γίνεται τίποτα. Δυστυχώς οι δημοκρατικοί θεσμοί δεν είναι ασφαλείς. Το κράτος δικαίου και ο πλουραλισμός των ε, ΜΜΕ έχουν αρχίσει να υποχωρούν στην Σερβία από το 2014 και όμως παριστάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα και συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις. Χωρίς τα βασικά όμως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Με τη νέα προσέγγιση μπορούμε να προχωρήσουμε όταν δούμε πρόοδο. Οι πιο φιλόδοξες χώρες πρέπει να περιλαμβάνονται σε όσο δυνατόν περισσότερες ευρωπαϊκές πολιτικές. Έτσι θα ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας και θα αλλάξουμε τις ζωές των πολιτών στην περιοχή. Η νοτιοανατολική Ευρώπη πρέπει επίσης να ενταχθεί στο πράσινο deal για να είναι η Ευρώπη κλιματικά οδέτερη μέχρι το 2050. Όμως πρέπει να τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Γιατί η απογοήτευση ε, από το Συμβούλιο του Οκτωβρίου δεν πρέπει να επαναληφθεί χρειάζεται να δοθεί επιγόντως το πράσινο φως στις δύο χώρες και να αναθεωρηθεί το καθεστώς βίζας καθώς πληρούν τα κριτήρια. Η νέα μεθοδολογία έχει νόημα αν την τηρούμε κι εμείς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για το ECR για ένα λεπτό η κυρία Στέγκρουντ. Fru talman! ευχαριστώ. Η Βρετανική σημαία κατέβηκε από το κτίριο και υλοποιήθηκε πλέον η μεγαλύτερη αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Βρετανοί έφυγαν εν μέρη Ε, λόγω των ε, εξελίξεων αυτών. Η Σουηδία, όπως και άλλες χώρες, έχει πρόβλημα με το μισθολογικό ντάμπινγκ, ε, την εγκληματικότητα, έλλειψη στέγης, έχουμε χαμηλή οικονομική ανάπτυξη και πρέπει να εδαχτούμε από το παρελθόν, αλλά δεν εστιάζουμε σε αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τους ε, Σουηδούς ε, συναδέλφους πώς γίνεται να διαπραγματευόμαστε με τις ε, χώρες αυτές όταν έχουμε εμείς τόσο κακή οικονομία και ενεργεία. Γιατί αυτά τα πληρώσει ο Σουηδός φορολογούμενος. Ευχαριστώ, Μπίλτσικ. Thank you very much, Madam President. And... Ευχαριστούμε πολύ, κυρία... Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε επίσης την Επιτροπή ως εισηγητής για την ε, Σερβία ε, και για το αντιπρόεδρος για το Μούνιο, χαιρετίζω την ε, πρωτοβουλία σας. Είναι το πρώτο βήμα βεβαίως ένα ταξίδι, ένα ταξίδι προς τη διεύρυνση ως πετυχημένη ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Οι εταίροι μας θα πρέπει να κερδίσουν εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή προοπτική και η επικοινωνία είναι το στοιχείο κλειδί εδώ. Χαίρομαι λοιπόν την περασμένη εβδομάδα σε μια κοινή επίσκεψη. Ε, το αποδείξαμε αυτό στην επίσκεψή μας στο Βελιγράδι όταν επισκεφθήκαμε τους ε, εταίρους μας. Τώρα έχει έρθει η ώρα να συμμετάσχει και το συμβόλιο το πρώτο βήμα είναι να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει το Μάρτιο με την ε, Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, γιατί μόνο τότε ε, μπορούμε να δεσμευτούμε ως προς τα ουσιώδη. Ε, το να, η διεύρυνση δεν μπορεί παρά να σημαίνει επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ε, η κυρία Σάντος για δύο λεπτά, δυόμιση, ενάμιση λεπτό. Η πολιτική διεύρυνση είναι μία από τι πιο σημαντικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η βάση για το κράτο δικαίου, για την ειρήνη και την ευημερία. Η πρόταση αναθεώρηση τη μεθοδολογία διεύρυνση είναι μία νέα φάση στην οποία μπαίνουμε και τώρα θα ενισχύσουμε τη διαδικασία ένταξης. Θα υπάρχει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα με βάση σαφείς στόχους που εξασφαλίζουν μια διαδικασία λήψη αποφάσεων που βασίζεται στην αξία του καθενός, ούτως ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Περισσότερες μεταρρυθμίσεις των θεσμών, σεβασμός του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών ελευθεριών. Ε, όλα αυτά τα θέματα μπαίνουν στο φάκελο της διεύρυνσης της εκάστοτε χώρας. Και αυτά ήταν θέματα που πάντα τα θέλαν οι σοσιαλδημοκράτες. Γι' αυτό ακριβώς ε, είμαστε χαρούμενοι για τη σημασία που δίδεται στο κεφάλαιο αυτό, στο σύνολο της πρότασης. Όμως δεν μπορώ πάνω να σας πω ότι υπάρχει μια δηλία με την οποία αναφερθήκατε στην παρουσίασή σας σε αυτά τα θέματα. Αντίθετα με αυτό που συνέβη σε άλλες συνεδριάσεις όπου είχε υποθεί ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εμπλακούν περισσότερο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφή μηχανισμό για τη συμμετοχή των κρατών μελών στη διαδικασία διεύρυνση. Θα πρέπει να υπάρχει μια οικονομική, πολιτική και πολιτική σύγκληση για να υπάρχει ε, επιτυχή ε, διεύρυνση και αυτό δεν τονίζεται επαρκώ. Ως ε, εισηγήτρια για την έκθεση για την Αλβανία πρέπει να σα πω ότι δεν θέλουμε αυτή η μεταρρύθμιση να χρησιμοποιηθεί ούτω ώστε να καθυστερήσουμε ή να εμποδίσουμε τη διαδικασία διεύρυνσης, ε, ειδικά με την Βόρειο Μακεδονία και την Αλβανία. Ε, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Κομισιόν έχουν αναλάβει σαφέστατες δεσμεύσει απέναντι σε αυτές τις χώρες. Ε, συγγνώμη, αλλά σα έκοψα γιατί πρέπει να ε, τηρήσετε το χρόνο σα. Κυρία Λουαζό, ένα λεπτό. Ε, είναι και η ώρα επιτέλου. Η, η συζήτηση για τη διεύρυνση ε, ε, ήταν παλιά μία συζήτηση ρουτίνα. Το να γίνει τώρα μια τέτοια συζήτηση είναι πολιτική επιλογή και θα πρέπει να ενδιαφέρει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι υποψήφιε χώρε. Χαιρετίζω την πρόταση τη Κομισιόν, η οποία βάζει σαφήνεια, προοδευτικό χαρακτήρα και περισσότερε ευθύνε για όλου του παίκτε τη διαδικασία διεύρυνση. Ε, αν, αν υπάρξει πρόοδο, πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μα. Αν υπάρχει οπισθοχώρηση, επίση θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα και να υπάρξουν συνέπειε. Χαιρετίζω την έμφαση που δίνεται στο κράτο δικαίου σε όλη τη διαδικασία προ την ένταξη στην Ένωσή μα. Το κράτο δικαίου δεν είναι ένα κουτάκι που βάζουμε νη ή ένα σημείο όπου βάζουμε την υπογραφή μα. Είναι το σημείο σύγκλησή μα. Έχουμε πάρα πολλού ε, αντιπάλου τη Δημοκρατία και τη Ένωσή μα και δεν θέλουμε να βάλουμε κι άλλου μέσα στην Ένωση τιμητέ μα. Δεν θέλουμε απλώ δηλώσει ε, ε, προθέσεων ή μεταρρυθμίσει στα χαρτιά. Αυτό που έχει σημασία είναι η πραγματικότητα, η καθημερινότητα και η υπεράσπιση των θεμελιωδών μα αξιών. Για να τελειώσω, θέλω να σα ε, κρούσω το ογκόδωνα αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μεγαλώσει, θα πρέπει να μπορεί να μεταρρυθμιστεί. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κι άλλα μέλη σε ένα νίκο, ο οποίο είναι σε διάλυση, ξεχαρβαλωμένο. Πρέπει να περάσουμε στην πράξη. Η διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη θα μα δώσει την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να βάλουμε στάξη τον, τον νίκο μα. Α την αδράξουμε. Για ένα μισή λεπτό, ο κύριο Ριβιέρ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η Επιτροπή προτείνει μια νέα μεθοδολογία προκειμένου να προσεγγίσει τι νέε ε, προσχωρήσει εκ μέρου των χωρών των Δυτικών Βελκανίων. 35 κεφάλαια θα αντικατασταθούν από ένα σύστημα διαπραγμάτευσης. Ωστόσο αυτή δεν είναι η επιλογή των λαών. Η Επιτροπή ε, θα προτείνει να ξεκινήσουν εκ νέου διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία και θέλει να προωθήσει ένα, ε, ε πολλές ε, επενδύσεις στις χώρες αυτές. Ε, δεν, θα, δεν ξέρω αν θα προσεγγιστούν θέματα όπως είναι η τρομοκρατία, η απόσπαση των εργαζομένων, ε, πολλά ουσιώδη θέματα τα οποία πάνε σε δεύτερη μοίρα. Η συνέντευξη των κεφαλαίων δεν μπορεί παρά να ενισχύσει την εξουσία της Επιτροπής. Ε, με τα κλάστερ αυτά θα περιθωριοποιηθεί η διαδικασία της ε, διεύρυνσης και το Συμβούλιο θα έχει το πάνω χέρι. Οι λαοί επιθυμούν να ξεκινήσει αυτό το, να, σταματήσει αυτά, να σταματήσουν αυτά τα κύματα συνεχών διευρύνσεων. Ε, το απέδειξαν στο ψήφισμα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ενίσχυση του τεχνοκρατικού ευρωπαϊκού πνεύματος σε βάρους σε βάρος των λαών. Ο κοροναϊός εκθέτει τους λαούς της Ευρώπης την ασφάλεια στον τομέα της υγείας για παράδειγμα και όλα αυτά είναι συνέπειες αυτής της ε, πολιτικής ε, τρέλας. Η κυρία Στρέκη, ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είμαστε ευτυχεί που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε αυτή την πρόταση, γιατί αναμένουμε τώρα από τα κράτη-μέλη ότι η έγκριση της πρότασης αυτής θα οδηγήσει σε έναρξη διαπραγματεύσεων με την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Η Επιτροπή και η Προεδρία μπορούν να μας διαβεβαιώσουν ότι αυτή η μεθοδολογία όταν θα εγκριθεί το Συμβούλιο θα δώσει και το πράσινο φως το Μάιο. Ελπίζω λοιπόν όλη αυτή η πίεση να ασκηθεί πραγματικά σε επίπεδο κρατών μελών. Καλώς ορίζουμε την έμφαση στο κράτος δικαίου και το σκέλος της ευελιξίας που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο τα κράτη-μέλη στη διάρκεια της διαδικασίας. Έχουμε κάποιες ανησυχίες σε ό,τι αφορά την ε, διαδικασία, ωστόσο. Όταν ε, πρόκειται για το θέμα της ε, ομοφωνίας, η οποία πλέον δεν απαιτείται σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό λοιπόν είναι δύσκολο για την αναστροφή κάποιων καταστάσεων και για την έρεξη κάποιων καταστάσεων. Πώς μπορούμε λοιπόν να αποφύγουμε την πολιτική αυθαιρεσία στη λήψη αποφάσεων και μεγαλύτερη ασφάλεια για τις υποψηφίες χώρες. Και αυτό μπορεί να αμφισβητηθεί και από θεσμική άποψη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια διαφορετική διαδικασία σε ό,τι αφορά την διαδικασία αναστροφής παρά την διαδικασία κίνησης. Παρακαλώ λοιπόν αναλύστε το θέμα αυτό. Η κυρία Τόμας, έτσι ένα λεπτό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 οι προτάσεις αυτές ικανοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα αιτήματα της ε, Γαλλίας και ανοίγουν το δρόμο στην ένταξη και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Και αυτό είναι καλό γιατί αυτές οι χώρες δεν θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα των εσωτερικών μας διαφωνιών. Ε, οι προτάσεις Κομισιόν προβλέπουν και ε, κυρώσεις ή ε, διακοπή των διαπραγματεύσεων και αυτό είναι καλό όταν παρουσιάζονται προβλήματα. Η διαδικασία ένταξη είναι μακρά και δυσχερής. Θα πρέπει να καταλαβαίνουμε, να κατανοούμε τα προβλήματα των υποψήφων χωρών, αλλά θα πρέπει να είμαστε και συνεπείς, έτσι ώστε να πληρούνται τελικά τα κριτήρια και να εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες για όλους. Είναι ο μόνος τρόπο προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ε, πίστευτη ε, και ταυτόχρονα να κρατήσει ανοιχτή την πόρτα της και σε άλλες χώρες. Κυρία Ζόβκο, για ένα λεπτό. Επίτροπε, συγχαρητήρια. Παρουσιάσατε την προηγούμενη εβδομάδα τη νέα μεθοδολογία διεύρυνση, ελπίζοντα ότι θα στείλετε ένα θετικό μήνυμα στι υποψήφιε χώρε και ελπίζοντα ότι ταυτόχρονα θα ικανοποιήσετε και τι ανησυχίε των κρατών μελών. Οι αντιδράσει και από τα κράτη-μέλη και από τι ε, χώρε των Δυτικών Βαλκανίων είναι πολύ θετικέ. Ε, προσπαθείτε να αποφύγουμε την επανάληψη του μπλοκαρίσματος που εμφανίστηκε πριν από μερικούς μήνες. Η, η αξιοπιστία και η πολιτική ε, ε διεύθυνση, η πολιτική εξουσία είναι πολύ σημαντικά κομμάτια της ένταξης. Από την άλλη μεριά και οι πολιτικοί ηγέτες των, κρατών, ε, των υποψήφιων χωρών θα πρέπει να αποδείξουν ότι ε, είναι ικανοί και διατεθειμένοι να προβούν σε απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Ως συνεισηγήστρια ε, για το για το όργανο προενταξιακής ε, βοήθειας ε, θεωρώ ότι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να ε, επικυρωθεί και να επιβεβαιωθεί στη διαδικασία ένταξης. Το, τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν υιοθετηθεί από μια πλειοψηφία μελών και δείχνουν το δρόμο προς τις υποψήφιες χώρες. Ε, εμείς είμαστε υπέρ της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων και γι' αυτό το λόγο ελπίζουμε ότι τα ψηφίσματά μας θα εισακουστούν. Ευχαριστώ. Colleagues. Συνάδελφοι, παρακαλώ, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, το καταλαβαίνω ότι θέλετε να προλάβετε, αλλά έχουμε πολλού στη δικασία του ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Οπότε δεν θα προλάβουν όλοι. Γι' αυτό προσπαθείτε να τηρείτε του χρόνου. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Σίντερ. Ευχαριστώ πολύ. Τα Βαλκάνια είναι τμήμα τη Ευρώπη. και έτσι λοιπόν υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά κοινά σημεία βασικά. Κάποια λοιπόν από αυτά τα κοινά σημεία είναι αυτή η έντονη παρουσία της νεολαίας σε αυτή την περιοχή της Ευρώπης. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν τις μεταρρυθμίσεις και οι νέοι κανόνες λοιπόν που προτείνονται σήμερα ακριβώς αυτό έχουν ως σκοπό στο επίκεντρο είναι το κράτος του δικαίου, το rule of law, ε, η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωση, η ελευθερία έκφρασης, η ανεξαρτησία και η συμμετοχική δημοκρατία. Αλλά το κράτος του δικαίου είναι ισχυρό μόνο αν καταφέρουμε στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαλείψουμε κάθε αμφιβολία για την τήρηση του κράτους δικαίου. Αυτό τι σημαίνει αν η ανεξαρτησία λοιπόν της δικαιοσύνης, αν το κράτος δικαίου είναι αυτό που επιθυμούμε, θα πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα στο μέλλον. Καλωσορίζω λοιπόν τους νέους κανόνες που προτείνονται, γιατί είναι σαφείς, διαρθρωμένοι και λογικοί και θα οδηγήσουν σε πλειοψηφικές αποφάσεις ε, στο Συμβούλιο. Οι διαπραγματεύσεις λοιπόν με τη Βόρεια Μακεδονία, η οποία έχει κάνει τόσο μεγάλες και βαθιές ε, μεταρρυθμίσεις και με την Αλβανία θα μπορέσουν να ξεκινήσουν. Αυτό θα ήταν λοιπόν το πιο χειρό και σαφές μήνυμα το οποίο χρειάζονται τα Βαλκάνια. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό ο κύριος Αστροβίτσιους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Η διαδικασία διευρύνσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τα πιο ισχυρά εργαλεία που διαθέτουμε. Αν πετύχει η προτινόμενη μεθοδολογία για να εναρμονιστεί αυτή η διαδικασία διεύρυνση, αξίζει τον κόπο να την εγκρίνουμε. Ωστόσο, η επιτυχία δεν ε, μπαίνει σε μια έξυπνη μεθοδολογία. Είναι η πολιτική βούληση ισχυρή αυτή που καθορίζει την επιτυχία και από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει σαφή πρόθεση να διευρυνθεί η ευρωπαϊκή οικογένεια με μια προσδοκία, με μια φιλοδοξία φυσικά να πληρούνται όλα τα κριτήρια για την έναξη τη διαδικασία αυτή. Θα πρέπει να τριετήσουμε λοιπόν την ακυριότητα τη διαδικασία αυτή, γιατί θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι οι για όλε τι χώρε και οι υποψήφιε χώρε θα πρέπει να δουλέψουν σκληρά και άκοπα και να μην κάνουν συμβιβασμού αν θέλουν να πετύχουν την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται βέβαια, κατανόηση και εμπιστοσύνη. Είναι βασικέ προποθέσει αυτέ. Αυτή η στρατηγική λοιπόν προσέγγιση θα πρέπει να μην υπόκειται σε πολιτικέ χειραγωγήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φέστη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, γιατί οι Βρετανοί εγκατέλειψαν την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι ήθελαν την κυριαρχία της χώρας τους. Όμως, εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να οργανώσει κεντρικά και το δίκαιο και την βούληση των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν λειτουργεί όμως αυτό. Η ανεργία των νέων σε πολλές χώρες έχει φτάσει σε δραματικά επίπεδα. Και γι' αυτό εγκαταλείπουν πολλές περιοχές οι νέοι. Η διάσωση του ευρώ και η σχετική πολιτική των χαμηλών επιτοκίων έχουν φέρει σε δυσφορία πολλούς Ευρωπαίους. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι εσείς συνεχίζετε να προσποιήσετε ότι δεν υπάρχει το Brexit, δεν υπάρχουν τα κίτρινα γυλαίκα στην ε, Γαλλία. Ε, θα πρέπει λοιπόν ακριβώς να κοιτάξουμε ότι αυτά τα κράτη ζητούν την διαφάνεια και θα πρέπει να δούμε την διεύρυνση που ζητάτε για αυτά τα κράτη με υψηλά ποσοστά διαφθορά. Δεν μπορεί να πληρώνουν πάντοτε οι Ευρωπαίοι πολίτε. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σκεφτεί εάν η διεύρυνση χρειάζεται για την ύπαρξή τη, αλλά προτού βρείτε τέτοιε λύσει, λύστε τα εσωτερικά προβλήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ίσω να μην χρειαστεί αυτό που προσπαθείτε τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό, κυρία Σάλντε Μόζε. Ο κύριος Μάντλ, με συγχωρείτε. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε. Έχουμε χάσει τη Μεγάλη Βρετανία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Και αυτό αποδυναμώνει την Ευρώπη. Δεν θέλουμε να χάσουμε και τα Δυτικά Βαλκάνια τώρα. Τα Δυτικά Βαλκάνια ακόμη δεν είναι κράτη-μέλη, όμως ε, κατα... τρόπον τεινά είναι ευρωπαϊκά κράτη με ευρωπαϊκή ταυτότητα. Η νέα μεθοδολογία για την ε, διεύρυνση και την προσχώρηση νέων μελών ήταν ε, κάτι το επιπλέον, επιπλέον που έπρεπε να γίνει για τη το επέβαλαν μια μικρή μειονότητα κρατών μελών στο Συμβούλιο μπλοκάροντα την διαδικασία διεύρυνση και εκπλήσοντα όλου μα. Βεβαίω οι έξι χώρε πρέπει να κάνουν πολλά. Πρέπει να αλληλοβοηθηθούν περισσότερο. Πρέπει να καταπολεμήσουν τη διαφθορά. Όμω οι διαπραγματεύσει με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία πρέπει να ε, ξεκινήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα. ίσως και πριν τι εκλογέ στη Βόρεια Μακεδονία. Η ε, ε, σχέση με, το, με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο μπορούν να προχωρήσουν εφόσον η Σερβία αναγνωρίσει το κοσυφοπαίδιο και ε, πάψουν οι δασμοί που επιβάλλει το Κωσυφοπέδιο, βέβαια από την πλευρά του κατά τη Σερβία. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με άλλε περιοχέ του κόσμου, δίνοντα έμφαση σε αυτή τη διαδικασία διαβρύψη. Νομίζω, Επίτροπε και η Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσεί έχετε σωστά θέσει την κατεύθυνση για ε, ευχαριστούμε και ελπίζουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να γίνει ξανά μέλο κάποτε. Και τώρα για ένα λεπτό η κυρία Σάλντε Μόζε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ας ε, ξεκινήσω επενώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά τα μέτρα που προτείνει έτσι ώστε να προσαρμόσουμε την, την μεθοδολογία διεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να εστιάσουμε περισσότερο στο κατά πόσο οι υποψήφιες χώρες συμμορφώνονται με το κράτος δικαίου. Γιατί αυτό έχει αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητο. Δεν θα έπρεπε καν να ξεκινούν διαπραγματεύσεις αν δεν επικρατεί το κράτος δικαίου και πολύ δε περισσότερο να εντάσσεται μια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επίσης σημαντικό να μπορέσουμε να αποφασίζουμε να διακόπτουμε ε, προσωρινά ή μόνιμα τις ε, διαπραγματεύσεις αν αυτό χρειάζεται. Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνουμε και την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία. Ευχαριστώ. Ο κ. Γκρόσελ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση για την καινούρια μεθοδολογία ε, έχει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, αποτελεί ένα συμβασμό. Είναι ένα συμβασμό ο οποίο ενισχύει την Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργεί συνθήκε για την ε, περαιτέρω διεύρυνση και προκειμένου να αποφύγουμε τον μπλοκάρισμα. Ε, διευκολύνει τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν ε, και με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε και την υποστήριξη των πολιτών. Το... Υπάρχει όμως, υπάρχουν όμως και κάποια κράτη-μέλη τα οποία φοβούνται την διεύρυνση, ιδιαίτερα στα Δυτικά Βαλκάνια ε, όμως αυτή η μεθοδολογία προβλέπει, δημιουργεί με καλύτερη, ε, μεγαλύτερη αξιοπιστία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο προβλέψιμες διαδικασίες. Είναι σημαντικό αυτό το καινούργιο πλαίσιο που θα επιτρέπει να παρακολουθείτε καλύτερα η πρόοδος που επιτυγχάνεται και να ανταμείβεται όταν χρειάζεται. Οι υποψήφιες χώρες θα έχουν ένα πλαίσιο πολύ πιο συγκεκριμένο και προβλέψιμο για την προσέγγιση τους με, συγκεκριμένους και, με συγκεκριμένους και αυστηρούς όρους. Οι χώρες οι οποίες πληρούν αυτούς τους όρους θα μπορέσουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε κύριο Σκουμπίλιους για ένα λεπτό. Επίτροπε, πρόεδρε, είναι σαφέ ότι σε αυτό το σώμα η πλειοψηφία συμφωνεί ότι η διεύρυνση ήταν μια από τι πιο επιτυχημένε ευρωπαϊκέ πολιτικέ που έχει συνεισφέρει στο να διευρυνθεί ο χώρο δημοκρατία και ευημερία σε όλη την Ευρώπη. Η ευημερία ε, των Ευρωπαίων πολιτών θα ήταν, ήταν πάντοτε προτεραιότητα και θα είναι και θεμέλιο για τι μεταρρυθμίσει όλε μα τι χώρε. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που πρότεινε ε, ο Επίτροπο με την ανακοίνωση τη Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικώ, είναι μια πολύ καλή στρατηγική λύση και ε, βήμα πρόοδου. Θα γίνουμε αξιοπιστότεροι. Όμω η αξιοπιστία εξαρτάται και από το κατά πόσον θα περάσουν σε μεταρρυθμίσει οι ίδιε οι χώρε τη διεύρυνση. Και επίση από την υπευθυνότητα των κατών μελών θα εξαρτηθεί. Θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον ένα μόνο κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μπλοκάρει την διαδικασία διεύρυνση χωρί κανένα ε, τράνταχτο επιχείρημα. Θα πρέπει όλη η διαδικασία ψηφοφορία για τι διαδικασίε ψηφοφορία για τι διαδικασίε διεύρυνση, συγγνώμη, να γίνει πιο αξιόπιστη. Κύριε Επίτροπε, η δική σα ε, πρόταση θα έχει την ισχυρή στήριξη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό ο κύριος Ντέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, πρέπει να επενέσω την ταχεία και αποτελεσματική δουλειά τη δική σας και κυρίως τη δικιά σας, κύριε Επίτροπε Χαλπέη. Ε, και νομίζω ότι η διαδικασία διεύρυνσης του το 2020 θα είναι ε, καθοριστική. Μπορεί μέχρι το 2025 να πετύχουμε κάποια κράτη να είναι και έτοιμα για το επόμενο βήμα της διεύρυνσης. Βλέποντας αντιδράσεις αυτά τα επιμέρου κράτη-μέλη και ε, το πώ βλέπουν τη διεύρυνση. Υπάρχει θετική στάση η νέα πρόταση. Μπορεί να κάνει τι διαπραγματεύσει διεύρυνση πολιτικότερου χαρακτήρα αλλά και πιο αποτελεσματικέ. Ιδίω με τη βοήθεια των θεματικών ε, ε, συνόλων θεμάτων που θα επιτρέψουν να ανοίξουν συγκεκριμένα κεφάλαια και να απελευθερωθούν κονδύλια τα οποία θα φέρουν πραγματική διαφορά στην πράξη σε εταιρείε και πολίτε στι ε, συγκεκριμένε χώρε. Επίση, ε, πρέπει κάτι να γίνει και για χώρε όπω η Σερβία που έχει ήδη προχωρήσει αρκετά στη διαδικασία των δημοτεύσεων. Ο μηχανισμό των clusters των ομαδοποιημένων αυτών θεμάτων μπορεί να επιταχύνει τι διαδικασίε διεύρυνση, να επιλογήσετε στη στήριξή μα. Σα ευχόμαστε καλή τύχη. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε τον κατάλογο των αγορητών και περνάμε τώρα στη διαδικασία προσέλκυση τη προσοχή του Προέδρου. Αν όλοι παραμείνετε αυστηροί στο ένα λεπτό και το τηρήσετε, θα δώσω το λόγο σε όλου. Για ένα λεπτό, κύριο Σόκορ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αντιπρόεδρε. Και όντω, καλώ ορίσατε την πρόταση αυτή. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. και να κοιτάξουμε το χάρτη για να καταλάβουμε ότι είναι η μοναδική πλευρά της Ευρώπης, η οποία ως τώρα δεν έχει ενσωματωθεί ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι γειτονικέ χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολλά τα πολιτικά συμφέροντα στην περιοχή. Τουρκία, Ρωσία και άλλες ε, σημαντικές ε, χώρες. Και η ευρωπαϊκή προοπτική λοιπόν των χωρών αυτών είναι πολύ σημαντική γιατί ενισχύει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες αυτές. Ασφαλώς, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανεβόρων. Οι όροι είναι απαραίτητοι και θα πρέπει να δοθεί υποστήριξη στις κυβερνήσεις εκείνες οι οποίες είναι υπέρ τη Ευρώπης και το καταδεικνύουν αυτό με πράξεις, όχι μόνο με κενά λόγια. Κάρλος ορίζω λοιπόν την αξιοπιστία ως τη νέα αξία επικέντρωση τη πρόταση αυτή, γιατί είναι σημαντικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τι χώρε αυτέ. Συγγνώμη, λέει η Πρόεδρο, που σα διακόπτω, αλλά πρέπει να είμαστε δίκαιοι για όλου. Ο κύριο Μπερικλέ, λοιπόν, για ένα λεπτό, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Μετά τα ασφάλματα του Οκτωβρίου, όταν το Συμβούλιο μπλόκαρε τη διαδικασία διεύρυνση, η πρόταση αυτή για την ε, αναθεωρημένη διαδικασία διεύρυνση αποτελεί λογικό βήμα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώ, βλέπουμε ακόμα μία προσέγγιση από πάνω προ τα κάτω. Αυτό διατηρεί τι πολιτικέ ελίτ, οι οποίε σε κάποιε περιπτώσει είναι τμήμα του προβλήματο και όχι τη λύση. Δεν δίδεται επαρκή προσοχή στην κοινωνία των πολιτών και στους πολίτες τους ίδιους ο μεγαλύτερο ρόλο των κρατών μελών θα σημαίνει και μεγαλύτερη λογοδοσία. Θα πρέπει να καταδείξουν ότι πραγματικά είναι σοβαρέ οι προθέσει του ε, στην διάσκεψη των Βαλκανίων και ελπίζουμε να μην χρησιμοποιήσουν ε, την διεύρυνση για εσωτερικά πολιτικά συμφέροντα. Θα πρέπει όμως και η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει να παίζει με αυτή την προοπτική ε, ένταξη. Θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά την το κρατοδικαίου ως όρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φλέγκαλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, η πολιτική διεύνηση είναι μία από τις βασικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, καμία οργάνωση δεν προοδεύει αν απομονωθεί και σε αυτή την περίπτωση, αν απομονωθεί δηλαδή, καταραίει με το χρόνο. Οπότε χρειάζεται οι χώρε των Δυτικών Αλβανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζουμε ότι το πράσινο φω θα δοθεί πριν από την σύνοδο κορυφή του Ζάγκρεπ. Υποστηρίζω ότι αυτέ οι χώρε, όπω και άλλε χώρε που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να γίνονται δεκτέ και να στηρίζονται στι προσπάθειέ του. θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την υποστήριξη γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να εγγυηθούμε και την ειρήνη στα Δυτικά Βαλκάνια αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ευχαριστώ πολύ ο κ. Σουόλης για ένα λεπτό. Και εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διευκολύνει ε, τα, τους υποψήφιες, υποψήφιες χώρες και να τις κρίνει λιγότερο, να είναι λιγότερο επικριτική. Ε, η εσωτερική οργάνωση μπορεί να έχει ελλείψεις σε ορισμένες χώρες, αλλά αυτό ισχύει και στις δικές μας χώρες. Για παράδειγμα, η διαφορά είναι ε, πολύ έντονο φαινόμενο σε αυτές τις χώρες και το επικρίνουμε. Ε, αλλά δεν κάνουμε το ίδιο με την διαφθορά σε ανώτατου αξιωματούχου ή μέσα σε ιδιωτικέ επιχειρήσει στι δικέ μα χώρε. Για παράδειγμα, στην Ιρλανδία ε, είχαμε μια τράπεζα η οποία ιδιωτικέ επιχειρησεις στι δικέ μα χώρε. 20 δισεκατομμύρια στην χώρα επαιζε επεσε εξω κοστησε 20 κανένας δεν διώχθηκε. <laughs> Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συνεπείς ως προς το πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις χώρες. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε ο κύριος Μπασέσκου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να σας συγχαρώ, κύριε Επιτροπέ. Να σας συγχαρώ ε, για αυτήν τη νέα μεθοδολογία που προτείνεται για να προετοιμαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποδεχτεί νέα μέλη στους κόλπους της. Θα είναι πραγματικά ε, επιτυχημένη, πιστεύω. Απλώς επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Το καθοριστικό ζήτημα για τα κράτη αυτά είναι να ε, ξεβαστούν το κράτος δικαίου πλήρως προτού γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης τους επιβάλλουμε να περάσουν σε οικονομία αγορών. Ε, για να γίνεται αγωνιστική αγορά τους και να λειτουργεί εύρυθμα θα χρειαστούν πολλές προσπάθειες. Γι' αυτό το λόγο η διαφθορά η οποία είναι ορατή πρέπει να παταχθεί δεν μπορούμε να περάσουμε σε μαζικές μεταρρυθμίσεις χωρίς να υπάρχει ε, ένα ισχυρό κράτος δικαίου, ένα σύστημα δικαιοσύνης που να εποπτεύει τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Χάσολ. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, η Μακεδονία άλλαξε το όνομά της για να ικανοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και όμως δεν προσεκλήθησαν σε διαπραγματεύσεις διότι ο Γάλλος πρόεδρος ε, που τελικά υποστηρίχθηκε από τις κάτω χώρες ε, δεν ήθελε την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Πολύ κακό μήνυμα που στείλαμε σε αυτές τις χώρες. Γι' αυτό καλωσορίζω την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τουλάχιστον εν μέρη θα αποκαταστήσει την ε, αξιοπιστία μας ως μεγάλου παράγοντα και πρωταγωνιστή στα διεθνή πράγματα στην περιοχή και που θα επιτρέψει στις χώρες αυτές να γίνουν πλήρως μέλος ε, μέλη αφού πληρώσουν όλα τα κριτήρια. θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στην όλη διαδικασία και μεγαλύτερη σαφήνεια ώστε οι χώρε να γνωρίζουν ε, ακριβώ τι πρέπει να κάνουν σε κάθε στάδιο και να μην ευνηδιαστούν όπω το περασμένο φθινόπωρο όταν περίμεναν διακαώ την έναρξη των διαπραγματεύσεων και τελικά απογοητεύτηκαν. Ευχαριστούμε. Τσε για ένα λεπτό. Thank you, Welcome. Ευχαριστώ και Επίτροπε, καλώς ήρθατε στο Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη νέα μεθοδολογία για τη διεύρυνση που προτείνεται. Και χάρηκα που είδα ότι προτείνεται σε διάφορε περιπτώσει, αντικειμενικά κριτήρια για να εκτιμηθεί το κράτο δικαίου στι χώρε προσχώρηση. Πιστεύετε ότι τα κριτήρια αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθούν και τρέχοντα κρατημέλη, γιατί ξέρω ότι πολλοί στην Επιτροπή εργάζονται από αυτού. Ίσως θα μπορούσατε να μα βοηθήσετε. Δυστυχώ, ο υπουργό τη Ουγγαρία. Θα αφιέρωσω ένα ολόκληρο άρθρο στο Euronews για να πει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια για να αξιολογηθεί το κράτο δικαίου. Σω όμω θα μπορούσατε να την πείσετε γιατί ότι το αντίθετο. Κάποιε ερωτήσει έχω να σα κάνω. Κατά τη γνώμη σα, τι μπορεί να συμβεί αν ένα υφιστάμενο κράτο μέλο ε, ήταν πιο χαμηλά σε επίπεδο αξιολόγηση κράτου δικαίου σε σχέση με ψηφία χώρα και. Αν έχετε κάποια πρόταση για να διατηρηθεί το επίπεδο αυτό υψηλό μετά την ένταξη, για να μην υπάρχει επαναχώρηση στα δημοκρατικά ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντέλη. Για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και νομίζω ότι είναι κάπως ειρωνικό ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση μία εβδομάδα μόλις ε, αφού χάσαμε ένα μεγάλο κράτος μέλος και κοιτάμε μια νέα μεθοδολογία διεύρυνσης, ίσως η περίοδος περισυλλογής θα έπρεπε να είναι λίγο μεγαλύτερη. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, ξέρουμε ότι το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι ως κριτήρια ένταξης. Ξέρουμε όλοι ότι κάποιες χώρες παραβιάζουν τακτικά αυτά τα, αυτές και υπάρχει αυτή, αυτός ο νεοφιλελευθερισμός στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο οποίος ποτέ δεν παραβιάζεται. Επικρατεί πέραν όλων ο ανταγωνισμός. Αυτό δεν νομίζω ότι οφείλει τους Αλβανούς, τους ε, οποιοδήποτε άλλη χώρα, ούτε και την Βόρεια Ιρλανδία. Και αυτές οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές οδήγησαν στην αποχώρηση, να ψηφίσουν υπέρ της αποχώρησης πολλοί που ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ε, Ιστορική λοιπόν απόρριψη του νέου φιλελευθερισμού. Αν θέλουμε και εδώ κρίνει το μικρόφωνο η πρόεδρο. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριε Ζωή Τεβέζα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαγκίνες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσίασή σας. Ε, δεν έχω να φέρω αντίρρηση στη νέα μεθοδολογία, μου φαίνεται μια χαρά. Συμφωνώ επίσης με την πλειοψηφία ότι θα έπρεπε να δώσουμε πλέον πράσινο φως στην διαδικασία ένταξης της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας για, τη, για τους λόγους οι οποίοι αναφέρθηκαν. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη κάτι το οποίο ακόμα δεν ελέγχθη καθόλου ούτε από τον Επίτροπο την συνταγματική διάσταση της διεύρυνσης. Δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να διευρύνεται χωρίς να εμβαθύνεται ταυτόχρονα. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ε, να αντιμετωπίζουμε με τον κανόνα της ομοφωνίας στο Συμβούλιο πολιτικές όπως ε, η, πολιτική, εξωτερική πολιτική. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει ούτε με τους 27, αλλά δεν θα μπορεί να γίνει ούτε και με τους 29 ή 30. Ευχαριστώ. Κυρία Γιουβέρα. Είμαστε ε, όλοι λέμε το ίδιο πράγμα. Πόσο σημαντικό είναι να αναθεωρηθεί η διαδικασία και η μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς αυτή τη μεταρρύθμιση η διεύρυνση δεν έχει και νόημα. Είναι αλήθεια από την άλλη μεριά ότι η διαδικασία διεύρυνσης έχει τύχει κατάχρασης, κατάχρησης ε, στο παρελθόν. Ίσως είμαι αφελής, αλλά ελπίζω ότι σε αυτήν την καινούργια μεθοδολογία τα πράγματα θα αλλάξουν. Πιστεύω ότι πια ε, έχουν ε, ικανοποιηθεί όλοι οι όροι, ακόμα και για την Γαλλία, η οποία θα πρέπει να συνενέσει με το πράσινο φως στην Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Θέλω να δω πώς θα λειτουργήσει βέβαια στην πράξη, κύριε Επίτροπε, και αυτό θα το δούμε μόνο αν αυτές οι δύο χώρες ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Οπότε δεν είναι δυνατό να απαιτούμε χωρίς να ανταμείβουμε. Το λάθος του Οκτωβρίου ήταν υπεραρκετό. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον Επίτροπο κύριο Βαρχέλη για να απαντήσει. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την συζήτηση και για την ανανεωμένη προσήλωσή του στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι ένα θετικό μήνυμα το οποίο πρέπει να απευθυνθεί, να αποσταλεί στην περιοχή αυτή. Είναι σαφής, σαφές επίσης από τη συζήτηση ότι θέλετε να δοθεί στα Δυτικά Βαλκάνια μια αξιόπιστη ευκαιρία να ενταχθούν οι χώρες αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σημείωσα διάφορες ερωτήσεις για τη νέα μεθοδολογία και για το πώς αυτή συνδέεται με το ενδεχόμενο έναρξης διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Καταρχήν να πω ότι η νέα μεθοδολογία προτείνεται προκειμένου να, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με αυτές τις δύο χώρες. Βέβαια, αποτελεί ένα κομμάτι μιας συνολικότερης στρατηγικής που δεν θα αφορά μόνο αυτές τις δύο χώρες. Όταν σχεδιάσαμε αυτή την καινούρια μεθοδολογία, είχαμε σαφές στο μυαλό μας ότι δεν θα θέσουμε καινούργιες, καινούργιους όρους, καινούργιες προϋποθέσεις. Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε επί τη βάση των κριτηρίων της Κουπενχάγης. Δεν έχουν αλλοιωθεί. Δεν έχουν αλλοιωθεί. Αλλά θα εφαρμοστούν με καλύτερο τρόπο, πιο αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς εξαιρέσεις, μέσω καλύτερη συμμετοχής όχι μόνο των κρατών μελών αλλά και του κοινού των πολιτών μας. Η διαδικασία εξακολουθεί να παραμένει ως ανταποδοτική. Όταν οι υποψήφιες χώρες αποδίδουν θα ανταμείβονται. Αλλά και όταν υποχωρούν, όταν υπαναχωρούν σε σχέση με τις δεσμεύσεις τους και εμείς θα έχουμε το δικαίωμα να υποχωρήσουμε στις δικές μας. Η ιδέα είναι να αντιμετωπίσουμε τα ουσιαστικά θέματα καλύτερα, πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη διαφάνεια. Ερωτήθηκα πώς είναι δυνατόν να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις ένταξης με χώρες που έχουν υψηλή ανεργία. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και το τρίτο στοιχείο της ε, στρατηγικής του πακέτου Ζάγκρεπ είναι αυτό της οικονομικής ενίσχυσης, της οικονομικής ανάπτυξης. Θέλουμε να δημιουργηθούν καινούριες θέσεις εργασία έτσι ώστε οι οικονομίες τους να είναι σταθερές και ισχυρές. Ευχαριστούμε Επίτροπε και συνάδελφοι. Έχει λήξει η συζήτηση για το θέμα αυτό και θα αναλάβει ο επόμενος Αντιπρόεδρος. Καλό σας βράδυ. Καλησπέρα σας. Να συνεχίσουμε με την διεξαγωγή της Ολομέλειας. Έπεται η πρόταση, η δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μάλλον η προφορική ερώτηση για τις διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Όπως ξέρετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ηλεκτρονικά μέσα ή τα παραδοσιακά για να εγγραφείτε στη διαδικασία CatchDI ή για το σύστημα της γαλάζιας κάρτας. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και καταρχάς θα δώσω το λόγο στην συνάδελφό μας Πέτρα Ντεζούτερ. Για πέντε λεπτά έχετε το λόγο. Πρόεδρε, Επίτροπε, ε, κύριε Λεβρετό, συνάδελφοι, η Επιτροπή για την Εσωτερική Αγορά και την Προστασία των Καταναλωτών διατύπωσε μια διαρωτήση για την αυτοποιημένη λήψη αποφάσεων και τις σχετικές διαδικασίες προλαμβάνοντα τι πρωτοβουλίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τεχνητή ευθεία, οι οποίε θα υποβληθούν την επόμενη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο. Για την Επιτροπή μα είναι ύψη τη σημασία σε οποιαδήποτε μελλοντική πρωτοβουλία για το θέμα να μην διασφαλίσουμε απλώς την ελεύθερη κυκλοφορία των ε, εγκεκριμένων ε, αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και την προστασία και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε αυτά τα νέα αγαθά και υπηρεσίες επειδή είναι πολυάριθμα και πάμπολα αυτά που προσφέρονται και καλύπτουν όλους τους τομείς της εσωτερικής αγοράς, γινόμαστε μάρτυρες μιας γοργά μεταβαλλόμενης ε, τεχνολογίας ε, για τα θέματα τεχνητής ευθείας και οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με αυτοποιημένη λήψη αποφάσεων όπως την ε, βοήθεια που προσφέρεται στον καταναλωτή από ιστότοπους στο τηλέφωνο με αυτοποιημένα συστήματα. Αυτό έχει πολλές ευκαιρίες αλλά και ε, δημιουργεί και προκλήσεις. Η τεχνητή ευθεία δημιουργεί απαιτήσει και περισσότερα αγαθά και υπηρεσίε υψηλή ποιότητα, όμω θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να γίνουν όλα αυτά πράξη. Ε, είναι πολλά τα εργαλεία που χρησιμοποιούν τέτοια αυτοποιημένα αυτοματοποιημένα συστήματα όμω μπορεί να προκαλέσουν διακριτική μεταχείριση κατά των καταναλωτών, λόγω χάρη λόγω διαφορετικών τομολογίων. Θα γνωρίζουν οι καταναλωτέ ότι η τιμή που παρουσιάζεται στι οθόνε του έχει προσαρμοστεί στην ε, υπολογιζόμενη αγοραστική του δύναμη, το και για επαγγελματικέ υπηρεσίε. Εάν σημαντικέ αποφάσει είναι αυτοματοποιημένε και γίνονται χωρί την εποπτεία κάποιου ανθρώπου με υψηλά επαγγελματικά προσόντα, μπορεί να υπάρχουν δυσκολίε. Και επίση, ο επαγγελματικό, οικονομικό και οικογενειακό βίο των καταναλωτών μπορεί να επηρεαστεί και εάν οι καταναλωτέ αισθάνονται ότι δεν. Ε, οι καταναλωτέ ότι οι αποφάσει λαμβάνονται από μη ανθρώπινα όντα, είναι διαφορετικό. Όπω επίση το σε ποιον θα απευθυνθούν εάν έχουν κάποια αντίρρηση, διαφωνία ή παράπονο. Πώ θα μπορούν να αντιστραφούν οι αποφάσει. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι θα κάνετε για να προστατεύσετε του καταναλωτέ από αθέμητε ή λανθασμένε αποφάσει και από ε, υπηρεσίες που προσφέρονται από συστήματα τεχνητής ευφύειας. Επίσης, ξέρουμε ότι υπάρχει το πλαίσιο ποιότητας και αξιοπιστίας των ευρωπαϊκών προϊόντων, όμως δεν καλύπτουν τα προϊόντα τα οποία μπορεί να είναι ελαττωματικά ή να μη σέβονται όλες τις νομικές διατάξεις και ε, τα οποία παρέχονται από αυτοκομματοποιημένα συστήματα Τεχνητή ευθεία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με αυτά τα αγαθά και υπηρεσίε. Όπως για όλα τα αγαθά και υπηρεσίε, πρέπει οι εταιρείε και οι καταναλωτέ να προστατεύονται από επιζήμιε αποφάσει, από ε, λανθασμένες αποφάσεις για σκοπούς ελεύθερης κυκλοφορίας και δίκαιο ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι τι πρωτοβουλίε να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βεβαιωθούμε ότι το πλαίσιο αξιοπιστίας ε, και ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ε, σκόπιμο. Τι θα γίνει επίσης με τις αρχές εποπτείας της εσωτερικής αγοράς. Διαθέτουν αρκετά εργαλεία και μέσα για να δράσουν εφόσον χρειαστεί. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί οι αρμόδιες αρχές, οι επιχειρήσει και οι καταναλωτές δεν έχουν παντότε πρόσβαση σε σαφεί πληροφορίε για το πώ ελήφθη μία απόφαση, για την τεκμηρίωσή τη. Πώ θα βεβαιωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα υπάρχει διαφάνεια προ αυτό. Και εν τέλει, μιλώντα για προκαταλήψει ή για σύνολα δεδομένων που έχουν αποσπαστεί παρανόμω, η Επιτροπή μα τονίζει την ανάγκη ο Γενικό Κανονισμό ε, Προστασία Δεδομένων να γίνει σεβαστό σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα, αλλά και τη χρήση μη προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να υπάρχουν φραγμοί και προποθέσει. Πρέπει αυτό να το επιλύσουμε στη φάση του σχεδιασμού. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τις εγγύησει αυτές, το privacy by design, η ιδιωτικότητα και προστασία της ε, βάσει σχεδιασμού. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν να φροντίσει να χρησιμοποιούνται υψηλή ποιότητα και χωρί ε, προκαταλήψει ε, δεδομένα την παροχή υπηρεσιών και αγαθών τεχνητής ευφύειας. Θα επηρεαστεί η καθημερινότητα σε πολλού τομεί τη εσωτερική αγορά και θα έρθουμε αντιμέτωποι με πολλέ άγνωστε προκλήσει. Θα πρέπει λοιπόν να τι αντιμετωπίσουμε ε, εγκαίρω και καταλήλω. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών θα είναι καθοριστική για την αποδοχή αυτών των νέων τεχνολογικών μέσων στην κοινωνία μα και στην οικονομία μα μακροπρόθεσμα. Σα ευχαριστώ εκ των προτέρων για αυτό το τόσο επίκαιρο και κοινωνικώ ε, σημαντικό ε, ζήτημα. Εγώ και ολόκληρη Επιτροπή Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών αναμένουμε διακαώ τι προτάσει σα την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Και τώρα να καλωσορίσω τον Επίτροπο Τιερή Μπρετόν και να του δώσω το λόγο για τρία λεπτά. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Αντεσούτερ για την ερώτηση αυτή που δεν είναι απλώς μια ερώτηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των εργασιών μας ε, αυτά που κάνουμε δηλαδή τους τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες στην Κομισιόν σε ό,τι αφορά τα θέματα τα οποία σχολιάσατε και επίσης και όλα τα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη ε, που θα αλλάξει την εσωτερική μας αγορά. Η η ερώτηση που θέτεται στην πραγματικότητα σημαίνει πώς αυτή η εξέλιξη θα μεταλλάξει τις συμπεριφορές των καταναλωτών αλλά και πώς θα μας επιτρέψει να ε, ενισχύσουμε το σύνολο της εσωτερικής μας αγοράς. Η λέξη κλειδί είναι προφανώς η εμπιστοσύνη, το κλίμα εμπιστοσύνης, το είπατε κι εσείς. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή αμφιβολίες, δισταγμοί σε σχέση με την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Ε, λογικό είναι, εμείς έχουμε ως καθήκον να δώσουμε απαντήσεις. Η Κομισιόν, το υπενθυμίσατε, στις 19 Φεβρουαρίου θα παρουσιάσει μια λευκή βίβλο ε, σε μια στοχευμένη διαβούλευση ε, εκεί, σε αυτή τη λευκή βίβλο, θα καταγράψουμε τη δική μας θέση, αλλά θα δείξουμε και τους, τις κατευθύνσεις προς τις οποίες θα μπορούσαμε να κινηθούμε στο μέλλον. Θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε σχόλια και προτάσεις έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε μαζί αυτήν την τόσο σημαντική εξέλιξη για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει καταρχήν να θέσουμε τους κανόνες ε, ε, της ανάπτυξης της ε, τεχνητής νοημοσύνης στο σωστό τους πλαίσιο. Αυτή η συζήτηση θα μας επιτρέψει μέσω αυτών των κανόνων να διευκολύνουμε τη δημιουργία μιας ενός ευρωπαϊκού κλάδου ε, τεχνητής νοημοσύνης. Συνεργάζομαι με τους υπόλοιπους επιτρόπους τις τελευταίες εβδομάδες προς αυτήν την κατεύθυνση και θέλουμε όλοι μαζί να σκεφτούμε και το θέμα των αλγορίθμων, όπως είπατε, αλλά και το θέμα των δεδομένων. Γιατί τα δεδομένα είναι το καύσιμο, θα έλεγα, που θα μας επιτρέψει μέσω της χρήσης συγκεκριμένων αλγορίθμων να αναπτύξουμε ε, εφαρμογές ε, στην καθημερινότητα των πολιτών μας. Η σημασία λοιπόν που έχουν τα δεδομένα ως προστιθέμενη αξία είναι τεράστια. Για να απαντήσω ορισμένα από τα ερωτήματά σας, θέλω να πω το εξή. Δεν ξεκινάμε από μηδενική βάση. Έχει ήδη γίνει πολλή δουλειά. Νομοθετική δουλειά και με τη δική σα συμμετοχή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχήν έχουμε την νομοθεσία περί προστασία του καταναλωτή. Καλύπτει εμπορικέ πρακτικέ, οι οποίε περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις ε, διακρίσεων. Επίσης, ε, πρέπει να ενημερώνουν οι κατανοητέ όταν η τιμή είναι εξατομικευμένη μέσω ενός συστήματος αυτοματοποιημένη λήψης αποφάσεων. Θα πρέπει επίσης να γίνεται μια ανάλυση αντικτύπου όταν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να δημιουργήσει υψηλού κινδύνους στα δικαιώματα και τι ελευθερίε των ατόμων. Επίση υπάρχουν και, άλλε προποθέσει για παράδειγμα, στην στελέχωση ε, και στην ηλεκτρονική πρόσληψη, θα πρέπει εκεί να αποφεύγονται οι διακρίσεις από τους αλγορίθμους. Θα πρέπει αυτοί οι αλγόριθμοι να εντάξουν στο εσωτερικό τους το σύνολο των αρχών και των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η ανθρώπινη παρέμβαση, η οποία μία ακόμα φορά θα πρέπει να επιτρέπει στους πολίτες να ε, ε, προσφύγουν και να αμφισβητήσουν την αυτοματοποιημένη απόφαση. Χρειάζεται να εξασφαλίσουμε επίσης ε, την διαφάνεια σε οποιοδήποτε αλγόριθμους ή μηχανές αναζήτησης κάνουν επιλογή ε, συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Θα πρέπει να σκεφτούμε την προσαρμογή της οδηγίας που αφορά τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, αυτήν για τις μηχανές, για, τα, για το ράδιο εξοπλισμό, καθώς επίσης και στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, που θα είναι πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη της ε, τέχνητης νοημοθυσίνης. Ο, ε, γνωρίζετε ότι ήδη εξετάζουμε το θέμα των αυτοκινήτων που θα έχουν σύνδεση με το ίντερνετ Έχουμε την ε, γενική οδηγία ε, ασφάλεια των προϊόντων και σε σχέση με την τεχνητή και σε σχέση με την κυκλική οικονομία. Και επίσης έχουμε και τις προετοιμασίες που θα μας επιτρέψουν να εξετάσουμε τα ε, συστήματα διαμεσολάβησης, συστήματα συστάσεων που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, καθώς επίσης και τα συστήματα ηλεκτρονικής διαφήμισης. Για τις επαγγελματικέ υπηρεσίε θα πρέπει να μην βασιστούμε μόνο στα ε, παραδοσιακά προσόντα, αλλά σε μια, ε, σε, και σε καινούριους όρους όπως ε, η γνώση των ε, ηλεκτρονικών μέσων κλπ. Η λευκή βίβλος πάνω στην οποία εργαζόμαστε και την οποία σύντομα θα δημοσιεύσουμε, θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα στοιχεία προκειμένου να τα θέσουμε υπόψη σας και να συνεργαστούμε μαζί σας γιατί γνωρίζουμε ότι πολλοί και πολλές από εσά εργάζονται για αυτά τα θέματα εδώ και μήνες ή εδώ και χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό και χρήσιμο αυτό για μας. Μέσω της Λευκής Βιβλίου θα δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για να ε, ανταλλάξουμε απόψεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ. Να δώσω το λόγο τους αγορητές που έχουν εγγραφεί. Και τώρα ο συνάδελφος Αρίας Ετσεβαρία. Για 1,5 λεπτό. Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε την τεχνητή νοημοσύνη ως προτεραιότητα για αυτή την νομοθετική περίοδο. Γνωρίζουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλές εφαρμογές. Ε, και τεράστιο δυναμικό βελτίωσης της λειτουργία των οικονομιών μας και των κοινωνιών μας. Γι' αυτό και εξαιτία αυτού πράγματι πρέπει να τη θέσουμε ως πρώτη προτεραιότητα. Όμως, προσοχή, ήδη χάσαμε το τρένο του ψηφιακού ε, όταν παλιότερα ε, ηγούμασταν της αγοράς μέσω εταιρεών όπως η Nokia αλλά που κατέρευσαν επειδή η Ευρώπη έχασε το τρένο. Δεν θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο λάθος με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει να εγγυηθούμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Εμείς δεν είμαστε εδώ όπως οι Ασιάτες ή οι Αμερικανοί. Εδώ βάζουμε πρώτη-πρώτη ε, την διαφάνεια και την ιδιωτικότητα. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι θέλουμε να πετύχουμε. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το πετύχει και για ποιους λόγους με ποιου στόχου. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει αυτέ τι πρώτε τρει ερωτήσει πριν αναλάβει οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία. Η διαφάνεια θα πρέπει να είναι ακρογωνιαίος λίθος οποιασδήποτε πρωτοβουλία σχετικής με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί χωρίς αυτήν οι πολίτες μας δεν θα μας πιστέψουν, δεν θα μας εμπιστευτούν και θα χάσουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί να έχουμε. Μόνο αν προσέξουμε και δούμε τα πράγματα από τη σωστή οπτική γωνιά, θα μπορέσουμε η τεχνητή νομοσύνη να αναπτυχθεί επαρκώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα εδώ πέρα που θα ευνοήσει του Ευρωπαίου και τα συμφέροντά του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Λεϊτάου Μάρκες για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Η αυτοματοποιημένη ε, μάθηση ε, είναι κάτι το δύσκολο. Η τεχνητή ευθεία που θεωρούμε εύκολη δεν είναι έτσι. Όπως τα συστήματα που σκοπό έχουν να διακρίνουν κάποια λόγο, όμως το καταφέρνουν όχι γιατί ακριβώς ε, πρέπει, μπορούν να διακρίνουν δύο διαφορετικά ζώα μεταξύ τους λόγω χάρη βάσει των εικόνων, αλλά γιατί ε, μπορούν ε, να διαχωρίσουν τον ε, κότοπο στον οποίο ζουν. Έτσι χώρισαν τα ζώα που ζούσαν σε βάση από αυτά που ζούσαν σε χιόνια. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις ψηφιακές πλατφόρμες που λαμβάνουν αυτοματοποιημένες αποφάσεις. Για κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να μην είναι ε, ακριβώ, να, να, μην παρουσιάζονται όπω είναι στην πραγματικότητα, αλλά να είναι πιο φανερά από ό,τι άλλα που κρύβονται. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε ποιο είναι το συλλογικό όφελο από τη χρήση του και πώ μπορούμε να βελτιώσουμε τι δημόσιε υπηρεσίες μα. Εάν φροντίσουμε να λάβουμε κάποιε εγγυήσει, κάποιε διασφαλίσει ε, ηθικές ε, νομοθετικού χαρακτήρα και ρυθμιστικού μπορεί τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια για τους αλγορίθμους οι οποίοι επιτρέπουν ακριβώς ε, να λειτουργεί τεχνητή ευθεία. Θα πρέπει να γίνεται μια τεκμηριωμένη επιλογή από τους καταναλωτές και κυρίως να υπάρχει εμπιστοσύνη όταν υπάρχει η διάδραση των καταναλωτών με τα αυτοματοποιημένα συστήματα και να ξέρουν εάν μιλούν με ένα ρομπότ ή με έναν άνθρωπο που είναι πίσω από το σύστημα. Τα συστήματα αυτά λοιπόν πρέπει να διασφαλίζουν ε, καλή ποιότητα για τα προϊόντα και να γίνονται βεβαίως σεβαστοί όλοι οι κανόνες ε, επιθενότητας σε περίπτωση που υπάρχουν ε, ελαττώματα. Επίσης για τα δεδομένα, τις βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούνται για να εκπαιδευτούν αυτοί οι αλγόριθμοι το ε, κρίσιμο σημείο, όπως είπαμε, πρέπει να έχουν την απαραίτητη ποιότητα και πρέπει να ε, διέπονται από σαφείς κανόνες διαχείρισης για να είναι ε, ξεκάθαροι οι κανόνες που ισχύουν στο διαδίκτυο και να μην υπάρχουν παρεκτροπές. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε ένα σύστημα που ε, μας ε, προειδοποιεί ανάλογα με το αν βλέπει δάσος ή κάτι άλλο, αν πρόκειται για σκύλο ή λύκο και μας λέει να μην ανησυχούμε. Ευχαριστώ, θα σας παρακαλέσω να τηρείτε το χρόνο ομιλία σας και τώρα ο λόγος στην ε, Ντίτα Χαράντσοβα για δύο λεπτά. Thank you, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Καλώς ορίζω ιδιαίτερο το γεγονός ότι αυτό το νέο κοινοβούλιο θα εγκρίνει το πρώτο ψήφισμα για την τεχνική νοημοσύνη. Δεν θα είναι το τελευταίο, φαντάζομαι. Η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ήδη επηρεάζει τις ζωές μας. Κάνει τις ζωές μας πιο εύκολες, με νέες καλύτερες υπηρεσίε και διάφορες βαρετές δουλειέ που τις, ε, μας παίρνουν χρόνο, μας παίρνουν χρόνο αν ναι, γίνεται σωστά, έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν ε, την ανθρώπινη μεροληψία και το ανθρώπινο σφάλμα σε ό,τι αφορά σημαντικέ αποφάσει. Αλλά, όπω κάθε νέα τεχνολογία, θα πρέπει να κοιτάξουμε και τα νομικά και ηθικά ερωτήματα τα οποία ανακύπτουν. Τα πιο πολλά θέματα λοιπόν μπορούμε να τα επιλύσουμε με τους εφιστάμενους κανόνες, αλλά ενδεχομένως να πρέπει να τροποποιηθούν. Χρειάζεται όμως μία λελογισμένη προσέγγιση. Θα πρέπει να αντισταθούμε στον ε, πειρασμό να κάνουμε υπερβολική νομοθεσία υπερβολικά γρήγορα για αυτές τις ταχαίω αναπτυσσόμενε τεχνολογίες. Αυτό όχι μόνο θα ανακόψει την κοινοτομία και τις εξελίξεις στην Ευρώπη, αλλά θα δημιουργήσει και πιο πολλά προβλήματα από ό,τι θα επιλύσει. Αντίστοιχα, δεν θα πρέπει να γενικοποιούμε την προσέγγιση μα οι κανόνες σε ό,τι αφορά τους αλγοριθμούς θα πρέπει να είναι αναλογικοί με τον κίνδυνο που συνεπάγεται η χρήση του αλγοριθμού. Υπάρχει διαφορά μεταξύ του αλγορίθμου ενός δικτύου ενέργειας και του αλγορίθμου σε ένα video game. Και για να κλείσω στο σημείο αυτό, οι άνθρωποι πάντα θα πρέπει να είναι στην ηγετική θέση, αλλά ας ε, αφήσουμε να μας οδηγήσει η λογική μας και όχι ο παράλογος φόβος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και πάλι για δύο λεπτά. Ο λόγος στη συνάδελφο Βιζίνη Ζωγόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί. Έλεγε ο Εξυπηρή ότι τα μάτια δεν βλέπουν καλά. Είναι τυφλά. Θα πρέπει να κοιτάξουμε με την καρδιά. Σήμερα βλέπουμε λοιπόν στο ίντερνετ ρομπότ, αλγόριθμους οι οποίοι αναλύουν τα δεδομένα, κάνουν profiling και μας προτείνονται λοιπόν ταξίδια, σύζυγοι και διάφορα άλλα προϊόντα. Μπορούμε λοιπόν να εμπιστευτούμε αυτά τα δεδομένα, είναι οι κανονικές τιμές, είναι σωστές αυτές οι προσφορές. Είναι βασικό τα κριτήρια αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται από τους αλγοριθμούς να είναι διαφανή. Γιατί μπορούμε να έχουμε υπερβολικά μεγάλη εμπιστοσύνη ή υπερβολικά λίγη εμπιστοσύνη σε τέτοια αυτοματοποιημένα συστήματα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πού βάζουμε την εμπιστοσύνη μας αύριο θα δούμε ότι όλο και πιο πολλοί οδηγοί θα χρησιμοποιούν τέτοια δεδομένα και συστήματα και, και αν γίνει ένα τύχημα, ποιος θα έχει τελικά την ευθύνη. Οι καταναλωτές ε, θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να ακυρώνουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι αλγόριθμοι και τα ρομπότ. Σε ό,τι αφορά την πρόταση του λοιπόν αυτού του κειμένου, δεν μιλάει για τη συγκέντρωση των δεδομένων σε μη ευρωπαϊκές εταιρείε και την αντιμετώπιση του θέματος αυτού που είναι απαραίτητη. Δεν πιστεύουμε ότι οι καταναλωτές είναι επαρκώς προστατευμένος ε, σε ό,τι αφορά τα κενά της νομοθεσίας των Βρυξελών. Το ξέρετε εδώ και πλέον και 30 χρόνια ότι οι εταιρείε βάζουν με μικρά γράμματα διάφορα στοιχεία για αποποίηση της ευθύνη. Πιστεύουμε λοιπόν ότι δεν θα είναι πιο αποτελεσματικές οι Βρυξέλλες για τον καθορισμό των κινδύνων που προκύπτουν από τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στους Γάλλους μηχανικούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα για 1,5 λεπτό η Αλεξάνδρα Γκίζα. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, τα αυτόματα συστήματα λήψης αποφάσεων θα αποφασίζουν ε, κυριαρχικά για τη ζωή μας, για τη ζωή των παιδιών μας, ε, το επάγγελμά μας, ε, την εκπαίδευσή μας, το διαμέρισμα που θα πάρουμε. Όλα αυτά επηρεάζονται. Είναι δική μας όμως απόφαση τι επιρροή θα ασκήσουν, σε ποια ζητήματα, σε ποια δεδομένα καλούνται να αποφασίσουν οι μηχανές και τι αποφασίζουν και τι όχι. Θέλουμε να ωφελήσει η τεχνητή νοημοσύνη όλους μας και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε ένα σαφές ναι στην τεχνική, τεχνητή νοημοσύνη για τη βιωσιμότητα, για το κλίμα αλλά με ένα σαφές και χειρό όχι όταν υπάρχει διακριτική μεταχείριση των ανθρώπων γιατί Ξέρουμε ότι υπάρχει και αυτή η διακριτική δράση. Ένα παράδειγμα. Αν για κάποιος, για παράδειγμα, είναι σε μία χαμηλόμιστη θέση απασχόλησης, αυτό θα καταχωριστεί στο δεδομένο και στο μέλλον το άτομο αυτό, η γυναίκα για παράδειγμα, θα καταλήξει σε άλλη μια θέση χαμηλόμιστη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε το δικαίωμα για ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίε. Αυτό το δικαίωμα όμω το πρέπει να μπορούμε να το επιβάλλουμε και γι' αυτό χρειάζονται υποπτικέ αρχέ με ευρείε αρμοδιότητε για να μπορέσουν να ελέγχουν την νομιμότητα των αλγορίθμων. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, η Ευρώπη έχει τη μοναδική ευκαιρία σήμερα να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο ανταποκρίνεται στις δημοκρατικές μας αξίες και θα αποτελέσει υπόδειγμα για όλο τον κόσμο. Ας ε, αδράξουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία με το Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αλεξάνδρα. Να δώσω τώρα το λόγο στη συνάδελφο Κονέτσνα για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Επίτροπη, Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Η τεχνητή νοημοσύνη εκτελείστε και εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα και αυτό δημιουργεί προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από νομικής πλευράς πιστεύω ότι θα επηρεάσει πάρα πολύ το μέλλον της ανθρωπότητας και την εσωτερική αγορά. Και Υπηρεσίε και αγαθά τα οποία χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοπαντομημένη λήψη αποφάσεων δημιουργούν τα ίδια προβλήματα που δημιουργούνται στι κοινωνίε γενικότερα. Για παράδειγμα, κίνδυνο διακρίσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν οδηγεί εξορισμού σε μια βελτιωμένη κοινωνία, σε μια άψογη κοινωνία. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να βελτιώσει τη σημερινή κατάσταση. Τη σημερινή κατάσταση όπου βλέπουμε ε, τους ε, νόμους να τυχάνουν χάνουν καταχρήσεων κλπ. Θα πρέπει επίσης να προστατεύσουμε τους επενδυτές από ε, επαγγελματικέ υπηρεσίες οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει αυτή η λήψη αποφάσεων να είναι διαφανής, απόλυτα διαφανής και να παρακολουθείτε από τις κατάλληλες αρχές οι οποίες θα πρέπει να χρηματοδοτούνται και επαρκώς. Θα πρέπει να θέσουμε κανόνες για την ποιότητα των δεδομένων και να αποφύγουμε ε, την μεροληψία και τις διαστρεβλώσεις των δεδομένων. Ε, δεν θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να το σκεφτούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Ραντακόφσκι. Για ένα λεπτό. Στηρίζω το ψήφισμα του Κοινοβουλίου για τις ε, αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ε, είναι πολύ σχετικό αυτό το ψήφισμα με την ελεύθερη κυκλοφορία. Η 8534 εδώ και δεκαετίες ε, προστατεύει τους καταναλωτές από ελαττωματικά προϊόντα. Και θα πρέπει όμως τώρα να ξαναορίσουμε τους όρους όπως ελάττωμα, λάθος, βλάβη κλπ λαμβάνοντας υπόψη τις ε, καινούριες, την καινούρια κατάσταση. Θα πρέπει να ξαναορίσουμε ποιοι έχουν την ευθύνη, με ποιο τρόπο και ποιος φέρει το βάθος απόδειξης. Ο προμηθευτής θα πρέπει πάντα να έχει το βάρος απόδειξης. Η αναθεώρηση λοιπόν αυτή της ορολογία και αυτών των ορισμών θα είναι πολύ σημαντική στο μέλλον. Θα πρέπει να την κάνουμε με πολύ προσοχή και να αποφύγουμε τις πιέσεις από λόμπι είναι πολύ σημαντικό για την προστασία των καταναλωτών, οι οποίοι είναι πάντοτε οι πιο αδύναμοι στην αλυσίδα. Θα πρέπει επίση να δούμε ένα καινούριο ορισμό για το δικαίωμα επαναχώρηση, επιστροφή ε, των, ε, της δαπάνης ε, αποστολής ε, και άλλους σχετικούς όρους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος των Τόμισλαβ Σόκολ για σε λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην... Τις περασμένες δεκαετίες η τεχνολογία εξελίχθηκε με αλματώδεις ρυθμούς. Εγώ ανήκω σε νεότερη γενιά, αλλά κάποιες φορές πραγματικά και εγώ μένω άφωνος, ε, βλέποντας τι είχα στη θέση μου παλιότερα ως νέο και τι έχω τώρα. οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψη αποφάσεων μπορεί να μειώσουν το ποσοστό ανθρωπίνου σφάλματος, όμως επιτρέπουν να υπάρξουν και άλλες μορφές παραποίηση των ε, στοιχείων. Η αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, η αναγνώριση προσώπων, η αναγνώριση όψης. Αυτά είναι εξελίξει που ε, οφείλονται στην ε, τεχνητή ευθεία και μπορούμε να, μπορούν να μας ωφελήσουν και σήμερα. Όμως θα πρέπει να βρούμε και το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, διότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, το γεγονός ότι ήδη έχουμε ε, λήψεις και κενά στο νομοθετικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις. Δεν θέλουμε να αναχαιτήσουμε ή να βάλουμε τροχοπέδι στην ε, εξέλιξη της τεχνολογίας, ιδίως βλέποντας ότι η Ευρώπη εξελιξη της τεχνολογιας ιδίω μείνει πίσω σε σχέση με τις είπα και άλλες περιοχές του κόσμου. Όμως το πρόβλημα αυτό πρέπει να το επιλύσουμε. Δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί με τέτοια κατάσταση όπου η ανάλυση των προσωπικών δεδομένων κάποιων καταναλωτών να επηρεάζει την ζωή τους με τρόπο ζημιογόνο. Λόγου χάρη όσοι έχουν εξάρτηση από τον τζόγο να, να βλέπουν συνέχεια μπροστά τους νέες ευκαιρίες μόλις έχει αναλύσει ε, κάποιος αλγόριθμος τα στοιχεία τους. Αυτού του είδους δραστηριότητε πρέπει να καταπολεμηθούν. Και επίση τα ανθρώπινα όντα θα πρέπει πάντοτε να παραμένουν σε έλεγχο σε ό,τι αφορά την διαδικασία λήψη αποφάσεων. Έχουν την τελική ε, απόφαση. Δεν θα πρέπει να γίνουμε στερικοί φυσικά σε σχέση με την τεχνολογία και απλώ να αντιμετωπίσουμε όλε τι περιπτώσει παραποίηση ή χειραγώγηση των δεδομένων με τρόπο εξισορροπημένο, λαμβάνοντα υπόψη τα ανθρώπινα συμφέροντα. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα για ένα λεπτό η Κρίστελ Σάλντεμόζε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πάσα πιθανότητα για την ώρα έχουμε δει μόνο την αρχή της επίδρασης της τεχνητής ευφύειας στην κοινωνία μας. Η τεχνητή ευφυΐα προσφέρει πολλές ευκαιρίες αλλά έχει και πολλές παγίδες. Και όταν μιλάμε για καταναλωτές, νομίζω οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να απαιτούν να γνωρίζουν ποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί αυτοματοποιημένως ε, για λογαριασμό τους και ποιε βάσει των δεδομένων του. Είναι σημαντικό οι καταναλωτέ να γνωρίζουν ε, ποια δεδομένα του ε, τηρούνται. Και σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο μέλλον θα πρέπει να κοιτάξουμε να ενισχύσουμε την νομοθεσία προστασία των καταναλωτών. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη διαφάνεια, καλύτερη προστασία των καταναλωτών και κυρίω να βεβαιωθούμε ότι αυτέ οι διαδικασίε ε, λήψη αποφάσεων που είναι αυτοματοποιημένε είναι και αντικειμενικέ. Θα είναι βεβαίω ιδιαίτερα ενδιαφέρον Ακόμη και στη συνέχεια της θητείας μας που θα κοιτάξουμε την νομοθεσία για τις πλατφόρμες και τα portals να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αλλά θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στη διαφάνεια που προσφέρεται στους καταναλωτές. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Σεζουρνέ ναι, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε και για την εισήγησή σας. Ε, έχω ένα λεπτουδάκι, ε, γι' αυτό θα κάνω μόνο μια παρατήρηση και ε, μια ερώτηση. Η παρατήρηση είναι ότι πράγματι για πρώτη φορά στην ιστορία της βιομηχανικής επανάστασης υπάρχει κάτι που δεν το είχαμε σκεφτεί σε σχέση με τους κανονισμούς μας. Καινοτόμες λύσεις που προτείνονται από ιδιωτικέ εταιρείε. Σε αντίθεση με τι βιομηχανικέ επαναστάσει και τα κύματά του προηγουμένω, όπου το κράτο μπορούσε να καθορίσει τι δομέ, καθώ το κόστο των υποδομών ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Οπότε τώρα προκύπτει για μα το εξή ερώτημα πόσο μπορούμε να φτάσουμε σε λεπτομέρειε στην ουσία τη νομοθεσία, που θα πρέπει ίσω και ετησίω να αναθεωρείται δεδομένων των αγοργών εξελίξεων στον επίπεδο τη τεχνητή ευθεία. Γι' αυτό τίθεται και το θέμα τη εμπιστοσύνη, Εφόσον η χρήση καθορίζει την εξέλιξη τη τεχνολογία και το δημόσιο χρήμα ε, σπανίζει για την ε, πρόθεση νέων λύσεων, πρέπει να δούμε πώς ε, η χρήση από του καταναλωτέ επηρεάζει τι εξελίξει. Αυτό ακριβώ νομίζω ότι είναι και το κίνητρο πίσω από το ψήφισμα του να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπία μεταξύ τη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μα, τη εμπιστοσύνη ε, των πολιτών, τη κοινή γνώμη σε σχέση με τα νέα προϊόντα και υπηρεσίε και ε, πώ θα είμαστε οι πρωτοπόροι και όχι ουραγοί στην ψηφιακή επανάσταση ε, παγκοσμίω. Η Λευκή Βίβλο δίνει κάποιε πρώτε ιδέε και καλό θα ήταν να τα δούμε κατά όλα αυτά τα σημεία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω σε λίγε μέρε θα έχουμε τι πιο απτέ σα προτάσει και ανυπομονούμε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος ε, Τσούλο για ένα λεπτό. Εφόσον βρίσκεται στην αίθουσα. Μάλλον δεν βρίσκεται. Οπότε, επόμενος ή επόμενη Κυρία Τότα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επιτροπέ. Η ψηφιακή αγορά συνεπάγεται νέε ευκαιρίε για να ενδυναμώσουμε την οικονομία και για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωή χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη και χάρη στην αυτοματοποίηση. Οι κινητέ πλατφόρμε και οι αυτοματοποιημένε πλατφόρμε αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία λόγω των ψηφιακών υπηρεσιών και αυτό έχει να κάνει με όλους τους τομείς της οικονομίας. Σημαίνει μεγάλες ευκαιρίες αλλά και πολλές προκλήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ενημερώνουμε επαρκώς τους καταναλωτές για τις ικανότητες που υπάρχουν για να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις. Για παράδειγμα, όλο και πιο συχνά στον τομέα τον ιατρικό, τον τεχνικό, και ούτω καθεξής, ε, δεν είναι οι άνθρωποι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Λαμβάνονται αυτοματοποιημένα αυτές οι αποφάσεις, χωρίς παρέμβαση ανθρώπου. Μπορούμε να ζητήσουμε όμω, για παράδειγμα, έλεγχο και αναθεώρηση των αποφάσεων αυτών από έναν εμπειρογνώμονα. Είναι σημαντικό ότι ε, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η αυτοματοποιημένη αυτή τη δικασία δεν μπορεί ποτέ να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Θα πρέπει να λάβουμε και περαιτέρω μέτρα για να καταστεί η ψηφιοποίηση αποτελεσματική, προκειμένου τελικά ο πολίτης, ο καταναλωτής και οι μικρομεσαίε επιχειρήσεις να είναι στο επίκεντρο της ψηφιακη αγορα Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. επομενο ομιλητη η κυρία Εύελιν Γκέπχαρτ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μεγάλες είναι οι προκλήσεις που συνεπάγεται αυτή η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και όλα αυτά δεν είναι καθόλου ουδέτερα από μόνο τους. Ανακύπτουν μεγάλα παντελογικά ζητήματα τα οποία θα κληθούμε να τα, να τα απαντήσουμε. Και γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να τα συζητήσουμε από τώρα. Οι αλγόριθμοι επί των οποίων βασίζονται οι διαδικασίε αυτές δεν δημιουργούνται από μόνοι τους. Του δημιουργεί ο άνθρωπος, ο οποίος εξορισμού δεν είναι ουδέτερο και ο, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν δεν είναι ουδέτερο. Γι' αυτό λοιπόν ένα από τα βασικά ερωτήματα στο πλαίσιο αυτό είναι η διαφάνεια. Οι πολίτες, οι καταναλωτές να μπορούν να ξέρουν από πού προέκυψε ο κάθε αλγόριθμος και τι δεδομένα χρησιμοποιεί ο κάθε αλγόριθμος για να προσφέρει μια απόφαση από την οποία ε, εξαρτάται για παράδειγμα η αγορά ενός ψυγείου. Γιατί να προτιμήσω τη μία μάρκα και όχι την άλλη. Για να αναφέρω ένα επουσιώδες θέμα. Ε, σε ό,τι αφορά την αυτόματη οδήγηση, ένα αυτοκίνητο το οποίο στη Μεγάλη Βρετανία ε, λειτουργεί και οδηγεί από τα αριστερά θα έχει πρόβλημα προφανώ στην Ευρώπη και εδώ θα πρέπει να προσέξουμε σε ό,τι αφορά τη λήψη τέτοιων αποφάσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Μελχιόρ για ένα λεπτό, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα μιλήσω στα δανέζικα αν μου επιτρέπετε. Ε, ότι λάμπει δεν είναι χρυσός, οπότε υπάρχουν ε, διαδικασίες αυτοματοποιημένες λήψης αποφάσεων που δεν αποτελούν τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε δεν μιλούμε μόνο για την τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή, αλλά για όλες τις αυτοματοποιημένες ε, διαδικασίες λήψης αποφάσεων και ήδη χρησιμοποιούνται πολύ τέτοιε διαδικασίε, ε, θα πολλαπλασιαστούν στο μέλλον, καλό είναι αυτό, αλλά θα πρέπει το πλαίσιο να αφορά όλη την τεχνολογία, όχι μόνο για την τεχνητή νοημοθυσίνη που αποτελεί τμήμα όλου αυτού. Γιατί χρειαζόμαστε ένα γενικότερο πλαίσιο, γιατί η διαδικασία, με οποιαδήποτε απόφαση δεν είναι αλάνθαστη επειδή την έλαβε ένα υπολογιστή. Και οι υπολογιστέ κάνουν λάθη, όπω κάνουν λάθη και οι άνθρωποι. Γι' αυτό το λόγο η τεχνολογία πρέπει να είναι διαφανής. Ε, εντάξει, ακούγεται vintage έτσι να μιλάμε για κώδικα, αλλά η, ε, απόφαση ε, δεν πρέπει να λαμβάνεται από ένα κώδικα. Ο άνθρωπος θα πρέπει και πάλι να παρακολουθεί και να επεμβαίνει όταν χρειάζεται. Θα πρέπει οι αποφάσεις να είναι λογικές και να βασίζονται σε συγκεκριμένα λογικά επιχειρήματα και κανόνες. Θα πρέπει επίσης να μπορούμε να αμφισβητήσουμε μια τέτοια απόφαση. Θα ήθελα να ακούσω τις, αποφάσεις, τις απαντήσεις της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο λόγος του κύριο Πόσπισελ για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, Άκουσα με πολύ προσοχή την εισαγωγή του Επιτρόπου. Πολύ καλά που προετοιμάζετε την Λευκή Βίβλο για την τέχνη νομοσύνη. Ε, παρακολουθούμε στενά το θέμα στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Είναι πολύ σημαντικό το ότι ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση η Κομισιόν. Το είχαμε συζητήσει βέβαια το θέμα αυτό ε, με πιο συγκεκριμένο όμως τρόπο, συγκεκριμένους τομείς και κλάδους κλπ. στην προηγούμενη θητεία. Ε, το είχαμε συζητήσει για παράδειγμα σε σχέση με τα ε, αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Τώρα θέλουμε ένα γενικότερο πλαίσιο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα καθορίζει συγκεκριμένους κανόνες για θέματα τεχνητής νοημοσύνης, προστασία του καταναλωτή, για παράδειγμα, είναι ένα κεντρικό σημείο. Ε, νέοι κανόνες για την νομική ευθύνη. Ποιος είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε βλάβη η ζημία προκύψει στον καταναλωτή από προϊόντα τα οποία έχουν ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απάντηση σε όλα. Έχουμε κάποιες απαντήσεις ήδη στην νομοθεσία μας, αλλά χρειαζόμαστε ένα γενικότερο πλαίσιο. Δεν είμαι υπέρ της ε, υπερβολικής νομοθέτησης, αλλά είμαι πεπισμένος ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ σημαντικό να ενταχθούν σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο ε, που θα καλύπτει και τα αγαθά και τις υπηρεσίες έτσι ώστε να εξακολουθήσει να αναπτύσσεται αυτή η τεχνολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λόγω στον κύριο Μπονιφέη. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι διαδικασίε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων από αλγοριθμούς έχουν όλο ένα μεγαλύτερο ρόλο στι κοινωνίε και τη ζωή μα. Γι' αυτό θα πρέπει να ληφθεί, για να υπάρξει μάλλον μια ταχεία και αποτελεσματική απόφαση, πρέπει να ληφθούν και δραστικά μέτρα για την προστασία των καταναλωτών, ιδίω των πλέον ευπαθών, οι οποίοι ε, μπορεί να πληγούν από ασφαλμένη λήψη απόφαση στον ιατρικό κλάδο ή για ένα ελαττωματικό προϊόν ή σε κάτι που αφορά τα τραπεζικά του. Θα πρέπει οι αλγόριθμοι να είναι μερόληπτοι και αντικειμενικοί, γιατί ε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να λάβουν υπόψη την πολυμορφία των ε, κοινωνιών μα και θα πρέπει και τα δεδομένα που χρησιμοποιούν να διαρκώ επικαιροποιημένα, αλλά και οι καταναλωτέ μα να γνωρίζουν ακριβώς ε, τι ε, αποφάσεις έχουν ε, ληφθεί, να μην είναι μετάκλητες οι αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί από άνθρωπο και να έχουμε τις απαραίτητες διατάξεις και κανόνες, τις ρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν την προστασία των καταναλωτών. Η ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία είναι απαραίτητη, αλλά θα πρέπει να ξεκινάει από τα πρόσωπα και όχι από το κέρδος. Θα πρέπει λοιπόν ο Επίτροπος Μπρετών να εργαστεί άοκνα για να γίνουν σεβαστές αυτές οι αρχές. Ευχαριστούμε. Και τώρα στη διαδικασία Catch the Eye, δύο εγγραφές μόνο να έχουμε. Να ξεκινήσω από τον συνάδελφο Πόλτσακ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να πω ότι καλώ ορίζω τη συζήτηση αυτή. Αυτή τη συζήτηση η οποία ξεκίνησε από την εισηγήτρια και μου άρεσε προσέγγιση. Σε ό,τι αφορά την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, έχει ε, κάποια ε, προτερήματα και πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά τις σύγχρονες τεχνολογίες και μπορούμε να συνεχίσουμε. Παρά όλα αυτά θα πρέπει να κοιτάξουμε και τους κινδύνους και τα μειονεκτήματα της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων. Γιατί? Συνεπάγεται αυτό είναι ανάγκη για την τελειότητα των αλγορίθμων αυτών και των ε, συστημάτων αυτών. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ε, ευθύνη της κύρωσης. Εμείς προφανώς και θα δώσουμε το παράδειγμα για πολλά κρατημέλη. Είναι καλό λοιπόν που υπάρχει αυτή η λευκή βίβλος και καλωσορίζω τη συζήτηση αυτή ε, εξ αρχής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φλέγκο. Για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, επίτροπε. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ως στόχο να δώσει καλύτερη ζωή σε όλους μας και καλύτερες υπηρεσίες και αφορά όλους μας σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, την γεωργία, το μάρκετινγκ. αυτή είναι οι τομή στου οποίου ε, βλέπουμε πιο έντονα την τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, οι καταναλωτέ θα πρέπει να είναι σίγουροι για τον τρόπο διοργάνωση τη λήψη αποφάσεων και θα πρέπει να εμπιστεύονται τη διαδικασία λήψη αποφάσεων και γι' αυτό θα ήθελα να προτείνω μία νέα ετικέτα αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία αυτή, αλλά επίσης να υπάρχει και μία ένδειξη και ένα σημάδι διαφάνειας. Είναι σημαντικό αυτό για την προσωπική ελευθερία όλων των ε, καταναλωτών. Η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να αποτελέσει μία ευπρόσδεκτη καινοτομία, η οποία θα βασίζεται όμως στην εμπιστοσύνη και δεν θα ενέχει κίνδυνο χειραγωγής. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Πατρίκ Ρέγερ θέλει το λόγο, πρόσθετος τελευταία στιγμή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κώδικας είναι νόμος. Αυτό που είναι εγγεγραμμένο στις μηχανές ε, είναι κάτι που ε, ουσιαστικά λειτουργεί ως νόμος, οπότε κάτι που είναι λανθασμένο εγγεγραμμένο είναι κακός νόμος στην πραγματικότητα. Δεν θέλουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου οι αλγόριθμοι πραγματικά ε, λαμβάνουν λάθος αποφάσεις. Θα πρέπει να κοιτάξουμε οι αλγόριθμοι να τίνουν προς συγκεκριμένες αποφάσεις ή να υποστηρίζουν αποφάσεις που βασίζονται σε τεκμηριωμένες ε, αποφάσεις. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τέτοιες περιπτώσεις διότι ο αριθμός δείχνει ότι ε, πολλές φορές μέχρι ε, τώρα οι αλγόριθμοι βρίσκουν αποφάσει και καταλήγουν σε αποφάσει που είναι παρόμοιε με του ανθρώπου. Όμω πρέπει να υπάρχει απαραίτητη διαφάνεια για να βεβαιωθούμε ότι οι αυτοματοποιημένες αποφάσεις είναι γνωστές και στους καταναλωτές. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει διαφάνεια και εκεί όπου οι αλγόριθμοι επηρεάζουν τις αποφάσεις ε, των ανθρώπων. Δηλαδή ένας άνθρωπος να γνωρίζει ε, τι απόφαση λαμβάνει και ότι αυτή βασίζεται σε πρακτικά δεδομένα και όχι μόνο σε θεωρίες ή ε, σε αφηρημένα δεδομένα. Ευχαριστούμε και τώρα για να κλείσει η συζήτησή μας ο λόγος των Επίτροπο Μπρετών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρίε και κύριοι βουλευτέ. Ειλικρινώ, δεν γνωρίζω πολλά κοινοβούλια παγκοσμίω όπου μπορεί κανεί για τέτοια θέματα τη σήμερον ημέρα να έχει τέτοιας, τέτοια ποιοτική συζήτηση πέραν των ε, διαφορών μας ε, λόγω των ε, κομματικών διαφωνιών έχουμε εν γέννη τις ίδιες, τα ίδια ερωτηματικά, τις ίδιες επιθυμίες, τις ίδιες, την ίδια βούληση. Και αυτό που θα κρατήσω την όλη συζήτηση είναι ένα πράγμα. Η εξέλιξη είναι ένα πράγμα. Η πρόοδος θα κρατήσει ίσως χρόνια και δεκαετίες ακόμα. Αυτό όμως που συμμεριζόμαστε όλοι εδώ στο Κοινοβούλιο ε, και μαζί σας ε, και ολόκληρη η Επιτροπή είναι η κεντρική θέση του ανθρώπου, του ανθρώπινου παράγοντα, του σεβασμού στις αξίες μας, του σεβασμού σε αυτό που πραγματικά είμαστε, την ακαιρεότητα των αποφάσεών μας, την ε, κατανόηση που θα πρέπει να υπάρχει των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα γύρω μας. Η κατανόηση και αντίληψη των καταστάσεων τι γίνεται, ποιο λαμβάνει απόφαση. Θα επηρεάσει αυτό τη ζωή μου, μπορώ να παρέμβω και να αλλάξω τα πράγματα. Μπορώ να στραφώ σε κάποιο όργανο που θα λάβει μια απόφαση την οποία δεν ήθελα, που έχει για κάποια απόφαση που έχει ληφθεί και που δεν ήθελα. Όλα αυτά ακριβώς θα περιλαμβάνονται στη Λευκή Βίβλο μας, κύριε και κύριοι βουλευτές που δεν το είπε ε, θα είναι ε, το θέμα τη η τεχνητή ευθεία μεν, αλλά η αρχή τη όλη μα συλλογιστική και μελέτη. Διότι αυτό που θέλουμε εμεί είναι να σκεφτούμε την αναδιάρθρωση ενό νέου χώρου. Ένα χώρου όπου πλέον καλούμαστε να εργαστούμε. ενός χώρου όπου θα πρέπει να μπορούμε να ε, σταθούμε και να ψυχαγωγηθούμε, να επικοινωνήσουμε. Δηλαδή το χώρο της πληροφορικής. Αυτό στην ουσία έχει να κάνει και με τους τρεις παράλληλους χώρους που παράλληλα συνεισέφεραν στο να διαμορφωθεί η σημερινή μας ταυτότητα και το πώς έχουμε διοργανωθεί ως κοινωνία. Πρώτα απ' όλα ο χώρος ε, ως ε, επικράτεια, ε, ο θαλάσσιος χώρος και ο εναέριος και τώρα και ο ψηφιακός. Ναι, η τεχνητή ευφυΐα είναι ένα από τα πρώτα στοιχεία και θα ε, περάσω και σε μια δεύτερη διατύπωση, διαπίστωση στην οποία κατάληξατε όλοι. Και είναι ένα αγώνα που τον έχω δώσει και εγώ στο παρελθόν και τον συμμερίζομαι. Ε, μέσα από τι ε, εφαρμογέ που θα πρέπει να διαχειριστούμε μελλοντικά και που θα καθορίζουν τι αποφάσει τη ζωή μα, τι αποφάσει τη τεχνητής ευφυία, αυτέ που πρόεδρε, τη είπατε αυτοπατοποιημένη λήψη αποφάσεων. Ε, εδώ υπάρχουν δεδομένα και αυτά τα δεδομένα ε, το λέμε όλοι μας, Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα, δεν έχουμε και τεχνητή θεία. Έχουμε την τάση να επικεντρωνόμαστε στους αλγορίθμους, τους κώδικε, ε, τι γραμμές κωδικών, όπως είπατε. Ίσως αυτό να μην είναι το μόνο. Όταν θα χρησιμοποιείται η κβαντική πληροφορική, ίσως τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Αλλά σήμερα αυτές οι γραμμές μας επιτρέπουν να εργαζόμαστε με την στενή συνεργασία αυτού του περιβάλλοντος με, τους, με τις μηδενικές γραμμές και την ε, εξέλιξη των υπόλοιπων για να καταλήξουμε στην απόφαση. Πέρα από αυτά όμως υπάρχουν τα δεδομένα. Το είπαν αρκετοί από εσά. Το είπαν και μάλιστα με την αλληγορία του λύκου και του σκύλου στο δάσος. Τι θέλετε να πείτε με αυτό. Ε, ότι όταν παίρνουμε δεδομένα που χαρακτηρίζουν ένα ζώο στο φυσικό χώρο κατοικίας του και πάρει κανείς το ίδιο ζώο σε ένα άλλο περιβάλλον, θα προκύψουν διαφορές. Διαφορές ως προς την ε, λειτουργία και την εφαρμογή των αλγορίθμων. Άρα και την διαδικασία που ονομάζουμε εκμάθηση, μηχανική εκμάθηση, machine learning. Βεβαίως, τα δεδομένα είναι καθοριστικά και αυτό είναι και ο αγώνας που θέλουμε να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. μεσά στο πλευρό μας, για να καθορίσουμε πώς αυτά τα δεδομένα θα χαρακτηρίσουν κι άλλο την ευρωπαϊκή κοινωνία και ταυτότητα. Και το είπαν κι άλλοι εδώ στην Ολομελία. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτό το τεχνολογικό άλμα και αυτή την ευκαιρία. Δεν νομίζω ότι έχουμε καθυστερήσει ω προ τι τεχνολογικέ εξελίξει. Δεν έχουμε χάσει χρόνο, αλλά σε αυτό το βήμα, σε αυτό το στάδιο πάλι δεν πρέπει να καθυστερήσουμε. Έχουμε δεδομένα μπροστά μα που θα μα επιτρέψουν να τροφοδοτήσουμε ευθεώ τι μηχανές τα δεδομένα που ε, συμπεριέχουν, ε, που ε, εκφράζουν τις αρχές και τα, τις αξίες μας. Πρέπει λοιπόν να δούμε και τα B2B, τα δεδομένα από επιχείρηση προ επιχείρηση, τα δημόσια δεδομένα, αυτά που αφορούν τον οικονομικό τομέα που είναι τόσο σημαντικά για όλου μα, τι μεταφορέ. Όλα αυτά ε, είναι μπροστά μα, είναι το μέλλον μα. Και το ξαναλέω, στου επόμενου 18 μήνε, το σύνολο των δεδομένων που αποτελούν τον ψηφιακό, το ψηφιακό χαρτοφυλάκιό μα θα έχουν διπλή αξία. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ταχύτητα που ήδη έχει αναπτυχθεί. Και θα πρέπει ακριβώ αυτό να δείτε ότι θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πολλά στοιχεία Πρώτον, ότι θα πρέπει να μην διευθετήσουμε από τώρα την έκβαση, γιατί τώρα μιλάμε απλώ για, για την τεχνητή ευφυα, αλλά θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη διαχείριση των δεδομένων. Όμω πρέπει να προσέξουμε σε σχέση με όσα θα προκύψουν. Όλα θα πρέπει να είναι συμβατά με τι δικέ μα αξίε. Την ελευθερία των πολιτών να επιλέξουν αυτό ακριβώς που λέω. Επιλογή. Ελεύθερη επιλογή. Όχι να είμαστε ε, όμοιροι ενός αλγορίθμου, κάποιου που διαχειρίζεται τα δεδομένα μιας πλατφόρμας. Όχι. Να έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε την ε, ελεύθερη επιλογή μας. Αυτό είναι ελευθερία στον χώρο της πληροφορίας. Πρέπει να εργαστούμε. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να εξεύρουμε λύσεις. Αυτό ακριβώς είναι και ο αγώνας μας. Και θα πρέπει εν τέλει να έχουμε τη δυνατότητα να γίνει αυτό σε απόλυτη ασφάλεια. Ασφάλεια νομοθετική, ε, ασφάλεια ηθική και βεβαίως στον κυβερνοχώρο. Ε, άκρο σημαντικό. Πρέπει λοιπόν με αυτήν την όλη συλλογιστική που έχουμε να σας προτείνουμε να δούμε και τις απαραίτητες υποδομές. Υπάρχουν υποδομές που επιτρέπουν να διαρθρωθούν αυτές οι ε, εφαρμογές σωστά. Επιλογές ευφυείς, επιλογές που κάνουν τη σωστή, λαμβάνουν τη σωστή απόφαση. Αυτέ θα πρέπει να υπερέχουν. Ε, δηλαδή, ε, μηχανές που θα χρησιμοποιούν για να σκηθούν αυτά τα δεδομένα. Πρέπει να έχουμε αυτή τη δυνατότητα να κοιτάξουμε επίση τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον από τη σκοπιά τη κατοχή των δεδομένων και να κοιτάξουμε να κάνουμε εμεί τη διαφορά. Δηλαδή να έχουμε τη δυνατότητα τη ελεύθερη επιλογή σε όλη αυτή την αλυσίδα παραγωγή και αυτό θα καθορίσει ακριβώ και ένα μεγάλο μέρο τη ζωή μα. Γιατί είμαστε άκρο προσεκτικοί ώστε αυτή η σφυριλάτηση του τέταρτου ψηφιακού χώρου να έρθει και να εδρεωθεί στο βάθρο και στο θεμέλιο των αξιών που καθορίζουν την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Ευχαριστούμε, Επίτροπε, για την τόσο ενδιαφέρουσα ομιλία σας. Και τώρα να σας ενημερώσω ότι έλαβα πρόταση ψηφίσματος ε, για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση και η οποία, το οποίο ψήφισμα θα ψηφιστεί την Τετάρτη. Ολοκληρώνουμε εδώ την εξέταση αυτού του σημείου της ημερήσιας διάταξης και ας περάσουμε απευθείας στο επόμενο. Έπεται δήλωση της Επιτροπής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βελτίωση της νομοθεσίας. Η συζήτηση θα ξεκινήσει και πάλι με την ομιλία του κυρίου Μπρετόν. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, περνάμε στον κόσμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, Παρ' όλα αυτά, η μετάβαση από το ψηφιακό κόσμο, τον κόσμο των δεδομένων, ε, θα επηρεάσει πάρα πολύ τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Οπότε αυτή η μετάβαση πρέπει να πω ότι είναι ομαλή από το ένα θέμα στο άλλο. Η πρόεδρος Κομισιόν, κύριε Φοντερ Λάιεν, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθύμησε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν ε, ό,τι είναι καλό και απαραίτητο στην οικονομία μα. Τα νούμερα τα γνωρίζετε. Είναι ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων από άντρε και γυναίκε επιχειρηματίε. Σχεδόν όλοι έχουν δημιουργήσει τη δική τους επιχείρηση και εργάζονται μέρα και νύχτα για αυτή την επιχείρηση. Ε, έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμα και εμπόδια τα οποία δικό μας καθήκον είναι να τα άρουμε. Το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα των θέσεων εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει να τις φροντίσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Οπότε στο πλαίσιο των δικών μου ευθυνών, εσωτερική αγορά, είναι ένα κρίσιμο στοιχείο έτσι ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να υποφεληθούν και αυτές των τεχνολογιών για τις οποίες μιλούσαμε, αλλά και να συμμετάσχουν στην νέα πράσινη συμφωνία, στην κυκλική οικονομία, στην πράσινη οικονομία κλπ. Για να βοηθήσουμε λοιπόν Τη μικρομεσαία επιχείρηση. Καταρχήν να πω ότι ένα σημαντικό στοιχείο ε, είναι ότι η πρόεδρος της Κομισιόν μου ζήτησε να ορίσω, να διορίσω έναν απεσταλμένο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έτσι τον λέμε εμείς στην Κομισιόν, που θα μου επιτρέψει να συνδεθώ, θα είναι δηλαδή ο σύνδεσμός μου με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι ώστε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν να φτάνουν στα αυτιά μου, να φτάνουν στο γραφείο μου. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να τις απελευθερώσουμε, να χρησιμοποιήσουν το δυναμικό τους και την ενέργειά τους για να ανθίσουν. Θα πρέπει βέβαια να βελτιώσουμε και την ομοθεσία. γιατί αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια που τις φρενάρουν, τις περιορίζουν και ταυτόχρονα περιορίζουν και την ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς. Καλύτερη νομοθεσία σημαίνει επίσης να εφαρμόσουμε το one in, one out. Όταν προτείνουμε μια καινού, ένα καινούριο νομοθετικό κείμενο να αναιρούμε και ένα παλιότερο. Το πρόβλημα προφανώς δεν είναι να μειώσουμε ε, υπερβολικά την νομοθεσία. Θέλουμε απλώς η νομοθεσία να είναι πιο ευέλικτη, πιο προσαρμοσμένη στις ανάγκες και στο περιβάλλον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σήμερα. Σήμερα όπου επικρατεί, επικρατούν οι ψηφιακές τεχνολογίες και επιφέρουν τεράστιες αλλαγές και στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Δημιουργούν καινούργιες σχέσεις μεταξύ προμηθευτών και πελατών. Το τεστ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί τμήμα της ε, τακτικής αξιολόγησης ε, αντικτύπου. Πάντοτε θα πρέπει να διατηρούμε αυτό που λειτουργεί σωστά και να διορθώνουμε αυτό που δεν λειτουργεί σωστά. Και αυτό το τεστ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα το αναπτύξω ακόμα περισσότερο με τη βοήθεια του απεσταλμένου ΜΜΕ νέα στρατηγική επί της εργαζόμαστε, την οποία επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή για τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα δώσει μια πιο ισχυρή φωνή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ε, στην πρωτοβουλία βελτίωση νομοθεσία Και θα προτείνουμε και μια σειρά δράσεων προ αυτήν την κατεύθυνση. Συνεργαζόμαστε στενά με τον Επίτροπο Σεύκοβιτς για αυτό το θέμα. Η πρόθεσή μας είναι όλες οι πρωτοβουλίες της Κομισιόν να βασίζονται στην αρχή του σκεφτόμαστε καταρχήν ε, σε, μικρή διάσταση ε, να σκεφτόμαστε το μικρό πριν πάμε στο μεγάλο. Θα δώσουμε ακόμα περισσότερη σημασία στην σορευτική, στο σορευτικό αντίκτυπο των νομοθετικών κειμένων που υιοθετούμε. Και εγώ ίδιο δημιούργησα μια μικρομεσαία επιχείρηση κάποτε. Όχι χτε προχτέ, παλιά. Αλλά γνωρίζω πώ είναι να αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι με το κεφάλι κάτω από την επιφάνεια τη θάλασσα, μέσα στο νερό και να πνίγεσαι. Θα πρέπει να το αποφύγουμε αυτό, να το αλλάξουμε. Έχουμε την εξαιρετική τύχη να διαθέτουμε μια εσωτερική αγορά 450 εκατομμυρίων καταναλωτών που διέπεται από κοινέ αξίες, από κοινά, κοινό πάθος και από κοινούς κανόνες. Είναι η αγορά μας. Πολλοί μας ζηλεύουν γι' αυτό. Και αυτό κάνει τη διαφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι υπάρχει αυτή η εσωτερική αγορά οδηγεί πολλούς να χτυπήσουν την πόρτα μας. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διαδώσουμε τις αξίες μας. Η κοινή αγορά, η ενιαία εσωτερική αγορά είναι και το εργαλείο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παρ' όλα αυτά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πολλά εμπόδια μπροστά τους. Δύσκολα πολλούν τα προϊόντα τους εκτός των συνόρων τους. Το γνωρίζω προσωπικά. Οπότε θα πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ εντατικά σε αυτήν την κατεύθυνση. Να αποφεληθούμε Πλήρω τη εξαιρετική ευκαιρία που μας παρέχει η ενιαία εσωτερική αγορά. Οι ψηφιακέ τεχνολογίες θα μας βοηθήσουν πολύ. Ήδη βλέπουμε ότι δημιουργούνται σημαντικές επιχειρήσει, μεγάλες, επιχειρήσει, που επωφελούνται τις ψηφιακέ πλατφόρμες για να πωλήσουν αγαθά και υπηρεσίες εκτός των συνόρων του. Αυτή την διαδικασία θέλω να τη φέρω και στι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Θα τελειώσω λέγοντας ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης της Νομοθεσίας, Εξέτασης Νομοθεσίας, θα κάνει το έργο της. Και θα πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Αυτή η Επιτροπή ελέγχει την ποιότητα της, των, της μελέτης αντικτύπου και να ελέγχει το κατά πόσον οι προτάσεις της Κομισιόν είναι φιλικές προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά προσεκτικά ε, ως και εγώ παλιάτρα μικρομεσαίος επιχειρηματίας ότι είναι σημαντικό να έχουν φωνή μικρομεσαίοι επιχειρηματίες κάθε φορά που ε, προτείνεται ένα καινούριο μαθητικό κείμενο. Και αυτή η Επιτροπή έχει να παίξει αυτό το ρόλο. Δεν θα είναι συμβουλευτική επιτροπή, είναι σημαντικό να διαθέτουμε την θετική της γνώμη κάθε φορά που η Κομισιόν υποβάλλει προτάσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, πρωτότυπο, που πιστεύω θα μας βοηθήσει να ακούσουμε τη φωνή και τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εμείς στην Κομισιόν και εσείς εδώ ως Ευρωβουλευτές. Αυτά ήθελα να σας πω εισαγωγικά. Είναι κρίσιμη σημασία θέμα ανοίγονται πολλές ευκαιρίες αλλά δημιουργούνται και πολλές προκλήσεις για το μέλλον. Θα, θα ακούσω με προσοχή και υπομονή την συζήτηση σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επιτροπέ να περάσουμε τώρα στις παρεμβάσεις. Δεν νομίζω ότι είναι εδώ η κυρία Φίρκμουνεν. Οπότε Α, βρίσκεται στην αίθουσα. Έχετε το λόγο για 1,5 λεπτό. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επιτροπή Μπρετών, που παρουσιάσατε τι απόψει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει αποτελούν πραγματικά τραχοκοκαλιά των ε, Τη οικονομία μα Είναι 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Είναι βασικό λοιπόν ο ρόλο του σε ό,τι αφορά την κοινοτομία, την αναγνωστικότητα τη Ευρώπη. Και χαίρομαι που η νέα Επιτροπή έχει πολλούς εξαιρετικούς ε, στόχους για τη βελτίωση της θέσης ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη για να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί ο ρόλος τους. Θα ήθελα εδώ να σημειώσω τρία σημεία. Καταρχάς, καλύτερη νομοθεσία, καλύτερη ρύθμιση που αποτελεί και το σημερινό μας ε, αντικείμενο. Μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα εφαρμόσετε το πώς θα εφαρμοστεί εξάντα και εξπόστ το κόστος υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ε, για να μειωθεί το κόστος στις επιχειρήσεις, αλλά να εξασφαλίσουμε και την τήρηση των περιβαλλοντικών και εργασιακών προτύπων. Ο αντιπρόεδρο Σεφκοβιτ είναι υπεύθυνο για τα θέματα αυτά, για τα θέματα καλή τη ρύθμισης. Θα μπορούσαμε να λάβουμε γραπτέ απαντήσει σε αυτή την ερώτηση, λοιπόν. Σε ό,τι αφορά το δικό σας χρωτοφυλάκιο, κύριε Μπρετόν, χαίρομαι καταρχάς που υπάρχει αυτός ο απεσταλμένος για τα μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το κοινοβούλιο το ζητούσε εδώ και καιρό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πού σκοπεύει να βάλει Πού σκοπεύει να τοποθετήσει την έδρα του απεσταλμένου αυτού και σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της στρατηγικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τις ε, καθυστερημένες πληρωμές. Γιατί αυτό το ακούμε επανειλημμένα και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από τους εμπλεκόμενους φορείς ότι όλο και πιο μεγάλα προβλήματα προκαλούνται και συχνά δεν ε, ακολουθείτε το χρονοδιάγραμμα. Ελπίζω να καταλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόβλημα αυτό και να το αντιμετωπίσει σε ό,τι αφορά τη νέα στρατηγική, γιατί η καλύτερη εφαρμογή της οδηγία για τις ε, καθυστερημένε πληρωμές θα πρέπει να εγγυηθεί. Ευχαριστώ. Η κυρία Τόγια, για ένα λεπτό. Να Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επιτροπή. Το πρόγραμμα που έχετε παρουσιάσει εδώ για μια στρατηγική για τις ΜΜΕ είναι πραγματικά ε, κάτι που μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος. Δεν βλέπουμε την ώρα να αρχίσουμε να εργαζόμαστε για τα θέματα αυτά. Τόσα χρόνια ζητάμε μια στρατηγική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρίς να έχουμε κάποιο ευτυχές αποτέλεσμα. Πρέπει να πω το πρώτο σημείο που βλέπουμε στην ε, ε, πρόταση είναι να κοιτάξουμε τους ορισμούς, τα κριτήρια για τους ορισμούς των μικρομεσαίων. Να θυμίσω, Επίτροπε, ότι το Κοινοβούλιο προσφάτως ε, πήρε θέση για το θέμα αυτό πριν αρχίσουν οι διαβουλεύσεις και επανεπιβεβαίωσε τα ισχύοντα κριτήρια, δηλαδή τον αριθμό των εργαζομένων και όλους τους εργαζόμενους που δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τις ε, ε, συνθήκε στις οποίες λειτουργούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν χώρες με μικροσκοπικές επιχειρήσεις, σε επίπεδο οικογενειακό δηλαδή. Για την συνολική στρατηγική πρέπει να και κάποια επιπλέον σημεία. Πρώτον, η δουλειά που κάνατε για τι αλυσίδε αξιών, παραγωγή αξιών είναι πολύ σημαντικέ. Πρέπει να συμπεριλάβουμε το μέγιστο δυνατό αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε, αυτές, σε αυτή τη στρατηγική για να ενισχύσουμε ε, τι επιλέξιμε εταιρείε και να μπορούν να ε, περάσουν στην επιτυχημένη μετάβαση. Μετά ο διάλογο μεταξύ ε, επιχειρήσεων εκπαίδευση και πανεπιστημίων ή ε, εκπαιδευτικών κέντρων, αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί καλά. Πρέπει λοιπόν στη στρατηγική να δούμε τα σχετικά σημεία, διότι νομοθετικά εργαλεία υπάρχουν, αλλά πρέπει να υπάρχει και το κατάλληλο περιεχόμενο για να υπάρχει κατάρτιση και. Ε, εκπαίδευση για να καλυφθούν οι αναγκέ δεξιοτήτων των επιχειρήσεων. Επίση, ψηφιακή εξέλιξη, καινοτομία, έρευνα. Πρέπει αυτό ε, να ε, το αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Θα πρέπει εδώ να κοιτάξετε, να πάρετε τα θετικά στοιχεία. Ό,τι είναι θετικό στην πρόταση νομοθεσία που κάνετε δεν πρέπει να ξεφύγει από το περιεχόμενο που θεωρούμε κέρια σημασία για τη στρατηγική. Ευχαριστούμε η κυρία Λαβάγιοβα Νταμπάλοβα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για όλα τα θετικά στοιχεία τα οποία αναφέρατε και είναι θετικό το ότι είμαστε τόσο φιλόδοξοι. Αναμένουμε λοιπόν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το όραμά της για τη νέα βιομηχανική αυτή πολιτική που θα δώσει νέα κίνητρα για ανάπτυξη, καινοτομία και θα έχει σωστά θεμέλια για να αντιμετωπίσει τις μερατικές προκλήσεις. Αυτό τι σημαίνει ότι ακόμα αναζητάμε τρόπους αντιμετώπισης του θέματος αυτού. Είχαμε ήδη συζητήσει τι πρέπει να κάνουμε για να υποστηρίξουμε τις δυναμικές εταιρείε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ στο Κοινοβούλιο κάποιοι συνάδελφοι πιστεύουν ότι πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες ανταγωνισμού. για να αποτρέψουμε το περαιτέρω, την περαιτέρω ανάπτυξη των μεγάλων επιχειρήσεων. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω το εξή. Καμία επιχείρηση δεν ήταν ε, μεγάλη από την αρχή. Όλες από κάπου ξεκίνησαν. Η Ευρώπη λοιπόν έχει ε, ένα τεράστιο πλανέκτημα, το μεγάλο δυναμικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και είναι σαφές τι εννοώ οι επιχειρήσει αυτέ έχουν δημιουργήσει πολλέ θέσει απασχόληση τα τελευταία χρόνια και αναπτύσσονται ταχύτατα. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσει ότι στην ευρωπαϊκή αγορά θα υπάρξουν μεγάλοι παίκτες, μεγάλες εταιρείες οι οποίες θα είναι επιτυχείς αλλά παράλληλα δεν θα καταπνίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες επίσης θα πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να έχουν επιτυχία και στην ευρωπαϊκή αγορά και στην διεθνή αγορά. Καλώ ορίζω λοιπόν τι προσπάθειέ σα για να επικεντρωθείτε στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Θα ήθελα όμω να ξέρω πώ θα εξασφαλίσετε ότι η αρχή του Think Small First, σκεφτόμαστε καταρχά τι μικρέ επιχειρήσει, θα επικρατήσει και θα διέπει όλε τι ε, πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε. Δύο σημειώσει προηγουμένω. Είμαστε στη φάση των αρχικών τοποθετήσεων από τι πολιτικέ ομάδε. Βάσει του ιστορικού κανονισμού δεν υπάρχει σε αυτή τη φάση διαδικασία γαλάζια κάρτα. Και ούτω ή άλλω έχουμε καθυστερήσει σε σχέση με το πρόγραμμα. Οπότε δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να υποσχεθώ ότι θα μπορέσουμε να έχουμε διαδικασία κάτι ε, πρώτα πρέπει όλοι να λάβουν τον απαραίτητο χρόνο αγορευσή του. Μετά ο λόγο στον κύριο Λεμπρετόν για 1,5 λεπτό. Merci, Monsieur le Président. Dans l'Union Européenne... Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι μικρομεσαίε επιχειρήσει αντιπροσωπεύουν πάνω από το 99% των επιχειρήσεων και το 2, τα 2 τρίτα των ε, θέσεων εργασία του ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρυνθεί η δράση του και η, ανταγωνιστικότητά του. Είναι ε, ε σημαντικές για την οικονομική ανάπτυξη. Η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές τεχνολογίες θα πρέπει να αποτελέσουν ευκαιρία για αυτές τις επιχειρήσεις και θα πρέπει να υποφεληθούν προκειμένου ε, να, να γιγαντωθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να βάλει τάξη στην οικονομική πολιτική τη. Θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβασή του σε χρηματοδότηση, ενθαρρύνοντα τι τράπεζε να δανείζουν χρήματα στι μικρομεσαίες επιχειρήσει και με εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επίση να δημιουργηθούν οι κατάλληλε συνθήκε υγιού ανταγωνισμού μέσα στην εσωτερική αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και επαναδιαπραγματευόμενοι τι συμφωνίε ελεύθερων ε, συναλλαγών που είναι υπέρ των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρήσεων. Θα πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες που πολύ συχνά τις αποθαρρύνουν από το να μεγαλώσουν. Επίσης, κύριε Επίτροπε, ε, δεν είμαι σίγουρος για την πραγματική επιθυμία της Κομισιόν να βελτιώσει την κατάσταση, γιατί, γιατί ο, διορισμός ενός ε, απεσταλμένου Κομισιόν επιχείρησης μου φαίνεται τέχνασμα. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό. Ο κύριος Μπόζελάγκερ Ντάμιον. Ευχαριστώ, Επίτροπε, που ήρθατε να συζητήσουμε το πολύ σημαντικό αυτό θέμα και χαίρομαι ιδιαίτερα που ε, και εσείς είσαστε επιχειρηματίας. Στα πολιτικά είναι λίγο διαφορετική η ατμόσφαιρα, αλλά είμαι πάντα μεγάλος υπέρμαχος της ανταγωνιστικότητας και των επιχειρήσεων. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζω την καλύτερη νομοθεσία για να μειωθούν οι αβεβαιότητες. Ξέρουμε ότι ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις, τις νεοφύσεις επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσουν αν υπάρχει νομική αβεβαιότητα. Αν λοιπόν αυτό μπορούμε να το επιλύσουμε θα είναι κέρδος. Ε, βλέπουμε επίσης μία τάση, λένε πολλοί συνάδελφοι, ότι θέλουμε να αποδυναμώσουμε την ανταγωνιστικότητα, λένε οι κυβερνήσει, για παράδειγμα, στην Γαλλία, στην Πολωνία. Αυτό είναι το αντίθετο τη ανταγωνιστικότητα. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον ανταγωνιστικό ε, χαρακτήρα χωρίς να αποδυναμώσουμε τη διάσταση του ανταγωνισμού. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Εκτό μικροφώνου δυστυχώς ο μιλητής. Εάν είναι έτσι η συζήτηση, ποιο είναι ο λόγος να κάθεται κανείς εδώ. Ευχαριστούμε. Εάν η διαμαρτυρία σας ε, έχει αυτό το περιεχόμενο, το σημειώνουμε. Αλλά Ξέρετε ότι η Προεδρία αποφασίζει για την διαδικασία της γαλάζιας κάρτας. Ούτως ή άλλως ο ιστορικός χρονισμός δεν προβλέπει το προς τον πρώτο γύρο των παρεμβάσεων των πολιτικών ομάδων να υπάρχει διαδικασία γαλάζιας κάρτας. Δεν θα αλλάξει η αποφασή μας σε σχέση με το θέμα αυτό. Και τώρα ο λόγος στον ε, συνάδελφο Γιουρίσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτό που χρειάζονται είναι λιγότερη γραφειοκρατία και ε, σταθερότητα, κράτος δικαίου και ανταγωνισμό. Η έγκριση μέτρων είναι στα χέρια των κρατών μελών για να εξασφαλίσουν ότι οι εταιρείε θα μπορέσουν να ε, δραστηριοποιηθούν και εκτός των συνόρων και στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς ε, τα εμπόδια. Ένα τέτοιο το εμπόδιο είναι η πρόσβαση στην χρηματοδότηση η οποία εκτός από το εκάστοτε κράτος μέλος είναι προβληματική. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν σαφέστεροι κανόνες για τις ευρωπαϊκές κεφαλαγορές και τέτοια είδους μέτρα θα έχουν ωφέλη και για τις μικρές επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές τους οποίους εξυπηρετούν στην τελική ανάλυση γιατί και οι δύο ομάδες τελικά από την ίδια πλευρά βρίσκονται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα για ένα λεπτό ο Αντιπρόεδρος Φάμπιο Καστάλτο. Ευχαριστώ πολύ. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, είναι η ραχοκοκαλιά της ε, οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, είναι αυτές που αποδεικνύουν ε, το ότι στην Ευρώπη έχουμε επιχειρηματική νοοτροπία. Χρειάζονται όμως και το κατάλληλο περιβάλλον για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η νομοθεσία να προσαρμοστεί στις ε, απαιτήσεις τους, ε, στις ανάγκες τους. Ο μηχανισμός Invest EU είναι πολύ σημαντικός, μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτό. Πολύ συχνά ε, είμαστε αποκομμένοι από τον κόσμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ακόμα και εμείς εδώ. Και θα πρέπει αυτό να το αποφύγουμε, προς συμφέρον όλων. Ευχαριστώ. Ο λόγος τον κύριο Κίσεκ. Για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμη πίτρο Πεμπρετών, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τη συνάδελφα την κυρία Βέρικονεν και να ζητήσω και από εσά και από τον ε, Επίτροπο Σεφκόβιτ ε, γραπτέ απαντήσει. Καταρχά, σε ό,τι αφορά το φίλτρο για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αναφέρεται λοιπόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ξεχωριστό τμήμα στην ε, αξιολόγησή σας. Πώ θα δημορφωθούν συγκεκριμένα τα μέτρα και πώς θα βελτιώσετε τα κριτήρια της αξιολόγησης ε, του μηχανισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε. Θα υπάρχει μελέτη αντικτύπου σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες συνέπειες ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ελέγχονται όλα αυτά πραγματικά. Και όλες αυτές οι ενώσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να δρουν ανεξάρτητα. Αυτό το πράσινο σύμφωνο επίσης τι ακριβώς συνεπάγεται. Είμαι βέβαιος ότι θα έχει σημαντικές ε, επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στο θέμα της ε, σωστής ε, ρύθμισης. Θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία της Σχετικής Επιτροπής για να είναι ένα εξάρτητο όργανο και ένα τρίτο θέμα σε ό,τι αφορά το εθνικό επίπεδο. Η... Γίνεται αυτό το gold plating και εδώ πέρα οι κανόνες είναι όλο και πιο αυστηροί. Και αυτό που είπατε στην αρχή για την, ε, τον εντεταλμένο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την αρχή one in, one out. Θα πρέπει να ξέρετε ότι σε όλα αυτά το ΕΛΚ είναι στο πλευρό σας. Ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Κονθάλεθ Κασάρες για ένα λεπτό. Κύριε Επιτροπέ, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει αποτελούν το 99% όλων των επιχειρήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και δημιουργούν 90 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Αποτελούν τη ραχοκοκαλιά τη οικονομία μας. Η Κομισιόν πράγματι έχει προτείνει ένα ειδικό πρόγραμμα για την εσωτερική αγορά ε, με προπολογισμό 1 δισεκατομμύριο ευρώ μόνον δεν αρκεί αυτό για να το καταστήσει στρατηγική σημασία. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζω ότι θα τη δω αυτή την προτεραιότητα στην βιομηχανική στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που θα συζητήσουμε του επόμενου μήνε. Με συγκεκριμένου στόχου. Μετρήσιμου στόχου. Και κυρίω φιλόδοξου στόχου προκειμένου να δώσουμε στον εαυτό μας τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε ε, την πρόκληση της ε, Πράσινης Συμφωνίας ε, και να κάνουμε πραγματικότητα την ψηφιακή μετάβαση. Χρειαζόμαστε επίσης ένα ισχυρό δημοσιονομικό χρηματοδοτικό πλαίσιο που θα δώσει οξυγόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπροστά από τις προκλήσεις των επόμενων ετών. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος στην κυρία Σράινα Μάρκερ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπη, συνάδελφοι. Την προηγούμενη Παρασκευή μίλησε ο Χάνς για ένα μια μια εταιρεία η οποία αναπτύχθηκε ήδη και ξεκίνησε από πολύ μικρή και έχει αναπτυχθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Έχουμε λοιπόν τέτοιε επιχειρήσει και χρειαζόμαστε τέτοιε επιχειρήσει με μεγάλο όραμα. Ο Χάντ λοιπόν συμφωνεί με αυτό το όραμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά δυστυχώ οι πολλαπλέ ε, νομοθεσίες και υποχρεώσεις ε, δυσκολεύουν τη ζωή του. Διοικητικά εμπόδια, δυσκολίες για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, όλα αυτά τα προβλήματα δυσκολεύουν τη ζωή τους. Αυτό δεν είναι ο σκοπό μα, γιατί οι εύκολε διασυνοριακέ συναλλαγέ είναι ένα από τα πιο βασικού στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν νομοθεσία θα πρέπει να ενισχύει του επιχειρηματίε και να απαντά στι συγκεκριμένε του ε, ανάγκε. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει αυτή την αρχή one in, one out, γιατί για κάθε μία νέα νομοθεσία και υποχρέωση θα πρέπει να αφαιρείται μία παλιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κυρία Σάινμακερ, έχετε γαλάζια κάρτα από τον κύριο Μάντελς. Τη δέχεστε? Ωραία. 30 δευτερόλεπτα εφόσον τη δέχεστε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, κυρία γιατί μας ε, δείχνει ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς ε, διαμορφώνονται τα εμπόδια και τα βάρη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μία ιδέα. Τι πιστεύετε για την ιδέα να εισαχθεί μία νόμιμη διαδικασία διατησίας με το Διεθνές Όλβιτ και το ECG να λαμβάνει αποφάσεις τα ταχείας αντιδράσεις προκειμένου στην τελική ανάλυση να ξέρουν τα κρατημέλη αν είναι ναι ή όχι. Ίσως και ο κύριος Μπρετών θα μπορούσε να μας απαντήσει στην ερώτηση αυτή. Κυρία Σράινε Μάχαρη, να απαντήσετε παρακαλώ. 30 δεύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Μάντλης, και σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά την πρότασή σας. Και δεν ξέρω πώς θα τέριαζαν και στο ευρωπαϊκό και ολλανδικό νομοθετικό πλαίσιο. Το γεγονός όμως ότι καθίσταται πιο εύκολη και λιγότερο χρονοβόρα ε, η διαδικασία αγωγής για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί μια εξαιρετική ιδέα και θα χαρώ να ακούσω και την απάντηση του κυρίου Μπρετών για το πώς ε, θα μπορούσαν να διαμορφωθούν λεπτομέρειες. Αλλά ναι, οποιοδήποτε τρόπο ε, θα μπορούσε να κάνει τη διαδικασία πιο συντόμα, θα με βρίσκει σύμφωνη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τώρα ο συνάδελφος Μπέκ για ένα λεπτό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, έχουν 56% της οικονομίας και ε, αποσχολούν ένα εκατομμύριο πολίτες είναι ε, σημαντική η πρόσβασή τους στην εσωτερική αγορά και οι πιστώσεις που λαμβάνουν από τις τράπεζες. Η πράσινη συμφωνία όμως ε, θα πρέπει να βρει και κονδύλια εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να υπάρξουν επενδυτές από τις μεγάλες τράπεζες διότι από το 2011 οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα ρευστότητας και δεν έχουν υποστηριχθεί. Εδώ ε, το ρευστό τρέχει σε, ε, όχι στην πραγματική οικονομία αλλά στην ε, αγορά των ακινήτων και σε άλλους προορισμούς. Μηδενικά επιτόκια και πολλοί περιορισμοί που ουσιαστικά διατηρούν ένα χρηματοοικονομικό σύστημα που δεν βοηθούν καθόλου την ευμερία των Ευρωπαίων πολιτών. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει το σύστημα αυτό. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο κύριος Χος για ένα λεπτό. Πρόεδρε, Επίτροπε, με προσοχή διάβασα την νέα στρατηγική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πραγματικά πολύ σωστέ οι προθέσεις, αλλά οι επιχειρηματίες είναι και εξαιρετικέφαλοι άνθρωποι. Έχουν το δικό τους όραμα και δεν μπορεί να τις ε, πείσει η αρχή, οι αρχές και μόνο. Και δεν έχουν οι επιχειρηματίε ε, ούτε χρόνο ούτε την όρεξη να το κάνουν αυτό. Και το λέω από δική μου προσωπική εμπειρία. Πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι με έξι α, διαφορετικές δράσεις, αλλά μειώνοντας τις α, Έτσι ο Τραμπ ε, υποστήριξε την αμερικανική οικονομία και έτσι διαγράφησαν οκτώ σχετικές ε, προδιαγραφές να κοιτάξουμε και τι γίνεται στο θέμα της ταξονομίας, γιατί εδώ υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να φροντίσετε λοιπόν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στη ε, χρηματοδότηση και να είναι γρήγορη η καταβολή των πληρωμών. Ευχαριστώ. You card από τον κύριο Σόκολ, τη δέχεστε? Yes. You have 30 seconds. 30 δευτερόλεπτα στον κύριο Σόκολ. Thank you very much. You mentioned many problems that SMEs are facing, but I think... Είπατε πολλά για τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά όλα αυτά έχουν πιο πολύ σχέση με την εθνική νομοθεσία, εθνικές διαδικασίες, εθνική φορολόγηση. Οπότε η ερώτηση είναι, Πιστεύετε ότι για να αποφύγουμε αυτά τα εμπόδια θα πρέπει να εναρμονίσουμε τα εθνικά συστήματα φορολόγησης με κοινού συντελεστέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί είναι ο μόνο τρόπο να έχουμε κοινού κανόνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αποφύγουμε και να άρουμε αυτά τα εθνικά εμπόδια. Χρειάζεται λοιπόν εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε κρατών φόρων Εν γέννη, πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι ευθύνη των κρατών μελών. Και δεν μιλώ μόνο για τους φόρους. Υπάρχουν και άλλοι κανόνες, όπως οι ε, κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, GDPR και ούτω καθεξής. Όλα αυτά επιβαρύνουν τα μέγιστα της μικρομεσαίας. Όμως η φορολογία είναι εθνική υπόθεση και δεν θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Ο κύριος Παπαδάκης για ένα λεπτό. Τα περί μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επικαλείστε στην πράξη αφορούν ορισμένες πιο δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που όντως σας ενδιαφέρουν στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι αυταπασχολούμενοι χωρίς ή με ένα δύο άτομα προσωπικό τις οποίες αντιμετωπίζετε ως διαρθρωτικό πρόβλημα. διαχρονικά έχει αποδειχθεί ότι όποια κονδύλια περισσεύουν από το φαγοπότι των μεγάλων ομίλων και δίνονται σε αυταπασχολούμενους, δεν είναι σε θέση να αντιστρέψουν το αδιέξοδο της αναδουλειάς της άγριας φορολόγησης των χρεών στην εφορία στις τράπεζες στα ασφαλιστικά ταμεία. δεν αναιρούν τον νόμο ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό πολύ περισσότερο που η απελευθέρωση υπηρεσιών ωραρίων και οι κανονισμοί της ευρωπαϊκής ένωσης ενισχύουν την τάση συγκέντρωσης των μεγάλων. η μεζούρα. Ε, φοροελαφρύνσεις της κυβέρνησης της νέας δημοκρατίας δεν ανατρέπουν την εικόνα στην ελλάδα ότι οι μικροί θα δίνουν μάχη επιβίωσης. μόνη διέξοδος υπάλληλοι αυταπασχολούμενων αυτοαπασχολούμενων μικροεπαγγελματιών όχι μόνο για την άμεση ανακούφισή τους από την αντιλαϊκή πολιτική ευρωπαϊκής ένωσης και κυβερνήσεων αλλά για την κοινωνική συμμαχία με την εργατική τάξη και τη μικρομεσαία αγροτιά προκειμένου να ανατραπούν τα μονοπόλια και εξουσία τους. Ο κύριος Πίπερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε την αίσθηση ότι οι μικρομεσαίοι ε, έχουν ε, μπει σε προτεραιότητα. Οι αρμόδιοι επίτροποι νιώθουν υποχρέωση απέναντι στις ΜΜΕ. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με χρηματοδότηση, ε, χρηματοδότηση, ε, ένωση κεφαλαίου. Ευχαριστούμε για τις καλές και πολλές προτάσεις για τις ΜΜΕ. Ευχαριστώ τον κύριο Μπρετό που είπε ότι η χρηματοδότηση και ε, δεν είναι τα πάντα, χρειάζονται και προϋποθέσεις πλαίσιο. Χρειάζεται εσωτερική αγορά χωρίς απομόνωση, μικρή περιορισμένη γραφειοκρατία, ψηφιακή οικονομία με δίκαιη πρόσβαση, σίγουρη πρόσβαση στα δεδομένα χρειάζονται πράσινες συμφωνίες και για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, πρόθεση της έρευνας. Ε, η πρόθεση των ΜΜΕ δεν περιορίζονται στη χρηματοδότηση. Θέλουμε μια κομισιόν λοιπόν η οποία θα βάζει στο επίκεντρο της ΜΜΕ. Ευχαριστούμε κυρία Μπρετών, αλλά όλα αυτά δεν αρκούν. Θέλουμε και η κυρία Φοντερ Λάιεν να ε, δεσμευτεί ως πρόεδρος της Επιτροπής. Αλλιώς ε, θα είμαστε κατακαιρματισμένοι. Τέλος, δεύτερος ε, ορισμός για τις ΜΜΕ που είναι η ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει όμως η δυνατότητα των μεγάλων κονσέρν. Και αυτό είναι ένα θέμα για την Κομισιόν. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πρέπει να συνδέονται με επιδοτήσεις. Θα πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις πλαίσιο για τις μικρομεσαίες. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, κυρία Κούταγιάρ. Grazie, Chair, Commissario. Żgur li taqbel miegħi li biex l-industrija tagħna tibqa' kompetittiva, li naddattaw Κύριε Επίτροπε, συμφωνείτε μαζί μου ότι πρέπει να προσαρμοστούμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Η στρατηγική για τις ΜΜΕ θα καθορίσει το ρόλο της Ένωσης σε παγκόσμια κλίμακα. Αν θέλουμε οι επιχειρήσεις μας να είναι ανταγωνιστικές, πρέπει να επιταχύνουμε την ψηφιακή μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Θέλουμε δεδομένα που θα αντικατοπτρίζουν τα σημερινά δεδομένα της τεχνολογίας. Οι ΜΜΕ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πόρους και χρηματοδότηση, σε δημόσιες συμβάσεις. Πρέπει να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες, να ενισχύσουμε το διάλογο στην αγορά. Πρέπει να βελτιώσουμε τα εργαλεία που διαθέτουν απέναντι σε αθέμητους κανόνες ε, στα κράτη-μέλη. Πρέπει να αυξήσουμε την ε, ενημέρωση σε σχέση με τα υφιστάμενα εργαλεία. Η ΜΜΕ είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δύο τρίτα των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται, δημιουργούνται από αυτές. Ε, τόσο σημαντικές είναι στις κοινότητές μας. Γι' αυτό πρέπει να υποστηριχθούν. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Mr. President. vous salue,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 Πολύ σκληρή έλεγχη σε κάποια κράτη-μέλη. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πολλέ φορέ υπάρχει και διαφθορά στον κρατικό μηχανισμό. Πολύ δύσκολα λοιπόν τα πράγματα. Και ακόμα και τα ευρωπαϊκά ταμεία δεν είναι προσπελάσιμα σε κάποια κράτη-μέλη για τι ΜΜΕ. Υπάρχουν ε, πραγματικά περίγραπτε διαδικασίε τόσο ε, που δεν μπορούν να εφαρμοστούν πρέπει να γίνει μια μελέτη η οποία θα καταδείξει τους λόγους για τους οποίους οι ΜΜΕ ε, πτωχεύουν και τι μπορούμε να κάνουμε για να τις βοηθήσουμε. Και, κύριε Επίτροπε, πρέπει να φροντίσουμε οι ευρωπαϊκοί κανόνες να βελτιωθούν και να μπορούν να εφαρμόζονται γρήγορα στα κράτη-μέλη. Και να, μην... Ε, ε,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 Και ε, γι' αυτό το λόγο αυτό το οποίο χρειάζεται είναι λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη καινοτομία, περισσότερη αποτελεσματικότητα. Αυτά χρειάζονται και λιγότερα λόγια και περισσότερες πράξεις. Το λόγο έχει κυρία Κέμπα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το είπαμε πολλές φορές άλλωστε αυτό. Αλλά οι πολλοί περιορισμοί, εσωτερικοί, εξωτερικοί, όπως γραφειοκρατία, οι βαριές διαδικασίες, ε, δυσκολεύουν τα πράγματα και είναι πολύ δύσκολο να διευθύνει κανείς μια μικρομεσαία επιχείρηση. Οι προϋποθέσεις και πλαίσιο είναι μακροπρόθεσμος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά στην πράξη τι συμβαίνει. Στην πράξη το, δημιουργήθηκε το πακέτο της κινητικότητας και έτσι η ανταγωνιστικότητα ε, υποβαθμίζεται. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, πτωχεύουν οι, οι επιχειρήσεις και έτσι αυξάνονται και τα, το κόστη μεταφοράς. Είναι οι ρυθμίσεις ε, προσανατολίζονται προς ανάγκες των κρατών μελών. Η απορρίθμιση, η απελευθέρωση του τομέα των υπηρεσιών, όπως λένε οι ειδικοί, ε, θα αυξήσει την ανάπτυξη κατά 1,7%. Και προς αυτή την κατεύθυνση του ανοίγματο των διαφόρων τομέων και της μείωσης ε, των υπερβολικών κανονισμών, ε, αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε που ήρθατε να μας μιλήσετε τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια μια που ξέρουμε όλοι ότι 90% περίπου των επιχειρήσεων της Ευρώπης είναι ΜΜΕ και έχουμε πάνω από 90 εκατομμύρια είναι οι εργαζόμενοι στις ΜΜΕ πάρα πολλά είπαμε και εγώ θέλω τώρα να επικεντρώσω την προσοχή μου σε δύο τινά Νομίζω δεν τα ανέφερε κανένας μέχρι τώρα και είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει επιπτώσεις στο αν θα μπορέσουν οι ΜΜΕ να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν όσον αφορά την τεχνολογία και όχι μόνο ε, την υποδομή της ψηφιακής τεχνολογίας. Έχουμε τώρα αυτόν τον ε, Ευρωπαϊκό Κώδικα, το 4G, οπτικές σύνες, 5G επίσης, ούτως ώστε να δοθεί αυτή η δυνατότητα και να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν την ψηφιακή αλλαγή η ΜΜΕ και να δούμε κατά πόσον υπάρχει υλοποίηση όπως πρέπει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και υπάρχει κάτι άλλο επίσης, ε, το οποίο δεν το προσέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτά τα δεδομένα χρειάζεται να υπάρχουν σχετικές δυνατότητες και για αυτό χρειάζεται κατάρτιση. Άρα χρειάζεται κάποιο πρόγραμμα δράσης φιλόδοξο, με στόχους ξεκάθαρους, μετρήσιμους, ούτω ώστε να δίνεται η όθηση στα κρατημέλη και να καλύψουν τα κρατημέλη το χαμένο έδαφος όσον αφορά την κατάρτιση και επίσης την εκπαίδευση στα ψηφιακά. Έχετε μία μπλε κάρτα, κύριε Λουκαστήγιο, λέει ο Πρόεδρος. Do Δέχεστε την μπλε κάρτα. I Εκτός μικροφώνου για την Έχετε μισό λεπτό, λέει ο Πρόεδρος. Μ' άρεσε αυτό το οποίο ότι πρέπει να βελτιωθούμε όσον την κατάρτιση και την εκμάθηση τη ψυχική τεχνολογία. Οπότε χρειάζονται στρατηγικέ Ένωση. Αυτό που θα σα ρωτήσω είναι ότι ε, πού βλέπετε τον ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ μπορεί να τα πάει καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το επίπεδο, με τα δεδομένα και την ανάλυση αυτών. Uh, uh, Θα σας τα πω στα ισπανικά. Υπάρχει μια σειρά από πρωτοβουλίε όσον αφορά τα δεδομένα ε, και ο Επίτροπος έχει τεράστια εμπειρία και είχαμε και την προηγούμενη ζήτηση που φάνηκε αυτό και ε, γι' αυτό νομίζω ότι θα μπορέσουμε να διχειριστούμε τα δεδομένα. Γι' αυτό και εγώ σα το λέω. Και εγώ γι' αυτό σα είπα δύο πρωτοβουλίε. Η μία έχει ξεκινήσει και είναι ο κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών για ανάπτυξη του το 5G και τη οπτική σύνα και επίση μια άλλη πρωτοβουλία, ένα άλλο σημείο. Κάτι να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κατάρτιση στα ψηφιακά, να γίνει πραγματικότητα αυτό, να μην ε, έχουμε εστέρηση. Επομένω αυτό θα πρέπει να δούμε. Αυτά που να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τηρούμε το χρόνο. Όπως με ενημερώνει οι συνεργάτες μου, είμαστε πίσω σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα 20 λεπτά. We are running of time about 20 minutes. Ε, επομένως, από εδώ και πέρα δεν θα επιτρέπω ε, μπλε για να κυλήσουμε ομαλά και να μην φτάσουμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριο Μπουσέιτ για ένα λεπτό.

Στην Πορτογαλία δημιουργήθηκε ένα σύστημα ενίσχυσης των ΜΜΕ. Μια εταιρεία μπορούσε να ε, συστήνεται μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ παλιότερα για να ιδρυθεί μια εταιρεία έπαιρνε μήνες. Η Βεβαίω, όταν προστατεύουμε τις επιχειρήσεις δεν σημαίνει ότι θα πάψουμε να προστατεύουμε τους ε, εργαζόμενους αλλά θα αξιοποιούμε την τεχνολογία για καινοτομίε, για διευκόλυνση και για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες. Πρέπει να έχουμε ευκολότερη στην εφαρμογή της νομοθεσία. Αυτό είναι σημαντικό για τις ΜΜΕ. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, μπορούν να φροντίσουν ότι θα συμμορφώνονται προς την ε, ε, νομοθεσία. Ε, έχουν τα διαθέσιμα κονδύλια που δεν τα έχουν οι ΜΜΕ και έτσι υπονομεύεται το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Και έτσι και υπολείπονται οι μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή μπλέκονται στη γραφειοκρατία και δεν μπορούν, οι κανόνες δεν είναι οι ίδιοι. Οι Είναι ο λόγος σας κύριε Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, υπάρχει ένα ισχυρό λόμπι το οποίο απεχθάνεται τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά αυτό έχει έμεσα και μεγάλες ε, ε, επιπτώσεις για τις ΜΜΕ. Ιδιαίτερα οι πράσινοι συνάδελφοι πιστεύουν ότι το κράτος μπορεί να λύνει καλύτερα τα προβλήματα με παρεμβατικό τρόπο από ό,τι η οικονομία. Δεν γίνεται αυτό όμως. Ξέρουμε εδώ και καιρό που βρίσκονται τα προβλήματα των ΜΜΕ. Ιδιαίτερα στον τομέα των φορολογικών επιβαρύνσεων και της γραφειοκρατίας. Η Πράσινη Συμφωνία, οι φόροι του άνθρακα τις επιβαρύνουν όλο και περισσότερο. Η γραφειοκρατία πλήττει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περισσότερο από ό,τι τις μεγάλες. Γι' αυτό είναι λάθος αυτό το σημείο της ημερησία διάταξης. Δεν έπρεπε να λέει better regulation, έπρεπε να λέει less regulation. Όχι καλύτερη, αλλά λιγότερη νομοθεσία και ρυθμίσεις. Αφήστε ε, την επιχείρηση να γίνει ξανά η κινητήρια δύναμη για την απασχόληση και την οικονομία μας. Επόμενος ομιλητής ο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε στην Ισπανία, όπως ανεφέρει η ΜΜΕ, είναι το 99% του επιχειρηματικού του. Παρ' όλα αυτά, έχουν πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά δυσανάλογη φορολογία, γραφειοκρατία και δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Επίσης, έχει ανέβει ο ελάχιστος ε, μισθός. Αυτά από τους κομμουνιστές και σοσιαλιστές που είναι στην εξουσία. 2.000 ευρώ περίπου για κάθε επιχειρηματοδότηση θέλουμε να έχουν αρκετά χρήματα οι εργαζόμενοι για να έχουν στέγη, να ζουν η οικογένειά τους, αλλά όχι εις βάρος των ΜΜΕ, όχι αυτές οι επιχειρήσεις να φορτώνονται το κοινωνικό ε, βάρος. Οπότε ε, θέλουμε κάτι να γίνει για το κοινό όφελος. Κάθε 10 επιχειρήσεις μία πεθαίνει κάθε 5 χρόνια. Οπότε θέλουμε να βελτιωθεί η νομοθεσία όλα αυτά καλοδεχούμενα, αλλά θα πρέπει να είμαστε τολμηροί. Να βελτιώσουμε την νομοθεσία σημαίνει κατάργηση νόμων και όχι με, με ρυθμό αργό. Ε, μαζικά να καταργούμε την γραφειοκρατία και να τους δώσουμε τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Δεν χρειάζονται νέες στρατηγικές. Χρειάζεται ελευθερία και ενυφαλιότητα. Η κυρία Καρβάλιο για 1,5 λεπτό. E κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και γι' αυτό δεν μπορεί να κατακλείζονται και να εξουθενώνονται από την εθνική και περιφερειακή γραφειοκρατία. Είναι σημαντικό να κάνουμε απλούστευση, απλοποίηση. Κάνοντας το αυτό, η Κομισιόν εστιάζει κυρίως στους κανονισμούς που αφορούν την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο ρύθμισης, ε, αλλά υπάρχουν και πολλά περισσότερα σημαντικά θεμελιώδη για τις επιχειρήσεις ολοκλήρωση μεταξύ άλλων της ε, ε, εσωτερικής αγοράς, ούτως ώστε εταιρείε από διάφορα κράτη-μέλη να μπορούν να έχουν ίσους ε, κανόνες ανταγωνισμού. Πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό πρέπει να είναι μια διαφανής διαδικασία με ενημέρωση και ευκολότερους κανόνες, ώστε να μπορούν να συγκρίνουν τους κανόνες που αφορούν τα διάφορα ταμεία. Π.χ. Ε, το Horizon, το 2020 ε, και η διευκόλυνση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πρόσβασή τους. Ε, λιγότερη γραφειοκρατία, καλύτερη και πιο ανοιχτή αγορά, αυξημένη πρόσβαση σε κονδύλια. Αυτά είναι οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για τις ΜΜΕ. Το λόγο έχει ο κύριος Ντάνιασον για ένα λεπτό. Tack för ordet. Eh, små och medelstora företag är naturligtvis Ευχαριστώ. Οι ΜΜΕ είναι πάρα πολύ σημαντικές για την οικονομία μας. Λιγότερη γραφειοκρατία, απλούστεροι κανόνες είναι σημαντικοί για την ανάπτυξή τους. Ένα όμως πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Αυτό που δεν είδε πρέπει να σημάνει περικοπή των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Όταν η Κομισιόν ε, μίλησε για το ενεντάουτα. Αυτό σημαίνει ότι οι ΜΜΕ θα επιβαρύνονται λιγότερο. Θα πρέπει όμως το εργασιακό περιβάλλον να παραμείνει στο επίπεδό του. Επουδενή δεν πρέπει η εργασιακή νομοθεσία να ε, γίνει χειρότερη την ε, πρωτοβουλία της προηγούμενης Κομισιόν που προέβλεπε ότι κάποιες επιχειρήσεις που είχαν ε, ένα λιγότερο... gospodine predsjedavajući mala i srednja poduzeća kralježnica su europske ekonomije pa njihova dobro. η τη ευρωπαϊκή οικονομία. Η ευημερία του έχει πολύ μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη και οι ευρωπαϊκέ κοινωνίε θέλουν να τους βλέπουν να ευημερούν. Χρειαζόμαστε λοιπόν θετικό επιχειρηματικό κλίμα, χαμηλού φόρου για να συμμετάσχουν σε κρατικέ προμήθειε, σε συμβάσει του δημοσίου, στην διαδικασία μάθησης και να μπορούν να συμπεριφέρονται όπω πρέπει στου υπαλλήλου τους. Οι πράσινε πολιτικές δεν πρέπει να θέσουν σε δυσμενέστερη μοίρα τι μικρομεσαίε. Η γραφειοκρατία και διάφοροι φόροι βαρύνουν υπέρμετρα τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Χρειάζεται λοιπόν μελέτη επιπτώσεων. Η Κομισιόν και τα κρατημέλη θα κάνουν ό,τι μπορούν για τι μικρομεσαίε. Υποστηρίζω λοιπόν όλε τι πρωτοβουλίε που στηρίζονται στην απορρίθμιση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει και κύριοι, είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει αυτό το πρόγραμμα στο οποίο να καλύψει και τις ΜΜΕ ως προτεραιότητα. Γνωρίζουμε ότι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία, όμως είναι ευάλωτες. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους φραγμούς. Η γραφειοκρατία είναι και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. έχουν πολλά να κάνουν με και δεν έχουν χρόνο να παρακολουθήσουν τις νομοθετικές εξελίξεις. Οπότε το νέο πνεύμα που διέπει το πρόγραμμα της Επιτροπής μία επιχείρηση για μία άλλη είναι κάτι που το θεωρώ θετικό. Να δοθεί δυνατότητα εξαγών της ΜΜΕ να έχουν απόδοση για το έργο τους και επίσης να καλυφθούν από την ψηφιακή οικονομία, να βοηθηθούν σε αυτό γιατί μόνες τους δεν το μπορούν. Επίσης, να υπάρχουν τέτοια προγράμματα που να βοηθήσουν, όπως και το έρασμος για τους νέους επιχειρηματίες. Κάνουν ό,τι μπορούν να οι για να δώσουν απασχόληση στους νέους. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να... Και ο κύριος Μπάλτ για ένα λεπτό. You have the... panie przewodniczący! komisarzu! średnie przedsiębiorstwa stoją wyzwaniami. Πρέπει να τους δώσουμε στήριξη με τη νέα στρατηγική, να βοηθήσουμε να επιτύχουν τους, τους οικονομικούς τους Αυτό θα ωφελήσει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από του σημαντικότερου στόχου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφορά την κλιματική αλλαγή. Πράγμα σημαντικότατο. Πρέπει να στηρίξουμε τις ΜΜΕ, ώστε να ενταχθούν στις νέε αυτέ πρωτοβουλίε, την Πράσινη Συμφωνία, ε, εκπαίδευση, κατάρτιση, την πράσινη οικονομία. Θα πρέπει να διαθέσουμε κονδύλια για τους ανέργους, για ανθρώπους που βρίσκονται σε μικρές ε, επιχειρήσεις. Σε κάποιες χώρες αυτό είναι πολύ, πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Πρέπει λοιπόν να δοθεί σωστή υποστήριξη στις ε, ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ δεν έχουν τα, τα απαραίτητα κονδύλια και την υποστήριξη για να αναπτυχθούν περισσότερο και να πετύχουν τις πρωτοβουλίες και τους στόχους. Ε, θα πρέπει να δούμε τις επιδοτήσεις που πηγαίνουν σε έργα για τις ΜΜΕ. Να ενθαρρύνουμε τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα δεδομένα αυτά Πρέπει να στηρίξουμε τις ΜΜΕ, ούτω ώστε να συμμετέχουν στο... Γόρμπον, για 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η αναβάθμιση των εργασιακών συνδικών στις ΜΜΕ είναι το πιο σημαντικό μα καθήκον, γιατί έχουμε γίνει ουραγοί στην παγκόσμια σκηνή. Άρα να έχουμε ένα πολιτικό πρόγραμμα αποφασιστικό να γίνουν ανταγωνιστικές η Ε. Η Κομισιόν είπε θα εφαρμόσει το one in one out για κάθε νέο νομοθέτημα θα, θα καταργείται ένα παλαιό και αυτό να ισχύσει τώρα αυτό το οποίο έχουμε τώρα είναι πολυνομία δεν αρκεί η πολυνομία για να είμαστε πρωτοπόροι στον κόσμο αυτό θέλουν οι σουηδικές επιχειρήσεις. Να μην αρκείστε στη θέση που έχουμε σήμερα. Θα πρέπει να βάλετε τον πύχη πιο ψηλά. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν ότι θα προσπαθήσετε κατά 30% μειώσετε την γραφειοκρατία. Αυτό θέλουν οι κεντρώοι στην ε, Σουηδία για τις... λεπτό tisztelt η βάση για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις που όμως αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλες δυσκολίες, γραφειοκρατία, πολλές διατάξεις. Είναι απαραίτητο λοιπόν να κάνουμε στην εσωτερική αγορά ό,τι είναι δυνατόν, ούτως ώστε οι ΜΜΕ να πρέπει να πληρούν τις ε, λογικές νομικές διατάξεις και να απελευθερώνονται, να απαλλάσσονται από τις άλλες. Ε, θα πρέπει να δούμε τα σοβαρά προβλήματα ανταγωνισμού που έχουν η ε, Σιγκαπούρη επικεφαλής των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας έχουν προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό το τομέα ε, εμείς έχουμε πάρα πολλές διατάξεις. Επίσης, η ευρωπαϊκή οικονομία θα πρέπει να δει ε, το θέμα της ψηφιοποίησης, ψηφιακής οικονομίας. Κύριε Επίτροπε, πρέπει να πάρουμε μέτρα, να προβούμε σε βήματα για να λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Η Κομισιόν πρέπει να κάνει τις νομοθετικές προτάσεις της προς αυτή την κατεύθυνση, να δει δηλαδή τι επιπτώσεις θα έχουν οι νομοθετικές προτάσεις της ΜΜΕ και την ανταγωνιστικότητά τους. Παρακαλώ λοιπόν να λάβετε τα σχετικά μέτρα και να βοηθήσετε ε, εισάγοντας ένα φίλτρο υπέρ των ΜΜΕ. Αυτό θα είναι προς το συμφέρον τους. Συνάδελφοι, επίτροπε, είναι θετικό κάνουμε αυτή την συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οικονομία. δέκα χρόνια είχα τη δική μου εταιρεία, οπότε κάτι ξέρω από το θέμα μας. Έχω δύο ερωτήσεις να σας υποβάλω. Πολλές ΜΜΕ ε, δυστυχώς διαπιστώνουν ότι έχουν τόσες υποχρεώσεις που προέρχονται από τις τελευταίες φάσεις των τριμερών διαλόγων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεν το έχει αντιμετωπίσει η Επιτροπή. Τι θα κάνει για να βοηθήσει, πώς αυτό θα επιληθεί. Δεύτερον, τι θα κάνετε για να βοηθήσετε την πρόσβαση των πράσινων ΜΜΕ στην παγκόσμια αγορά με συμφωνίες εμπορικές Προσφέρονται πολλές ευκαιρίες από την ενιαία αγορά, όμως επειδή υπάρχει το πρόβλημα της αλλαγής του κλίματος, θα πρέπει να δούμε πώς οι ΜΜΕ, οι ευρωπαϊκές, θα κάνουν τη διαφορά στην παγκόσμια σκηνή. Για Περέιρα για ένα λεπτό senhora presidente as pequenas e médias empresas surgem a miúdo no discurso da comissão europeia quase sempre com fins justificativos de legislação seja de Η Κομισιόν μόνο φορμές βρίσκει για περισσότερους κανόνες. Αυτά δεν γίνονται για τις μικρομεσαίες. Οι περισσότερες υπόκεινται αυτό που χρειάζονται είναι βοήθεια. Δυστυχώ είναι οι πρώτε που υποφέρουν κάθε φορά που η οικονομία δεν πηγαίνει καλά. Και κάθε φορά που προβλέπει περαιτέρω απορρίθμιση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ή όταν αντιμετωπίζουν τι μεγάλε επιχειρήσει και τι τράπεζε. Είναι πολύ σημαντικό να τι βοηθήσουμε. Έχει στρατηγική σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία και πρέπει να τις προστατεύσουμε κατά των μεγάλων τραπεζών. και να αποφύγουμε αυτά που λέει. Αυτό ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των εγγεγραμμένων ομιλητών και από ό,τι με ενημερώνουν είμαστε 25 λεπτά πίσω από το χρονοδιάγραμμα. Έχω δεχθεί για τη διαδικασία του Catch the Eye ε, αρκετά αιτήματα. Μπορώ να κάνω δεκτά μόνο δύο από κάθε πολιτική ομάδα, δεν μπορώ περισσότερα. Το λόγο έχει ο κύριος Κάνεφ για ένα λεπτό.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 να υπάρξει ενιαία διαδικασία υπαγωγής στον ΦΠΑ. Ας πούμε ποιος έχει πάνω από 100.000 ε, τζίρων υποχρεωτικά να εγγράφεται στην εφορία για ε, ΦΠΑ στην ε, Βουλγαρία. Έχουμε αυτό το όριο, αυτό το ποσό. βέβαια το αντίστοιχο για μας είναι 25.000 ευρώ και δεν είναι δίκαιο για μας. Επίσης, έχω και άλλη μια πρόταση να σας ε, κάνω. Να έχουμε ε, κάποιο ελάχιστο φορολογικό όριο, ελάχιστο φορολογικό συντελεστή μάλλον. Έτσι, θα έχουμε πιο δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των ΜΜΕ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κύριος Χάσελ, για ένα λεπτό. Η πράσινη συμφωνία και η μετάβαση προς πιο πράσινη ψηφιοποιημένη οικονομία θα είναι μεγάλο βάρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί από τη μια είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, αλλά από την άλλη είναι πολύ ευάλωτες. Απέναντι σε οποιαδήποτε κρίση μπορεί να υπάρξει στο μέλλον. Τι χρειάζονται λοιπόν. Χρειάζονται το κράτος δικαίου να εφαρμόζεται, να ισχύει και πρέπει να προστατεύονται στο, από τον ανταγωνισμό. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Κομισιόν. Χρειάζονται οι ΜΜΕ επίσης ένα σταθερό νομικό περιβάλλον, γιατί δεν, μπορούν, δεν έχουν τη δυνατότητα να απορροφούν όλες τις αλλαγές που προκύπτουν. Γι' αυτό είναι καλό που η Κομισιόν ε, εισήγαγε αυτό τον κανόνα του One In, One Out. Το γραφειοκρατικό φορτίο είναι το μεγαλύτερο απ' όλα για τις ΜΜΕ. Χρειάζονται ακόμη περισσότερη χρηματοδότηση για να μπορούν να... Thanks very much, uh, Mr. President. Um, I don't accept for a minute that good regulation... Δεν δέχομαι ότι όλα αυτά βοηθούν τις μικρομεσαίες. Θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημα. Κάποιοι λήθοι γραφειοκράτες, αυτό είναι το πρόβλημα για τις μικρομεσαίες. Αυτά είναι που βλάπτουν τις μικρομεσαίες. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Δεν βάζουμε κανόνε στι τράπεζες που επιβαρύνουν τις μικρομεσαίες, που κάνουν δύσκολη τη ζωή των μικρομεσαίων. Έχουμε το κόστος της ενέργεια. Πολλές φορές ε, δεν υπάρχει αρκετή νομοθεσία από τα κρατημέλη. Στην Ιρλανδία η νομοθεσία σκοτώνει τις μικρομεσαίες. Γιατί, Γιατί δεν υπάρχει ρύθμιση ας πούμε, των ενοικίων, όπως φαντάζομαι και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η έλλειψη λοιπόν καλών κανόνων αυτή σκοτώνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εννοείται ότι φταίει επίση η στήριξη από τις κυβερνήσεις. Χρειαζόμαστε άμεσε επενδύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Νίμπλερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Οι εταιρείε μας, οι επιχειρήσεις μας ε, υποφέρουν από την υπερβάλλουσα γραφειοκρατία. Συγκεκριμένο παράδειγμα που δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα για πολλές γερμανικές, βαβαρικές επιχειρήσεις. Η, το πιστοποιητικό Α1, δηλαδή το πιστοποιητικό που πρέπει να έχει κανείς όταν παρέχει υπηρεσία σε άλλη χώρα μέλος. Θα πρέπει δηλαδή να αποδεικνύει ότι έχει κοινωνική ασφάλιση. Και όταν ε, πρέπει κανείς να συναρμολογήσει αλλού ένα μηχάνημα θα πρέπει να έχει το πιστοποιητικό. Γιατί αν δεν μπορεί ε, θα πρέπει να πληρώσει μεγάλο πρόστιμο. Αυτό δημιουργεί προβλήματα χωρίς τέλος. Κύριε Επίτροπε, υπολογίζω σε εσάς ε, ξέρετε ε, την ψηφιακή ε, τεχνολογία θα πρέπει να έχουμε ένα συνολικό σύστημα για το πιστοποιητικό ε, Α1 το οποίο θα ισχύει για όλη την Ευρώπη και θα μπορεί να παρακολουθείτε και ηλεκτρονικά. Θα ήταν πάρα πολύ καλό να μπορούσε να ερμονιστεί το... Ευχαριστώ το λόγο κυρία Ντέιλι για ένα λεπτό. Thank you, um, I'm very glad... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που μιλάμε για τις μικρομεσαίες. Απασχολούν περισσότερους ανθρώπους, πληρώνουν περισσότερους φόρους, σίγουρα στην Ιρλανδία και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται είναι απίστευτα εχθρικό, ιδιαίτερα αν σκεφτούμε τις άμεσες ξένες επενδύσεις και το τι χάρες κάνουμε στις πολυεθνικές και πόσο υποστηρίζουμε τους αγρότες. Στην Ιρλανδία οι μικρομεσαίες φέρουν το μεγάλο βάρος, το φορολογικό, το οποίο δεν φέρουν οι πολυεθνικές. Και βεβαίω είναι οι πρώτε που πλήττονται όταν ε, έχουμε καιρού λιτότητα. Είναι ντροπή νομίζω. Να μην φορολογούμε την Apple για τα δισεκατομμύρια που χρωστάει και να ρίχνουμε το βάρος στις μικρομεσαίες. Λοιπόν, συμφωνώ με αυτά που είπαν και οι προλαλήσαντε, δεν μπορούμε να μην θεσπίζουμε καλού κανόνε. Δεν μπορούμε να υπερασπιζόμαστε του γραφειοκράτε. Χρειαζόμαστε καλού κανόνε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για την απασχόληση, για τι μικρομεσαίε, για την προστασία του περιβάλλοντο και τι μικρομεσαίε. Σα ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Catch the Eye. Λυπάμαι που δεν μπορώ να δώσω το λόγο σε όσε και όσου επιπλέον ζήτησαν. Σε αυτή τη φάση είμαστε 25 λεπτά πίσω από το χρονοδιάγραμμα. Εξ ονόματο τη Επιτροπή, το λόγο έχει ο κύριο Μπρετόν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευχαριστώ πολύ για μια πλούσια συζήτηση που δείχνει ότι συμμερίζεστε την προβληματική η οποία αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι η ραχοκοκαλιά, όπω είπαν πολλοί, τη οικονομική μα δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όλοι συμφωνούν, πιστεύω, με τα εξή. Έχουμε καθυστερήσει πληρωμών. Υπάρχει ανάγκη ένταξη των μικρομεσαίων στην αλυσίδα αξία. Χρειάζονται οικονομική στήριξη. Έχουμε υπερβολική γραφειοκρατία. Πρόβλημα πρόσβαση στις ε, πιστώσεις, πρόβλημα ψηφιοποίησης. Συμφωνούμε όλοι με αυτά, πιστεύω. Ανησυχούμε με τον ίδιο τρόπο. Από την πλευρά μου θα προσπαθήσω να απαντήσω εντάχει επί όλων αυτών των θεμάτων που θίξατε. Πολλά από αυτά απαντώνται με το σχέδιο που προτείνουμε για την βιομηχανική πολιτική, αν και είναι αλήθεια ότι οι αλυσίδες αξίας τις οποίες ε, στηρίζεται μια σωστή βιομηχανική πολιτική πρέπει να ενσωματώνει εννοείται όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά τα κόστη. Μίλησαμε με τον Επίτροπο Σεύκοβιτς, τον συναδελφό μου. Οι κατευθυντήριες γραμμές ήδη σας δίνουν μια ιδέα της μεθοδολογίας που ακολουθούμε, όμως η ανακοίνωση περί καλής νομοθεσίας διαλαμβάνεται των λύσεων που προτείνουμε. Να Επιμείνω όμως στο εξή. Μιλούμε για τη σώρευση στοιχείων κόστος που πιέζει τις μικρομεσαίες. Πολλές επιβαρύνσεις προκύπτουν από εθνική νομοθεσία. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Όσον αφορά τον υπεύθυνο για τις μικρομεσαίες δεν έχουμε ακόμη καταλήξει ποιος ή ποια θα είναι. Αλλά θα σκεφτούμε αυτή τη λύση, ήδη σκεφτόμαστε από σήμερα. Το βέβαιο είναι ότι το πρόσωπο αυτό θα έχει δική του ομάδα, θα αναφέρεται σε μένα και θα ασχολείται 100% με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πράξη. Για να αφουγκραστούμε το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να κάνουμε κάτι επιτέλους για αυτές. Μόλις επιλεγεί το κατάλληλο πρόσωπο, αν δεν έχετε αντίρρηση, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, θα σα παρουσιάσω την αρχιτεκτονική αυτή τη νέα λειτουργία. Η καθυστέρηση των πληρωμών. Ουσιαστικό το θέμα, το δείξατε πολλοί από εσά. Πρόκειται για θέμα το οποίο παρακολουθώ στενά. Πρέπει να κατανοήσει κανεί πώ λειτουργούν οι αλυσίδε αξία για να καταλάβει γιατί έχουμε καθυστερήσει πληρωμών. πρέπει οι μικρομεσαίε να αποκτήσουν μεγαλύτερη οικονομική ανεξαρτησία. Το παρακολουθούμε, όπω είπα, πολύ στενά. Για να μην σα καθυστερώ, ένα άλλο θέμα το οποίο θίξατε. Διτησία. Είναι πολύ ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν είναι ένα θεσμό που μπορεί να λειτουργήσει, αλλά σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο το γνωρίζω και εγώ προσωπικώ. Πολλέ ε, μικρομεσαίε δεν καταφεύγουν στην δικαιοσύνη γιατί ξέρουν ότι θα πάρει πολύ χρόνο, είναι δαπανηρό. Οπότε η λύση της διαιτησίας είναι πιθανότερα μια πολύ ενδιαφέρουσα λύση την οποία θα εξετάσω. Το περίφημο gold plating. Όπως προείπα, η υπερβολική νομοθεσία επιβαρύνει τις μικρομεσαίες. Δεν υπάρχει καμία εμφιβολία. Πρέπει να δούμε πού έχουμε υπερβολικούς κανόνες, περιτούς κανόνες, κάναμε κάποια πράγματα, θα κάνουμε όμω περισσότερα και θα επανέλθω να σα ενημερώσω. Σίγουρα χρειάζονται να γίνουν περισσότερα και πιο γρήγορα. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση υψηλή σημασία. Είμαστε στην ψηφιακή μετάβαση. Είναι θέμα το οποίο θα ξανασυζητήσουμε. Έχουμε πει στα περιφερειακά ταμεία, πολύ σημαντικό θέμα και αυτό, το κόσμο, για παράδειγμα, με 30 δισεκατομμύρια ήδη ευνόησε 300.000 επιχειρήσεις το InvestEU και αυτό βελτιώνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Επίσης κινητοποίησαμε επιπλέον 11,2 δισεκατομμύρια μέσω του InvestEU. Δεν είναι αρκετό, αλλά σίγουρα έχουμε εργαλεία τα οποία είναι σημαντικά και τα οποία έχουν ακριβώς αυτόν τον ρόλο, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και γιατί άλλο το φίλτρο των μικρομεσαίων. Κάνουμε ανάλυση επιπτώσεων. Κάποια στιγμή θα πάρουμε και τη σχετική απόφαση. Τι είναι μικρομεσαία. Αλλά ε, σας θυμίζω ότι θα κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει. Το φίλτρο αυτό είναι αποκεντρωμένο και θα εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας για να ξεκριβώνουμε, για να βεβαιωνόμαστε κάθε φορά ότι η νομοθεσία λαμβάνει υπόψη τη τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Και σε αυτό θα συμμετάσχουν όλε οι υπηρεσίε τη Κομισιόν, ε, σε συνεργασία βεβαίω με τον ε, ε, μελλοντικό υπεύθυνο για τι μικρομεσαίε. Πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις. Πολύ σημαντικό, μιλάμε για το 90% των επιχειρήσεων μιας χώρας, πρέπει αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν καλύτερη πρόσβαση, προνομιούχου θα έλεγα, πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις. Και περιλαμβάνω εδώ και τις startup, τις νεοφύης επιχειρήσεις, που έχουν την ίδια ανάγκη. Και όσον αφορά το νομικό πλαίσιο των ε, δημοσίων προμηθειών, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο και πώς. Τέλος, είναι κάτι το οποίο έθιξα και στην εισαγωγή μου, η εσωτερική αγορά οι μικρομεσαίες μας πρέπει να εποφελούνται από αυτήν την εσωτερική αγορά. Αυτό είναι το κλειδί. Δυστυχώς σήμερα διαπιστώνουμε ότι μία ή δύο πλατφόρμες που δεν είναι ευρωπαϊκές μάλιστα αυτές είναι οι κλειδούχοι που ελέγχουν την πρόσβαση στην αγορά δυστυχώς και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας οθήσει να κάνουμε κάτι Θέλω να σας βεβαιώσω επίσης ότι η ψηφιακή μετάβαση θα δώσει στις μικρομεσαίες μας προσβέσει σε αγορές εκτός των εθνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Ακούσαμε ευρωπαϊκές, ε, ενδιαφέρουσες ιδέες σχετικά με, την, με τις δυνατότητες αυτές πρόσβεσης. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα βεβαίω, ειδικά όσον αφορά την εισπράξη των φόρων, αλλά θα λυθεί σε εθνικό νομίζω επίπεδο. Τέλο, ένα θέμα το οποίο αποδείχθηκε αυτό σήμερα, το one in, one out. Η αρχή δεν μπορεί να εφαρμοστεί με τρόπο μηχανιστικό. Παρακολουθούμε βεβαίω τι γίνεται στην αγορά. Δεν πρόκειται για ένα μηχανισμό απορρίθμισης, ούτε θα μειώσουμε, θα αποδυναμώσουμε την προστασία των εργαζομένων. Αλλά θα δούμε πού πηγαίνουμε, τι άλλαξε. Ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος εξελίσσεται ταχύτατα και δει υπό την πίεση της ψηφιακής εποχής. Εμείς θέλουμε η Ευρώπη να πάει μπροστά με βάση το Πράσινο Σύμφωνο και όλα αυτά, όπως είπα, εξελίσσονται. Εξελίσσεται και η γεωπολιτική, ο συσχετισμός δυνάμεων με τις άλλες υπήρους. Αυτά λοιπόν πρέπει να δούμε, πρέπει να εξεγνωριστούμε. Κυρίε και κύριοι, αυτά είχα να πω απόψε. Διαπιστώνω το έντονο ενδιαφέρον σας. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. όταν έρθει η ώρα να παρουσιάσουμε την στρατηγική μας για την βιομηχανία που θα μιλήσουμε βέβαια και για τις μικρομεσαίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Η συζήτηση έληξε. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με τον κανονισμό ενωσιακών έργων κοινού ενδιαφέροντος και την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας και πιο συγκεκριμένα προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 του κανονισμού Ενωσιακός Κατάλογος Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος. Εισαγωγικά σας λέω ότι επειδή έχουμε καθυστερήσει 30 λεπτά σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα δεν θα δεχθώ μπλε κάρτες στη συζήτηση αυτή παρά μόνο περιορισμένα τη διαδικασία του Catch the Eye. Το λόγο έχει για πέντε λεπτά ο κύριος Μπουσόη, συντάκτης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Ο κανονισμός για τις κατευθυντήριες γραμμές ε, εν προκειμένου θέτει κανόνες διαλειτουργικότητας, λειτουργία θέτει προτεραιότητες που πρέπει να εφαρμοστούν ούτω ώστε να αντιμετωπιστούν οι στόχοι στην ενέργεια και το κλίμα στην Ένωση, εντοπίζει δε έργα κοινού ενδιαφέροντος για να γίνουν όλα αυτά. Ε, προβλέπονται και διάδρομοι προτεραιότητας και δίδονται κατευθυντήριες γραμμές για την επιλογή των έργων κοινού ενδιαφέροντος. Ε, τα σχέδια κοινού ενδιαφέροντος, PCIs, ε, εγκρίθηκαν το 2013, τώρα είμαστε στον τέταρτο κατάλογο που στις 31 Οκτωβρίου του 19 ε, ολοκληρώθηκε με 151 τέτοια PCI έργα. Όπως ε, φάνηκε και από την ε, πρώτη ανάγνωση στις 17 Απριλίου για την πρόταση κανονισμού για την διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη, οι συνομοθέτες προσωρινά συμφώνησαν ότι η Κομισιόν θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και πολιτική συνοχή της, ε, του κανονισμού. Για την αξιολόγηση θυμίζω ότι η Κομισιόν έπρεπε να δει μεταξύ άλλων τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους μέχρι το 2030, ε, ε, την μείωση του, της χρήσης του άνθρακα και η ενεργειακή μετάβαση. Ο κανονισμός εγκρίθηκε πριν από την έγκριση της Συμφωνίας των Παρισίων. Ε, που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για το πέρασμα στην οικονομία χωρίς τη χρήση άνθρακα. Ε, τα συστήματα ε, μείωσης του άνθρακα χρειάζονται ούτως ώστε να επιτύχει τα φιλόδοξα σχέδιά της η Ευρώπη και να παίξει παγκόσμιο ρόλο, ενώ παράλληλα θα διασφαλίσει ήπια μετάβαση και φροντίζοντας για την ενεργειακή απόδοση ε, και ενεργειακή επάρκεια. Η ε, βιωσιμότητα, η ανάπτυξη ε, αλλά και η ανταγωνιστικότητα είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες εδώ. Και η Κομισιόν θα πρέπει μια υψηλής απόδοσης υποδομή για τις μελλοντικές της ενεργειακές ανάγκες. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας θα πρέπει να ακολουθούν την ανάπτυξη του συστήματος ενέργειας και να διατηρούν τη συνοχή και τη συνέπεια με άλλες ε, πολιτικές της Ένωσης ε, στο πλαίσιο της μείωσης του άνθρακα. Η ε, χρήση προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά για την επίτευξη των στόχων. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για την ενεργειακή απόδοση, να αυξήσουμε τη χρήση καθαρών τεχνολογιών, να αυξήσουμε την διασυνδεσιμότητα και να ε, διευρύνουμε τη χρήση του στην εσωτερική αγορά. Ήδη ε, δέκα κατευθυντήριες γραμμές ε, βάσει του Συμφωνίας των Παρισίων έπρεπε να αναθεωρηθούν. Υπάρχει ανακοίνωση ότι η αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τα ε, TEN-T ε, θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οι ε, υποδομές ε, θα πρέπει να παρακολουθούνται για 40-50 χρόνια και περισσότερο καμιά φορά. Οι υποδομές αυτές στο μέλλον θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά βιοαερίου, υδρογόνου και όχι στο μακρινό, πολύ μακρινό μέλλον και στη φάση της μετάβασης ε, η αγωγή, οι διασυνδέσεις παίζουν σημαντικό ρόλο για να διασφαλίσουν τον ενεργειακό εφοδιασμό και τη βιωσιμότητα ε, του συστήματός μας. Χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη, ρεαλιστική προσέγγιση, ε, ούτως ώστε να είμαστε ουδέτεροι ως προς τη χρήση άνθρακα. Και ακόμα έχουμε ε, πολλές ε, περιοχές που ακόμα στηρίζονται ε, στον άνθρακα και πρέπει να υποστηριχθούν. Η κυρία Τουσέν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Ο πλανήτης πεθαίνει. Οι εμπειρογνώμονες μας λένε τέρμα στα ορυκτά καύσιμα και όμως οι δηλώσεις μας δεν συνάδουν με τις πράξεις μας. Ένα τρίτο των έργων που προτείνεται αφορούν ορυκτά καύσιμα και σας ζητούμε σήμερα να το ξαναδείτε. Πρόκειται για επιστημονικό και οικονομικό λάθος, κυρίως για πολιτικό λάθος. Πρόκειται για επιστημονικό λάθος, διότι γνωρίζουμε εδώ και καιρό ότι 94% των ορυκτών πόρων που χρησιμοποιούμε σήμερα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Είναι οικονομικό επίση λάθο, γιατί επενδύουμε σε πανάκριβα έργα τα οποία υπονομεύουν την δυνατότητά μα να επενδύσουμε εκεί που πρέπει, εκεί που υπάρχουν πραγματικέ ανάγκε. Κάτι δεν πάει καλά, κυρία Επίτροπε. 29 δισεκατομμύρια που πρέπει να πάνε στο κλίμα. Και είναι και πολιτικό το σφάλμα. Διότι ο κατάλογος που προτείνεται είναι επικίνδυνη για τον πλανήτη και εν τέλει για τους πληθυσμούς μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να αναθεωρήσουμε τον κατάλογο αυτό το συντομότερο δυνατόν, διότι η Ευρώπη δεν, ε, πρέπει, δεν μπορεί να συνεχίσει να επενδύει στα ορυκτά καύσιμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα νέο κατάλογο εκτό πλέον ορυκτών καυσίμων. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ιστορία μα δείχνει το δρόμο. Μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χτίσαμε την Ευρώπη πάνω στον Χάλιβα και τον Άνθρακα. Σήμερα μιλάμε για πράσινε μορφέ ενέργεια. Έτσι θα επανοικοδομήσουμε την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη δικαιοσύνη για τους πληθυσμούς μας. Κύριε Επιτροπέ, θα έπρεπε να έχετε απορρίψει αυτόν τον κατάλογο, αυτήν την πρόταση που κληρονομήσετε από τον προκατοχό σα. Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλοί έχετε τι αμφιβολίε σα, το ξέρω. Ήρθε η ώρα να διατυπώσουμε τι αμφιβολίε μα, τι αντιρρήσει μα. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε μοντέλο για να προστατεύσουμε το μέλλον. Ήρθε η ώρα να δείξουμε τον δρόμο την Τετάρτη λοιπόν να ψηφίσουμε για το Πράσινο Σύμφωνο και ας πούμε όχι στον καταλόγο αυτόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής έχει η Επίτροπος κυρία Σίμψον. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πριν από δύο μήνες παρουσίασα τις απόψεις μου ενώπιον της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Είχα πει ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό και το λέω και σήμερα. Στο ψήφισμα για το Πράσινο Σύμφωνο του Ιανουαρίου, το Κοινοβούλιο υπογράμμισε την ανάγκη νέων έξυπνων καθαρών υποδομών ενέργειας για να υλοποιήσουμε λοιπόν την Πράσινη Συμφωνία. Συμμερίζομαι το με αυτό. Πρέπει όμως τώρα να το κάνουμε πραγματικότητα. Ήδη από το 2013 είχαμε ξεκινήσει αυτές τις προσπάθειες και νομίζω ότι όλοι ευθυγραμμιζόμαστε με το πνεύμα αυτό. Αν θέλουμε η Ευρώπη το 2050 να είναι η πρώτη ενεργειακά ουδέτερη ε, ήπειρο, έχουμε να κάνουμε πολλά. Η Κομισιόν θα προβεί σε μια αξιολόγηση της κατάστασης των δύο ευρωπαϊκών δικτύων φέτο. Θα επιταχύνουμε μάλιστα αυτή την ε, αξιολόγηση και θα αναθεωρήσουμε και τον σχετικό κανονισμό ε, για να υποβάλουμε πρόταση τον Δεκέμβριο του 2020. Ο κυρίως στόχος είναι να δημορφώσουμε ένα μελλοντικό πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει να χρηματοδοτήσουμε τις υποδομές που χρειαζόμαστε για να υλοποιήσουμε το πράσινο σύμφωνο. Χρειαζόμαστε περισσότερες καθαρές ενέργειες και μάλιστα με τον πιο αποδρικό τρόπο. Το 2050 το μερίδιο του ηλεκτρισμού στην κατανάλωση ελπίζουμε ότι θα έχει διπλασιαστεί. Χρειαζόμαστε σχετικές υποδομές για τον ηλεκτρισμό αλλά και για έξυπνες μορφές ενέργειας, ε, ολική, ενέργεια από τα κύματα, καταβόθρες άνθρακα και ούτω Το νέο πλαίσιο πρέπει να προάγει επίση την κοινοτομία. Σα διαβεβαιώ ότι θα μιλήσουμε όλου του εμπλεκομένου στη διαμόρφωση αυτή τη πρόταση και εννοείται θα συμμετάσχει και το Κοινοβούλιο από την αρχή. Θα κάνω λοιπόν ό,τι μπορώ για να επιταχύνω αυτήν την διαδικασία. χωρί όμω υποχωρήσεις. Γι' αυτό και ο στόχο μα, όπω είπε, είναι ο Δεκέμβριο του 2020 για την έγκριση του σχετικού κανονισμού. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξουν αυτέ τι προτάσει, θα τι εξετάσουν το συντομότερο δυνατόν, θα τι αντιμετωπίσουν ω προτεραιότητε, όπω άλλωστε έκαναν και στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε τον πέμπτο κατάλογο του 2021. Γι' αυτόν τον λόγο όμως συζητούμε την επιλογή των έργων του πέμπτου καταλόγου έργων κοινού ενδιαφέροντος. Θέλουμε να αντικατοπτρίζουν ακριβώς την πράσινη συμφωνία. Δηλαδή πρέπει να είναι βιώσιμα, να πληρούν κριτήρια βιωσιμότητας, να είναι έργα στα οποία θα λαμβάνουν υπόψη μα τι εκπομπέ άνθρακα και μεθανίου. Επίση θα ενσωματώσουμε περισσότερα έργα ενεργειακή μετάβαση. Ιδιαίτερα έξυπνα έργα για την συλλογή του διοξιδίου του άνθρακα. Θα κάνω ό,τι μπορώ προ την κατεύθυνση αυτή. Και τέλο θα διευκολύνω τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιλογή των έργων. Ακόμα και σε περιφερειακό επίπεδο η Επιτροπή σα και εγώ θα συνεχίσουμε να μιλάμε. Στόχος μας κοινό είναι καινοτόμα έργα, χωρίς άνθρακα, που θα επιτρέψουν την περαιτέρω ένταξη του ηλεκτρισμού σε έξυπνα δίκτυα. Το θέμα είναι τι θα γίνει με την χρηματοδότηση αυτών των έργων. Πρώτα απ' όλα τα έργα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως έργα κοινού ενδιαφέροντος για να μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα διορθωτικά ταμεία. Θα σε για την διαδικασία αυτή και τη διαδικασία αξιολόγησης. Ξέρω ότι ήδη δίνεται προτεραιότητα σε έργα ηλεκτρισμού. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, σα είπαμε δύο λόγια τη απόψη μου για το μέλλον. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα υπερψηφίσει τον πέμπτο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντο, στον οποίο περιλαμβάνονται βασικά έργα μεγάλου ενδιαφέροντο που θα αυξήσουν το μερίδιο των ανανεώσιμων μορφών ενέργεια. Θα βελτιώσουν την ασφάλεια του εφοδιασμού και θα προωθήσουν τον εξυγχρονισμό των ενεργειακών μα υποδομών. Τα έργα εξηλεκτρισμού είναι τρία τέταρτα του συνόλου των έργων. Η αντίρρηση περί του πέμπτου καταλόγου σημαίνει ότι αναγκαστικά θα κινηθούμε με βάση τον τρίτο κατάλογο και δυστυχώ εκεί έχουμε 40% περισσότερα έργα που βασίζονται σε, που προκαλούν εκπομπές γι' αυτό λέω ας υποστηρίξουμε τον εξηλεκτρισμό και τα έργα μετάβασης όπως ε, τα έργα αιωλικής ενέργεια στην Βόρειο Θάλασσα και θα είναι κρίμα πραγματικά να μην χρηματοδοτηθούν αυτά από το Συνδέοντα στην Ευρώπη. Έχουμε μπροστά μας μια πολιτική για το μέλλον. Εγώ θα συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου. Περιμένω τις απόψεις σας, τις γνώμες σας για να βελτιώσουμε αυτή την πολιτική, να είμαστε ο κινητήριος μοχλός που θα κάνει την Ευρώπη ουδέτερη ενεργειακά. Ευχαριστώ. Εδώ Προχωρούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος το λόγο έχει η κυρία Καρβάλιο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Πρέπει να αναθεωρηθούν αυτές οι κατευθυντήριες για αυτά τα έργα και αυτό να είναι κάτι το οποίο να συνάδει με τους στόχους μας για το κλίμα, για το περιβάλλον και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους στόχους, ε, τους στρατηγικούς και βιώσιμους ε, για ε, μια ενεργειακή αποτελεσματικότητα, έρευνα, λογικές τιμές ε, και να σταματήσουμε να έχουμε τεχνολογίες άνθρακα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα δημοσιοποίησε αυτό τον τέταρτο κατάλογο των έργων ε, κοινού ενδιαφέροντος. Δεν λαμβάνεται όμως ε, υπόψη ο στόχος της κλιματικής αλλαγής. Την Τετάρτη πρόκειται να γίνει ψηφοφορία για αυτή τη λίστα. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι εάν απορριφθεί αυτή η λίστα, τότε τι θα γίνει. Ε, μιλούμε για 40% περισσότερα έργα φυσικού αερίου, όπως είπατε, Επίτροπε. Και επομένως έχει χαμηλώσει ο πύχη σε σχέση με τους ε, στόχους μας. Εγώ ζητώ να γίνει μία τροποποίηση, μία αναθεώρηση ε, για κάποια από αυτά τα έργα. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι είναι μεγάλες οι ανάγκες ορισμένων περιοχών, περιφερειών Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών η κυρία Ντάλη για δύο λεπτά. Thank you, Chair, Commissioner. Ευχαριστώ. Επίτροπε, συζητάμε συγκεκριμένα έργα που πρέπει να ευθυγραμμίζονται με αυτά που συζητούσαμε εδώ πριν από λίγες εβδομάδες στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Θέλουμε το 2050 να είμαστε ουδέτεροι ως προς τον άνθρακα. Άρα πρέπει να επενδύσουμε σήμερα στη σωστή υποδομή. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό συνειδητοποιώντας ε, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα παντού. Πρέπει να κατανοήσουμε ταυτόχρονα ότι χρειάζονται επενδύσεις σε πιο ε, καθαρές ε, πηγές. Στην, ε, στον κατάλογο που συζητάμε υπάρχουν ακόμα ε, έργα εφοδιασμού με πετρέλαιο. Χρειάζεται βέβαια να υπάρχει συνέχεια του εφοδιασμού η αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών που είναι αποσυνδεδεμένα μέχρι σήμερα μεταξύ τους. Αλλά ο τέταρτος κατάλογος πάει πιο μακριά και ανοίγει την πόρτα για αγωγούς και υποδομές που στηρίζονται στα ορυκτά καύσιμα. Τα πράγματα άρα, άλλαξαν πολύ από τότε που δημιουργήθηκε ο τέταρτος κατάλογος. Ε, τα, ε, ε, υπάρχουν κράτη-μέλη που αμφισβήτησαν ένωση, αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτό λείπει από τη διατύπωση του καταλόγου. Τώρα, ο κατάλογος των έργων δεν είναι αυτό που χρειάζεται. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε έργα που θα μας βοηθήσουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτούς τους λόγους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει όλες τις αξιολογήσεις βιωσιμότητας που χρειάζονται, ώστε τα χρήματα να επενδύονται σε έργα που θα κάνουν την Ένωση το 2050 ουδέτερη ως προς τον άνθρακα. Έτσι θα φροντίσω, πρέπει να φροντίσουμε ότι θα έχουμε έργα που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους μας στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας. Ομάδα Renew Europe, το λόγο έχει ο κύριος Πέτερσεν για δύο λεπτά τα uh, πω στα δανέζικα, Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα. Χαίρομαι που βλέπω ότι η Επίτροπος είναι κάπως ε, καλύτερα στην υγεία της κατόπιν του ταξιδιού την περασμένη εβδομάδα στην πατρίδα μου. Εκεί είχατε την ευκαιρία να δείτε ε, τι κάνουμε όσον αφορά την ολική ενέργεια στην Βόρειο Θάλασσα, Επίσης, ε, διαπιστώσατε ότι χρειαζόμαστε διασυνοριακές επενδύσεις στην περιφερειά μας, οι οποίες επενδύσεις θα πρέπει σε σχέση με τα έργα που συζητούμε τώρα να είναι στο επίκεντρο της προσπάθειας. Ενιαία αγορά στην ενέργεια. Αυτό χρειάζεται, να συνδέσουμε τις αγορές. Η πράσινη αλλαγή, η πράσινη μετάβαση είναι ολόκληρο πολιτικό κίνημα που πάει προς τα εκεί να ε, εντοπίσουμε στο πού πρέπει να επενδύσουμε. Γι' αυτό συστάμε ε, αυτό το σημαντικό ζήτημα απόψε, να γίνουν οι σωστές επενδύσεις. Όχι μαύρες, πράσινες επενδύσεις. Όχι επενδύσεις σε έργα που τελικά παραμένουν μαυσολία. Οπότε ανανέωση και πρόοδος αλλά πρέπει να αλλάξουν τα κριτήρια που έχουμε για τις ε, επενδύσεις. Και να είμαστε φυσικά στη γραμμή της Συμφωνίας των Παρισίων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο μπορεί να εξετάσει τα έργα αυτά και να εξασφαλίσει ότι ό,τι κάνουμε βοηθάει για τους στόχους μας. Χαίρομαι που είπατε Επίτροπε ότι θα επιταχύνεται τη διαδικασία αλλαγής των κριτήριων. Επίγει το θέμα. Πράσινες επενδύσεις. Επίσης, συμφωνούμε με τους ε, προλαλήσαντες. Προτιμούμε αυτή την γραμμή τέσσερα. ID, το λόγο έχει για 1,5 λεπτό Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πρέπει να, είμαστε, να λειτουργήσουμε ως κοινοβούλιο, να περιορίσουμε τα λόμπι. Δύο παράγοντες είναι σημαντικοί. Πρώτον, ε, ευνοϊκός ενεργειακός ε, εφοδιασμός και ασφαλής. Ε, γι' αυτό χρειάζεται διαφοροποίηση. Οι εξαρτήσεις πρέπει να αποφεύγονται. Ο ενεργειακός εφοδιασμός θα πρέπει να στηρίζεται σε πολλές πηγές και το LNG δεν θα πρέπει να αποκλείεται. Ακούω ότι οι πράσινοι θέλουν ε, διαφορετικά έργα, ε, μειώνοντας ε, την συμβολή των ορυκτών καυσίμων. Όμως έχουν σκεφτεί ότι μπορούν έτσι να καλύψουν τον ενεργειακό εφοδιασμό. Επίσης χρειάζεται μείωση του κόστους. Δεν γίνεται ιδιωτικές επιχειρήσεις ε, να ε, μεταφέρουν στους φορολογουμένους τα βάρη των επενδύσεων. Ένα πρέπει να είναι σαφές. Ο εφοδιασμός σε ενέργεια και, ε, και ηλεκτρική ενέργεια είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν θα πρέπει να σημαίνει αυτό ότι θα πέσω με στα χέρια εκβιαστών στην πολιτική αυτή. Ο κύριος για ένα λεπτό. Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Πρέπει να πω, όταν διάβασα την Πράσινη Συμφωνία της Κομισιόν φάνηκε πολλά υποσχόμενη. Δηλαδή νέος δρόμος προς νέα οικονομία της Ευρώπης. Απομάκρυνση από επιδοτήσεις βλαβερές. Παράλληλα όμως ε, υπογραμ... Ε, ε, προστατεύομαι εδώ τον τέταρτο κατάλογο που βεβαίως είναι επιδοτήσει για τα ορυκτά καύσιμα. Δηλαδή στηρίζεται περισσότερο τα ορυκτά καύσιμα. Πού είναι η υπόσχεση για το νέο δρόμο Ακόμα και στην ομιλία σας ε, ε, είπατε ότι όλα θα γίνουν καλύτερα όταν πάμε στον πέμπτο κατάλογο, αλλά τώρα πρέπει να δεχτούμε τον τέταρτο κατάλογο. Δεν φαντάστηκα εγώ έτσι τη νέα κομισιόν, μια φιλόδοξη κομισιόν. Οι συνάδελφοι έλεγαν ότι εντάξει δεν είναι ιδεώδη τα πράγματα, αλλά α προχωρήσουμε έτσι. Οι ίδιοι όμως έλεγαν πριν από ε, μήνες ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση τώρα, υπάρχει κατεπίγουσα ανάγκη. Τώρα το αποτέλεσμα είναι ότι ενισχύουμε περισσότερο τα ορυκτά καύσιμα που θα μας κάνει πιο εξαρτημένοι και δεν θα έχουμε ουδέτερη οικονομία ως προς το κλίμα που τη χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Η νέα... Αυτά τα έλεγε η παλιά Κομισιόν. Η νέα Κομισιόν μπορεί να... Για την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών το λόγο έχει ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η προπαρασκευή για αυτό το πρόγραμμα είναι μία επένδυση. Είναι μία επένδυση εύστοχη. Έτσι έχουμε αγωγούς φυσικού αερίου. Όμως οι συνάδελφοι δεν θέλουν το φυσικό αέριο θέλουν να απαλλαγούν από αυτό. Μα αυτό είναι αφελές, αυτό που πιστεύουν. Θέλουν ε, αιωλική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, ναι, αλλά τι γίνεται. Χρειάζεται πλάν B όταν δεν έχουμε αρκετό αέρα, αρκετό ήλιο. Οπότε αυτό το οποίο χρειάζεται μια λύση αξιόπιστη όσον αφορά την ενέργεια, μια ενέργεια σε λογικές τιμές, κάτι που είναι σημαντικό για την οικονομία. Έτσι λύσαμε το πρόβλημα στην ε, Ολλανδία και έχουμε 8 εκατομμύρια συμπατριώτες μας και έτσι... Της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, το λόγο κυρία Ρέγκο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο παρελθόν θα ήταν αδιανόητα να καμία τέτοια συζήτηση και αυτό το δυνατό, κυρίω λόγω των νέων οι οποίοι δίνουν την όθηση στα πράγματα και κατεβαίνουν στο πεζοδρόμιο και αυτό και η δική μας πολιτική ομάδα ε, θεώρησε ότι σήμερα θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτή την ένσταση για τα έργα τούτα. Αλλιώς δεν θα υπήρχε δικαιολογία από πλευρά περιβάλλοντος ή οικονομία. Τι γίνεται στον Βυσκακό κόλπο. Είναι τεράστιο φαραωνικό το κόστος και θα ωφεληθούν από αυτό το έργο μόνο κάποια ολιγοπόλια. Δεν θα λυθεί το ενεργειακό πρόβλημα της ε, Ισπανίας. Για όλους αυτούς τους λόγους παρακαλώ να ξαναβρούμε αυτό το πνεύμα, το πνεύμα της νιώτης της νεολαίας που δίνει τη μάχη στον δρόμο και έτσι να έχουμε κάποια έργα τα οποία να βοηθούν τόσο ώστε να έχουμε την ανάπτυξη στις πατρίδες μας. Στον ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων, το λόγο έχει ο κύριος Κοράου για ένα λεπτό. Thank you, Mr. Chair. <clears throat> As one of the 17 MEP ως ένας από τους βουλευτέ υπέρ του ΒΕΤΟ κατά του τετάρτου καταλόγου επιβεβαιώνω αμετάκλητα την πρόθεσή μου να καταψηφίσω τον πέμπτο κατάλογο. Μετά από τόσες υποσχέσεις για ένα πράσινο μέλλον βλέπω πού φτάνουμε σήμερα. Να είμαστε σαφείς. Επιτρέψαμε αυτόν τον τέρτο κατάλογο. Επιτρέψαμε την επαναφορά από το παράθυρο των ορυκτών καυσίμων. Δισεκατομμύρια σε εγκαταστάσεις που θα είναι πεπαλαιωμένες σε πολύ λίγα χρόνια. Ας πούμε λοιπόν όχι στον καταλόγο αυτών και ναι στις φιλοδοξίες των νέων ανθρώπων που βγήκαν στους δρόμους και που ζητούν ένα πιο πράσινο μέλλον. Δεν μπορούμε να τους αγνοήσουμε. Πρέπει να σταματήσουμε να δείχνουμε αδιαφορία προς αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό και Υποστηρίζω την αντίρρηση και με κατά του καταλόγου των έργων που είναι προσβολή για τη νέα γενιά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Πίπερ για 1,5 λεπτό. Μάικρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι θέλουμε την ενεργειακή μετάβαση όσο γίνεται πιο γρήγορα και γι' αυτό χρειάζονται διασυνοριακά δίκτυα, κατασκευάζομαι ε, στα σύνορα δίκτυα. Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος είναι πολύ σημαντικά για μια γνήσια εσωτερική αγορά που τη χρειαζόμαστε πολύ. Όμως προετοιμάζει και την εποχή του υδρογόνου. Ε, γι' αυτό χρειαζόμαστε ενεργειακή αποθήκευση, χρειαζόμαστε ιδιαίτερα στην Ανατολική ε, ε, Ευρώπη ε, όλα αυτά. Για να περάσουμε στις ανανεώσιμες πηγές ε, χρειαζόμαστε ευέλικτα ε, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι πράσινοι, πώς μπορούμε να είμαστε κατά. λένε δεν επενδύουμε στο αέριο, δεν επενδύουμε στα ορυκτά καύσιμα, ε, με το κατάλογο. Αυτό είναι λαϊκισμός που μετά θα επιστρέψει στις βασικές μας γραμμές. Χρειαζόμαστε ε, ε, το αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια. Ε, σίγουρα υπάρχει όμως υπεραξία ε, στις πολιτικές μας και αυτό το κάνουμε γιατί είμαστε σοβαροί σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα και την αξιοπιστία. Για 1,5 λεπτό. Grazie Presidente. ci rendiamo conto che questa lista contiene anche... Να συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται εδώ πέρα για κάποια πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα σε ε, αυτή την ε, λίστα. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι η τα μέλη της ΣΥΤΡΕ των Σοσιαλδημοκρατών έχουμε κάποια ισορροπία ισορροπία στη λίστα, γιατί υπάρχουν κάποια έργα χρήσιμα για την ε, μετάβαση. Είναι ενδεικτική αυτή η λίστα, γιατί δεν θα εγκριθούν όλα αυτά τα έργα, αλλά θα πρέπει να εξεργαστείτε αυτή την ε, λίστα. Μην την ε, θεωρείτε μία βίβλο. Επίση τι θα κάνουμε. Πάμε στον κατάλογο τον προηγούμενο, τον τρίτο, για να απορριφθεί αυτό ο κατάλογος ο τέταρτο. Όμως ο τρίτο είναι χειρότερο πλέον περιβάλλοντο. Άρα θα πρέπει να στρωθούμε στη δουλειά. Γιατί ε, η επόμενη λίστα και αυτή η λίστα εμπλέκει πολύ το κοινοβούλιο. Άρα θα πρέπει να σκεφτείτε ότι έχετε μέχρι το Μάρτιο ένα περιθώριο και θα πρέπει να αλλάξετε κάποια σημαντικά έργα, της προτεραιότητες, αλλά να αποφασίσετε και για τη μεθοδολογία. Γιατί στις επόμενους, στόχους θα πρέπει να λάβετε υπόψη το περιβάλλον και την κλιματική επιβαλλοντική μετάβαση και την εγκατάλειψη του άνθρακα. Γι' αυτό και εμείς αυτή την ένσταση. Λόγο έχει κύριος Γκρούντλερ για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να αναπτύξουμε τα διενεργειακά δίκτυα για να δώσουμε στους πολίτες μας προσιτή ενέργεια με ασφάλεια και με βιωσιμότητα, με εφορία. Εάν καταψηφίσουμε τον κατάλογο, επανέρχεται ο κατάλογος του 17 με 53 έργα για το αέριο, έναντι 32 του σημερινού καταλόγου. Δεν είναι τέλειος ο σημερινός καταλόγος, αλλά βαίνει προς την κατεύθυνση του, της Πράσινης Συμφωνίας. Το 90% των νέων έργων είναι καλά έργα υπέρ του περιβάλλοντος. σας. μην το γνωρούμε αυτό. Και να σταματήσουμε τώρα το λαϊκιστικό ψυχόδραμα. Όχι στα έργα που αφορούν το αέριο ή τα ορυκτά καύσιμα. Τα ίδια δίκτυα αύριο θα μεταφέρουν πράσινα αέρια, φυσικό αέριο και άλλους πόρους. Ναι λοιπόν στο νέο κατάλογο. Ας βελτιώσουμε τα κριτήρια, ας βελτιώσουμε τη διαβούλευση με την Κομισιόν, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να καταρτήσουμε ήδη από σήμερα τον κατάλογο του 21, που θα είναι ένας πράσινος κατάλογος. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Πάουλους για ένα λεπτό. Thank you, Chair. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε που είστε ε, ε, Επίτροπε. Θα συνεχίσω στα γερμανικά ενημερώνω τους διερμηνείς. Πολλές φορές είπαμε ότι ο τρίτος κατάλογος είναι χειρότερος από τον τέταρτο. Αλήθεια είναι, δεν το αμφισβητεί κανείς. Αλλά τα μεγάλα έργα που υπήρχαν στον τρίτο κατάλογο είτε ολοκληρώθηκαν είτε διακόπησαν προπολού. Άρα όταν πάμε πίσω στον τρίτο κατάλογο ε, αυτό δεν είναι τόσο κακό Είπα αυτή την έννοια. Επίσης ε, δεν είδε κανείς ε, τη μελέτη που πρόσφατα δημοσιεύτηκε και δείχνει ότι μέχρι το 2050 για να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες και να μπορούμε να μεταφέρουμε τις, ε, το υδρογόνο δεν χρειάζεται νέα υποδομή. Άρα λοιπόν όπως αναφέρθηκε εξοικονομούμε χρήματα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε για γνήσια ενεργειακή μετάβαση. Ε, ε, Το λόγο έχει η κυρία Κλοκ για ένα λεπτό. Ε, Αγαπητέ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, διαβάζουμε αυτή την λίστα, την υπαριθμούν τέσσερα και βλέπουμε ότι έχει προηγηθεί με διάφορους εμπλεκόμενους διαβούλευση με αντιπροσώπους των καταναλωτών αλλά και οργανώσεων που ασχολούνται με το περιβάλλον. Πρόκειται για ψήφισμα το οποίο δεν θα περάσει αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την παραγωγή του άνθρακα στην Ευρώπη. Ε, μέχρι το 19 έχει δημιουργηθεί το 24% και τώρα έχουμε τις ενώσιμες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται περισσότερο και είναι το μισό ε, των ε, ενεργειακών πόρων το άλλο μισό είναι το φυσικό αέριο. Έχουμε τον πύχη ψηλά, δεν μπορούμε να επικεντρωθούμε μόνο στο φυσικό αέριο αλλά δεν το καταλαβαίνουν αυτό οι χώρες Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα από το βράδυ μέχρι το πρωί, γιατί ακόμα θα χρειαστεί ο άνθρακας. χρόνο. Το λόγο έχει ο κύριος Μποτέγκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Να αλλάξουμε τους κανόνες τώρα. Μας παρουσιάζεται έργα τα οποία ρηπαίνουν, δισεκατομμύρια τα οποία πηγαίνουν σε έργα που σκοτώνουν. Μιλάμε για δηλητήριο για το περιβάλλον, δηλητήριο για τον πλανήτη, δηλητήριο για την εποχή μας, τα παιδιά μας. Προτείνω λοιπόν να επενδύσουμε τα χρήματά μας, τα χρήματα των φορολογουμένων, όχι στο δηλητήρια. Ας πάρουμε αυτά τα κονδύλια και ας τα βάλουμε στις ε, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Αλλιώ ο κόσμο δεν καταλαβαίνει. Και είναι και κάτι άλλο το οποίο με ενοχλεί. Την περασμένη εβδομάδα συζητούσα με συναδελφού σα στην Κομισιόν και έθεσα το ερώτημα. Ε, τι μου είπαν. Δεν θα πάρω σοβαρά αυτή την απάντηση. Ε, μου είπε να φορολογήσουμε περισσότερο για να βρούμε χρήματα. Μα είναι, είναι δυνατόν να βάλουμε φόρους επί αυτών των έργων. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Σίντσιτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Μιλάμε εδώ για στρατηγικά έργα, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσουν τους πολίτες και τα νοικοκυριά. Θα μιλήσω για ένα έργο το οποίο ε, πάει ενάντια στον κατάλογο αυτών και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως το έδαφος του κράτους δικαίου. Είναι στο νησί του Κέρκ που ε, αυτό το έργο δεν είναι καθόλου οικονομικό, είναι φρικτό και αντιβαίνει ε, ενάντια στα συμφέροντα του νησιού και ενάντια στα συμφέροντα των πολιτών. Επίσης, αντιβαίνει τη σύμβαση του άρχους, σύμφωνα με την οποία ο κόσμος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συναποφασίζει. Δεν ξέρω πώς κατέληξε να μπει στον κατάλογο το έργο αυτό. Θα πρέπει να υπάρχουν δύο χώρες υπέρ του έργου. Εκτός από την Κροατία, κανένας δεν ήταν υπέρ. Ε, μιλάμε για 2,5 δις κυβικά μέτρα αερίου που κανείς δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει αργότερα. Αν... Ε, Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπέρεντσεν για 1,5 λεπτό. Συνάδελφοι, είναι δύσκολη αυτή η υπόθεση και θα πετύχουμε μόνο να κάνουμε τις σωστές επιλογές και να προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Ε, μιλώ για τις ε, λύσεις, για τις επενδύσεις που πρέπει να είναι κάτι το εφικτό. Δεν μπορούμε με μια γραμμή να σβήσουμε κάποιους ενεργειακούς πόρους γιατί απλώς δεν μας αρέσουν και η αποθήκευση των πόρων είναι πάρα πολύ σημαντική άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα επενδύσουμε στη Βόρεια Θάλασσα. Επίσης είναι καλή η ιδέα να μετακινηθούμε σε κάποιες χώρες από τον άνθρακα στο φυσικό αέριο. Αυτό γίνεται. Αυτό ε, έχει ένα κόστος λογικό. Είναι μια λογική επιλογή να επενδύσουμε στις ε, υποδομές στην Ευρώπη. Έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι ε, όχι σε επίπεδο κράτου μέλους, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τα κράτη-μέλη ας κάτσουν να αποφασίσουν πώς θα παράξουν ενέργεια, οπότε θα πρέπει ε, όλοι να δούμε τι θα κάνουμε σε κάθε φάση που κορυφώνεται η ζήτηση ή όταν είναι λίγη και αυτό θα χρειαστεί ευελιξία και δεν μπορεί αυτό να το κάνουμε μόνοι μας για να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος θα πρέπει όλοι να συμμετάσχουν και αυτό θα το καταφέρουμε μόνο άμα τους εμπνεύσουμε, τους δώσουμε κίνητρα και να εξασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε σωστές επιλογές. Χάισελ για 1,5 λεπτό. pán Ja chápem že... Καταλαβαίνω γιατί υπάρχει προβληματισμός θα πρέπει να επενδύσουμε σε εναλλακτικέ πηγέ ενέργεια, όχι μόνο σε ορυκτά καύσιμα, αλλά αυτή η λίστα υπερθύμων 4 αποτελεί βήμα πρόοδο σε σχέση με την τρίτη, την προηγούμενη λίστα που είχε πάνω από 50% ε, σχεδόν 30% έργα ε, φυσικού αερίου. Τώρα στον τέταρτο κατάλογο έχουμε 40% λιγότερα. Άρα ε, θέλουμε τώρα διασυνδέσεις, ηλεκτρικά δίκτυα, διασυνδεόμενα δίκτυα και ξέρω ότι αυτή η πρόταση δεν είναι τέλεια, αλλά είναι μια καλή αρχή. Έτσι μπορούμε να πλησιάσουμε τους στόχους που έχουμε τάξει στη νέα πράσινη συμφωνία. Όμως, εάν εγκρίνουμε ε, αυτό τον κατάλογο, θα πρέπει να επιμείνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, να θεωρήσει τα σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα ε, γιατί τα κριτήρια επιλογής που υπάρχουν ε, σήμερα δεν είναι σωστά. Άρα θέλουμε και στην επόμενη λίστα να καλυφθούν έργα για ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας, για διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας και ευφυή δίκτυα. Αυτό είναι πρόοδος, αν θέλουμε να πλησιάσουμε στους στόχους της Νέας Συμφωνίας. Αυτό το λόγο ο κύριος Χόησιτ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσαμε να περιμένουμε μέχρι να εκδοθεί ο εξαιρετικό αυτός πέμπτος κατάλογος, θα ήταν όλα πράσινα, αλλά τι μα λένε οι επιστήμονες. Μας λένε να ακούσουμε τους επιστήμονες, όχι τον κοσμάκι. Ωραία, ναι, να ακούσουμε τους επιστήμονες, οι οποίοι μα λένε δεν υπάρχει χρόνο να περιμένουμε ω τον πέμπτο κατάλογο. Κάθε ευρώ που έχουμε στη διάθεσή μας πρέπει να πάει στη μετάβαση. Δεν μπορούμε να πετάμε χρήματα από το παράθυρο. Δεν μπορούμε να ζήσουμε πια με αυτόν τον τέρτο κατάλογο. Βεβαίω δεν είναι όλα μαύρο-άσπρο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν περισσότερα καλά έργα σε σχέση με το παρελθόν. Τι πρέπει να κάνουμε. Πολύ απλά να απορρίψουμε τον κατάλογο και η Επιτροπή σα να καταρτήσει αμέσως μια νέα εκδοχή του τετάρτου καταλόγου όπως πρέπει που να πηγαίνει προς την Πράσινη Συμφωνία. Και αυτό μπορείτε να το κάνετε για την Ευρώπη και τον πλανήτη. το λόγο έχει ο κύριος Ροπέ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε, συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε. Λυπούμε διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα ή να στηρίξει ή να απορρίψει όλο τον κατάλογο των έργων, χωρίς να εξειδικεύσει συγκεκριμένα έργα. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που μίλησαν για τις μεγάλες επενδύσεις στην ε, υποδομή αερίου. Συμφωνώ με τον κατάλογο γιατί συμπεριλαμβάνει ένα έργο εξυγχρονισμού της ηλεκτρικής ενέργειας που στο μέλλον θα βοηθήσει να αναπτύξουμε αιωλικό δυναμικό στη Βαλτική. Για το πέμπτο κατάλογο θα ήθελα να δω εκεί κατευθυντήριες γραμμές για την διατλαντική ενεργειακή υποδομή. Ώστε και ε, καλό είναι να... έχει ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, να σας πω μια ιστορία. Ήταν ε, μια κομισιόν που υποτίθεται υποστήριζε τους ε, νέους που είχαν ως προτεραιότητά της την μετάβαση προς ένα πιο οικολογικό μέλλον. Και μας έδωσαν και μια υπόσχεση, την ε, πράσινη συμφωνία, για να μας αποδείξουν ότι το εννοούν. Και όμως ήρθε η ώρα των αποφάσεων και άλλα έγιναν. Είπε η Κομισιόν, ε, όχι πολύ γρήγορα, να μεταρρυθμίσουμε την υγειοργική πολιτική. Πολύ αργά. Να σταματήσουμε τα ορυκτικά καύσιμα. Ε, θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Η Κομισιόν, λοιπόν, υποστηρίζει σήμερα πιο πολλά έργα για τα ορυκτά καύσιμα. Ως εάν δεν υπήρχε άλλη λύση. Έτσι θα φτάσουμε το 2050 στην ενεργειακή ουδετερότητα. Ναι, αλλά να μην ενοχλήσουμε τα λόμπι του φυσικού αερίου. Λοιπόν, αυτή η λυπηρή ιστορία πρέπει να τελειώσει. Πείτε όχι στα αντικολογικά σχέδια και μιλήστε επιτέλους τη γλώσσα της αλήθειας. Να είμαστε αυτοσυνεπείς. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Νίμπλερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Η Πράσινη Συμφωνία θα λειτουργήσει μόνο με σταθερό ενεργειακό εφοδιασμό. Γι' αυτό χρειάζεται ενεργειακή υποδομή και ε, γι' αυτό χρειάζονται τα έργα που αναφέρονται στον κατάλογο. Εγώ υποστηρίζω τον κατάλογο αυτό με βάση αυτά που είπατε κύριε Επίτροπε. Είναι σωστό ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε και τα έργα του αερίου. Είναι μια τεχνολογία γέφυρα το αέριο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Είναι μια χώρα όπως η Πολωνία ε, που πρέπει να φύγει από τη χρήση άνθρακα θα πρέπει να περάσει μέσα από μια μετάβαση ε, στο αέριο. Ε, συμφωνώ να επενδύσουμε σε αυτή τη μεταβατική τεχνολογία και για την τεχνολογία του υδρογόνου και εδώ νομίζω ότι χρειαζόμαστε ε, υποδομές, δεν έχουν κατασκευαστεί όλα. Και στη Βαβαρία, τη δική μου ιδιαίτερη πατρίδα, ακόμα δεν έχει κατασκευαστεί ούτε ένα χιλιόμετρο αυτών των αγωγών και χρειαζόμαστε, ε, τα χρειαζόμαστε κατεπηγόντως. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την πρόταση και παρακαλώ παρακαλώ τους συναδέλφους να προσέξουν πώς θα προχωρήσουν. Αν θέλουμε την πράσινη συμφωνία θα πρέπει να επενδύσουμε σε μια μεταβατική περίοδο στο αέριο. για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συναδελφοί. Δυστυχώς, η απάντηση πρέπει να είναι ένα ναι ή ένα όχι. Δεν μπορούμε να προκρίνουμε επιμέρους έργα και εκεί έχω πολλά να πω. Πρώτον, δεν έγιναν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ποιες είναι οι επιπτώσεις του σημερινού καταλόγου επί της Πράσινης Συμφωνίας. Φοβούμε ότι τα επόμενα 10 χρόνια θα ζήσουμε με τα ορυκτά καύσιμα θα ξοδέψουμε δισεκατομμύρια από τα χρήματα των φορολογουμένων για τέτοιου είδους έργα. Και επειδή μιλάμε για χρήματα φορολογουμένων, ο σημερινός κατάλογος περιέχει πάνω από 20 έργα στον Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία δεν συνδέονται καν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα χρηματοδοτούμε το Ηνωμένο Βασίλειο και την Νορβηγία, όταν ξέρουμε ότι άλλε περιφέρειε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται χρήματα για τη μετάβαση. Ο μόνο τρόπο να ενημερώσουμε τον κατάλογο είναι να καταψηφίσουμε τον παρόντα. Θέλουμε έναν κατάλογο που υπηρετεί το κοινό συμφέρον. Μια αηφορική Ευρώπη. Από τη συνάδελφη ψηφίστε όπως εγώ. Κατά. Υπέρ της αντίρρησης. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Νιίστο για ένα λεπτό. Mr. President, three months ago in this parliament... Πριν από τρεις μήνες, ε, Πρόεδρε, εδώ στο Κοινοβουλίο, κηρύξαμε την επίγουσα κατάσταση για το κλίμα των συναγερμών και ήρθε μετά η Κομισιόν και είπε ότι η απάντηση είναι το, η νέα πράσινη συμφωνία ε, που υποτίθεται είναι φιλόδοξη και σήμερα βλέπουμε αυτόν τον κατάλογο έργων που έχει χρηματοδότηση έργων ορυκτών καυσίμων. Αυτό ε, δεν αντιστοιχεί σε κάποια πρωτοπορία που προσδοκούμε από εσά. Είναι προδοσία, είναι διάψευση του ίδιου του εαυτού σας αυτοδιάψευση. Οπότε δεν θα πρέπει να συνεχίσετε τα λάθη του παρελθόντος, θα πρέπει να επενδύσετε στο μέλλον. Και είχαμε αυτή την έκθεση που έλεγε ότι οποιαδήποτε τέτοια ε, επένδυση είναι λάθος όπως και αυτή η αγωγή φυσικού αερίου. Χρειαζόμαστε βιώσιμη ε, επένδυση σε πράσινους, σε, πράσινου, σε βιώσιμους πόρους. Αυτό πρέπει να κάνουμε. έχει ο κύριος Γουάλλας για ένα λεπτό. Αυτό είναι η πιο κρίσιμη στιγμή μας. Έχουμε αυτή την λίστα των έργων που περιέχει 55 έργα ορυκτών καυσίμων. Και λέτε ότι θα έχουμε ασφάλεια παροχής με φυσικό αέριο. Μα ήδη έχουμε τέτοια υποδομή για φυσικό αέριο για την ασφάλεια της ε, παροχής φυσικού αέριου Οπότε έχουμε 39 δις που θα επενδύσουμε σε τέτοια αχρίαστα έργα. Δεν είναι καύσιμο για την ενεργειακή μετάβαση. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή τη φάση και τον άνθρακα. Αυτά είναι μη ασφαλείς λύσεις. Όλα αυτά θα είναι αγώγημα στα κράτη-μέλη. Θα ακυρωθούν αυτά τα έργα και κάνατε αυτή τη λίστα χωρίς να λάβετε υπόψη το περιβάλλον. Εάν δεν εγκρίνουμε αυτό, τότε σημαίνει ότι δίνουμε δεκάρα για τη Συμφωνία των Παρεσίων και ότι η Πράσινη Συμφωνία... Το λόγο έχει η κυρία Βάις για μισή λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί επιτροπέ, Η πράσινη μετάβαση έγινε τώρα ε, ένα λόγος ε, για να τσακωνόμαστε. Ε, και αυτό για, να, για λόγους προβολής. Βλέπουμε πράσινο λαϊκισμό εδώ κατά τη συζήτηση του καταλόγου. Και δεν είναι καλό αυτό για την πράσινη μετάβαση. Ο ο τέταρτος ε, κατάλογος ε, προβλέπει έργα για την Νορβηγία, την Αγγλία, τη Γαλλία, ε, έργα που μπορούν να καλύψουν το 20% των ενεργειακών αναγκών. Αυτό, αν το απορρίψουμε, θα αναβληθεί και δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Ε, ε, αυτοί που θέλουν να καταψηφίσουν είναι κατά των, το κατά των έργων με το αέριο παρά το γεγονός ότι θα παίξει το ρόλο της γέφυρας στη μετάβαση. 32 ε, είναι τα νέα έργα και 52 ήταν στο παλιό κατάλογο. Η μετάβαση ενεργειακή είναι πολύ σημαντική και δεν πρέπει να αφήνεται στα χέρια των πράσινων λαϊκισμών. Ε, χρειάζεται ασφαλής... Εδώ έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Κονσάλες Καθάρες. Κομισάρια... Κυρία Επίτροπε, θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση εάν η επόμενη λίστα πραγματικά ήταν αντικείμενο διαβούλευση με το Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, χώρες που δεν τηρούν τους στίχους για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 20 ε, θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειες γιατί έχουμε τους ουραγούς σε αυτή την προσπάθεια που δεν μπορούν να μας πούνε ότι θα σταματήσουν τον άνθρακα ότι τα πράγματα είναι έτσι απλά και δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το φυσικό αέριο. Θα πρέπει επομένω να σχεδιάσουμε για το μέλλον. Έχουν πάνω από 60% κατανάλωση τη ενέργεια που αφορά ε, ε καύσιμα. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει στην επόμενη γενιά και αυτό να γίνει με δίκαιο τρόπο και να μην έχουμε απογοητεύσεις και αρνητικές συνέπειες, ανανεώσιμες πηγέ ενέργεια, ε, ε ηλεκτρική ενέργεια, εφή δίκτυα, ηλιακή και ολική ενέργεια. Οπότε, τέρμα στην ε, τέταρτη λίστα και που θα πάμε στην τρίτη. Όχι είναι η απάντηση α, ε, λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια λέμε εμείς. Ε, αν δεν δώσετε ε, εγγυήσει για τα δίκτυα, τα ΕΦΗ, e, τίποτα. θα, πληρώσουμε, θα ψηφίσουμε κατά. Αλλιώς κορυδεύετε τον κόσμο. Να λάβετε υπόψη τους κλιματικούς στόχους Εγγύησεις για την ενεργειακή ασφάλεια για τα κράτη-μέλη. Κάντε κάτι για την ενεργειακή ουδετερότητα, φιλοδοξία, αλλά και αποφασιστικότητα. Τέρμα στον ε, άνθρακα. Αυτό είναι η πρώτη προτεραιότητα. Το λόγο κυρία Χάν για ένα λεπτό. Κυρία Επίτροπε, μας είπατε ότι στη διαδικασία των έργων πρέπει θέλετε να προχωρήσετε το ταχύτερο δυνατόν. Αυτό δεν φτάνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υποβάλλει κατάλογο με ενεργειακά έργα που πρέπει να είναι προς κοινό συμφέρον. 32 όμως είναι με ορυκτά καύσιμα. Ο κατάλογος αυτός μας δεσμεύει υπέρ των ορυκτών καυσίμων και κατά της Πράσινης Συμφωνίας, της Συμφωνίας των Παρισίων και τη γνώμη του Κοινοβουλίου. Ε, δαπανά τα λεφτά των ε, φορολογουμένων σε μια Ευρώπη που μέχρι το 2050 πρέπει να είναι ουδέτερη ως προς το κλίμα. Μεγάλος παραλογισμός. Θέλουμε ε, να φύγει αυτός ο κατάλογος της λίθινης εποχής. Θέλουμε ένα νέο κατάλογο. Τώρα, όχι το ταχύτερο δυνατόν, τα ε, Θέλουμε να αντικαταστήσουμε τα έργα με τα ε, ορυκτά καύσιμα, ε, με ευφυή δίκτυα, με ε, ηλεκτρική ενέργεια και θέλουμε να, στη βιομηχανική πολιτική της Κομισιόν να βρίσκεται στο επίκεντρο το, η προστασία του κλίματος. Αυτό το θέλουμε αυτή τη βδομάδα τώρα, εδώ και τώρα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Καφ για ένα λεπτό. Είπαμε έκτακτη ανάγκη και τώρα έχουμε μπροστά μας όλη τη δουλειά. Να ελοπίσουμε τη Συμφωνία των Παρισίων, να μειώσουμε τις εκπομπές κατά 55% στο 30%. Ε, δεν θα το κάνουμε με σταθμούς ε, για αέριο ή άνθρακα. Ούτε θα αφήσουμε το, ούτε αφήνοντας το μεθάνιο να κατακλείσει τον πλανήτη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να καταστρέφουμε τον πλανήτη. Οτιδήποτε δεν είναι συμβατό με την Πράσινη Συμφωνία πρέπει να καταργηθεί. Οπότε, υπεράκτια αιωλικά πάρκα, υψηλότερη απόδοση, χαμηλότεροι λογαριασμοί ρεύματο, να σώσουμε του Ευρωπαίου. Όλοι έχουμε να κερδίσουμε από αυτό. Λοιπόν, επίτροποι, αυτό και από την αρχή. Θέλω να καλωσορίσω τους νέους συναδέλφους από τους πράσινου και να καλωσορίσω και τους συνεκλογέντες ε, ε, Ιρλανδούς. Ναι, στο πράσινο κύμα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Καρασνοντέψκη για 1,5 λεπτό. Dziękuję panie przewodniczący, pani komisarz. Ε, moim zdaniem ten wniosek odrzuca. Ευχαριστώ. Επίτροπε, η πρόταση απόρριψης αυτού του καταλόγου, απόρριψης του τέταρτου καταλόγου, που μετά από μήνες διαβουλεύσεων προέκυψε και μετά από μήνες νομοθετικού έργου είναι κάτι που θα πρέπει να σταθμιστεί σε σχέση με την ε, ενεργειακή ασφάλεια και τους ε, περιβαλλοντικούς στόχους. Κάποιοι συνάδελφοι συνήθως από παρόμοιες χώρες που πάει καλά η οικονομία τους να λένε πράγματα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι αυτό το ψήφισμα ε, αντιστοιχεί στην κοινή λογική ή ότι διαπνέεται από κοινή λογική. Ε, δεν είναι ούτε συνεπές με τα νομοθετήματα που έχουμε εδώ εγκρίνει. Και γνωρίζω ότι Όταν μιλούμε για καθαρή ενέργεια, τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλουν κάποιες ε, διασυνδέσεις διασυνοριακές. Θέλουν να μειώσουν τις εκπομπές. Περί αυτού πρόκειται. Έτσι θα γίνει η ενεργειακή μετάβαση να φύγουμε από τον άνθρακα, να πάμε στο φυσικό αέριο. Να προσπαθήσουμε να έχουμε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών. Είναι αυτονόητο. Γραμμένων ομιλητών. Προχωρούμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Έχω δεχθεί οκτώ αιτήματα. Είναι αδύνατο να τα κάνω όλα αποδεκτά θα επιλέξω έναν από κάθε πολιτική ομάδα, τον πρώτο ή την πρώτη που δήλωσε ε, ενδιαφέρον. Το λόγο έχει η κυρία Σπυράκη για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε Σίμψον, ασφάλεια εφοδιασμού, διαφοροποίηση πηγών ενέργειας και ενέργειας σε χαμηλές τιμές για τους πολίτες και τη βιομηχανία είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους οφείλουμε να κινούμαστε εν ώψη της μετάβασης στην οικονομία χωρίς άνθρακα το. 2050. η διαδικασία της μετάβασης είναι απαραίτητο να υποστηριχτεί από έργα κοινού ενδιαφέροντος αλλά και από το καύσιμο μετάβασης που είναι το φυσικό αέριο. χώρες που καθορίζουν την επιτυχία του εγχειρήματος του green deal όπως η γερμανία στηρίζονται στην ενεργειακή ασφάλεια που προσφέρει το φυσικό αέριο στον τέταρτο κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται ο east med ο igb το fsru στην αλεξανδρούπολη και η αποθήκη φυσικού αερίου στην καβάλα. είναι όλα έργα μετάβασης και σημαντικής γεωπολιτικής σημασίας. καλύπτουν την ασφάλεια εφοδιασμού στην ελλάδα και είναι απαραίτητο να γίνουν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον δρόμο προς την πλήρη απολιγνητοποίηση. σημασία έχει οι υποδομές αυτές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για υδρογόνο και για πράσινο φυσικό αέριο όχι να πυροβολήσουμε σήμερα τα πόδια μας όχι να επιστρέψουμε στον τρίτο κατάλογο όχι να στερήσουμε από τις χώρες που δεν έχουν τις δυνατότητες τις οικονομικές τη δυνατότητα να προχωρήσουν στη μετάβαση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. σας ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Αρένα για ένα λεπτό. Καταλαβαίνω τους πολίτες που αρχίσει να μην μας πιστεύουν τους αιρετούς ε, ευρωβουλευτές. Πρόκειται για εμπορική συμφωνία που έχουμε κάνει με κάποια δικτατορία που καταπατεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και από την άλλη μεριά έχουμε 29 δις για το φυσικό αέριο σε αυτή τη λίστα. Τι γίνεται με το περιβάλλον. Μα αυτά δεν κολλάνε. Επίσης γνωρίζουμε ότι το 1 τέταρτο της ε, υπερθέρμανσης οφείλεται σε αυτές τις παλιές μορφές ενέργειας και επίσης ε, έχουμε ένα σώρο παραδοσιακές μορφές ενέργειας που μολύνουν την ατμόσφαιρα αλλά και τα ύδατα. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς ε, με τις δεσμεύσεις μας, συνεπείς με αυτά που λέει η επιστήμη. Χρειάζονται μέτρα θα πρέπει να απορρίψουμε αυτήν τη λίστα, αλλά θα πρέπει να έρθετε με έναν διαφορετικό κανονισμό και διαφορετική λίστα, κύριε Επίτροπε. Όχι, κυρία Ντέιλι, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύμφωνα με τους συναδέλφους που είπαν ότι πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που έχει να λάβει το Κοινοβούλιο. Εάν δεν απορρίψουμε τον κατάλογο, θα παραμείνει ως μνημείο υποκρισίας στον χρόνο. Γιατί έχουμε μπροστά μα κρατη τα οποία δεσμεύτηκαν να σταματήσουν να χρηματοδοτούν τα ορυκτά καύσιμα ως το 20 και ξαφνικά συμφωνούν να κάνουν ακριβώς το αντίθετο για τα επόμενα 40 χρόνια. Πρόκειται για τρέλα. Για μια ένωση που θέλει να είναι ως προς τον άνθρακα έως το 2050. Έχουμε άλλα έργα μετά, τα οποία δεν είναι βιώσιμα. Μιλάμε για 29 δισεκατομμύρια, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αλλιώ. Επίσης, η εισαγωγή αερίου από fracking με μορφή υγροποιημένου αερίου πρόκειται για τρέλα. Πέρα από τα θέματα ασφαλεία, πέρα από τα θέματα των επιπτώσεων στη μεταβολή του κλίματος. Όλα αυτά κατόπιν των πιέσεων του Τραμπ και των άλλων για να μην μιλήσω για την παρουσία στρατητικών στην Πολωνία. Αυτά δεν είναι για το περιβάλλον, κύριε Πρόεδρε. Το λόγο έχει κυρία Εύη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ή το ένα ή το άλλο. Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή καταλαβαίνει και κατέβασε όμως ε, αυτήν την λίστα που είναι ε, λάθος ε, και δεν λάβατε υπόψη ότι θέλουμε κάτι για το μέλλον, κάτι για την κλιματική αλλαγή. Ή από την άλλη μεριά είναι ένα μεγάλο ψέ, μεγάλη απάτη η νέα συμφωνία. Και τι γίνεται, θέλουν οι Ευρωπαίοι να ε, χρηματοδοτείτε τέτοιες πηγές ενέργειας όπως τα αρκετά κάψουν. Αυτό είναι απαράδεκτο. Σήμερα να κάνετε τέτοιες υποδομές ε, και να γίνονται αυτά μαυσολία ως επενδύσεις, όχι θα πρέπει να κάνετε κάποιες υποδομές ε, όχι σαν και αυτές που ήδη υπάρχουν, δηλαδή νέους αγωγούς για το φυσικό αέριο. Εσείς οι ίδιοι έχετε κάνει κάποια προγνωστικά, τη στρατηγική, την μακρόπνοη, που λέτε τι πρέπει να γίνει για να ε, καλύψετε 90% της ανάγκης. Εμείς δεν είναι δυνατόν να εγκρίνουμε αυτή τη λίστα γιατί είναι σαν να κορδεύουμε τον κόσμο τη λίστα της Κομισιόν. Θα την απορρίψουμε, δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε αυτό το λάθος, δεν έχουμε χρονικά περιθώρια. Το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής έχει η Επίτροπος κυρία Σίμψον. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, άκουσα πολύ προσεκτικά. Έχω να πω τα Άκουσα διστάμενες απόψεις επί του καταλόγου έργων Εκείνη όμως ήταν η έκκληση για περισσότερες δράσεις, περισσότερη φιλοδοξία για το περιβάλλον. Η Κομισιόν συμμερίζεται αυτή την έκκληση. Δεσμευόμαστε να κάνουμε την Ευρώπη την πρώτη ενεργειακά ουδετερία προς τον άνθρακα το 2050. Και χαίρομαι που οι περισσότεροι από εσά υποστηρίζουν το ε- σχέδιο αυτό της Κομισιόν να τροποποιήσει ως τον Δεκέμβριο του 2020 τον σχετικό κανονισμό γιατί χρειαζόμαστε πιο έξυπνες υποδομές, πιο αιφορικές υποδομές για να διευκολύνουμε τη μετάβαση στον τομέα της ενέργειας, να περάσουμε στις, σε περισσότερες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Έτσι θα φυγραμμίσουμε και τα διευρωπαϊκά δίκτυα με τον στόχο μας που είναι η προστασία του κλίματος. Θα υποστηρίξουμε επενδύσεις οι οποίες θα αποφέρουν περισσότερες λύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της καινοτομία. Ως προς τον τέταρτο κατάλογο, ο τέταρτο κατάλογος, κοιτάξτε, είναι άλλο ένα βήμα προς τα εμπρός, προς πιο καθαρές υποδομέ. Υποστηρίζουμε έργα ηλεκτρισμού, περισσότερες ανανεώσιμες, περισσότερα έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα. Και έχουμε στο μυαλό μας φυσικά την Πράσινη Συμφωνία. Γι' αυτό διατυπώσαμε έτσι τον κατάλογο. Είναι φυσικά σαφές ότι ο πέμπτος κατάλογος ήταν πολύ διαφορετικός. Δύο χρόνια μετά από την Πράσινη Συμφωνία, η εφορία θα είναι κριτήριο για την υλοποίηση κάθε προγράμματος. Μαζί με το κόστος. Πρέπει κάθε έργο να είναι επιλέξιμο από την άποψη αυτή. Έτσι, το περιβάλλον θα έχει το δικό του λόγο στην επιλογή των έργων, περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Προσβλέπω σε συνεργασία στο μέλλον για να ελοπίσουμε το κοινό μας όραμα για έναν πιο σύγχρονο κανονισμό TEN ή για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, για περισσότερη ασφάλεια, για καλύτερο εφοδιασμό, για πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η κοινή συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία σχετικά με την αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 του κανονισμού σχετικά με τον Ενωσιακό Κατάλογο Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος θα διεξαχθεί την Τετάρτη. Η ψηφοφορία για την περάτωση της συζήτηση των προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή ε, θα διεξαχθεί κατά την περίοδο Συνόδου του Μαρτίου. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι αγορεύσεις διαρκείας ενός λεπτού, σύμφωνα με το άρθρο 172 του κανονισμού. Θα ήθελα, επειδή έχουμε ένα μακρύ κατάλογο, σχεδόν 30 ομιλητών, να ζητήσω από όλους να είναι αυστηρά συνεπείς στο χρόνο του ενός λεπτού και να ευχαριστήσω προκαταβολικά εξ ονόματος όλων τους διερμηνείς που θα χρειαστεί για ένα χρονικό διάστημα πέραν του προγραμματισμένου να μας βοηθήσουν για να ολοκληρώσουμε την απόψινή συνεδρίαση. Το λόγο έχει ο κύριος Σόκολ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες είδαμε την αρχή ενός ευρωπαϊκού εγχειρήματο καταπολέμησης του καρκίνου. Ακούσαμε πολλές μαρτυρίες, ακούσαμε πόσα πολλά μπορεί να κάνει η Ευρώπη για αυτό το πράγμα. Ελπίζω να μην μείνουμε εκεί. Υπάρχουν πολλά μέσα αριθμιστικά που διαθέτει η Ένωση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην καταπολέμηση του καρκίνου. Ένα βασικό θέμα είναι η διαφορετική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας ε, στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ Νότιας Ευρώπης και Ανατολικής Ευρώπης και Βόρειας και Βορειοδυτικής Ευρώπης από την άλλη. Θέλω να καλέσω λοιπόν την Κομισιόν να επενδύσει στην ανάπτυξη ε, κέντρων αριστείας για την καταπολέμηση και τη θεραπεία του καρκίνου, ώστε να έχουμε το ίδιο επίπεδο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Μαροκό είναι εταίρος προτεραιότητος και όσον αφορά επίσης τα Κανάρια αλλά και την Ισπανία γείτον χώρα. Με τίποτα δεν θα πρέπει μονόπλευρα το Μαροκό να ορίσει τι όρια θα υπάρχουν στα ύδατα του Ατλαντικού εκεί που βρίσκονται τα Κανάρια νησιά, γιατί αυτά είναι η κυριαρχία της Ισπανίας. Πρέπει αυτό να ρυθμιστεί θυμερός. Πρόκειται για καταπάτηση του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Πρόκειται για παραβίαση των συνόρων ενός κράτους μέλους. Χλιαρές αντιδράσεις δεν χωρούν εδώ. Θα πρέπει ενεργά να φρενάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις μονομερείς ενέργειες του Μαρόκο. Και επίση, μεταξύ Λονδίνου και Ραμπάτ υπάρχουν συμφωνίες σε σχέση με την ντομάτα, αλλά αυτά θα τα πούμε ε, λίαν προσεχώς. Πάντως, σε αυτή μου την πρώτη παρέμβαση απαιτώ και για τα δύο θέματα που σας ανέφερα. το λόγο έχει ο Μπασέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τις τελευταίες μέρες έχω την αίσθηση ότι αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο από όλα τα άλλα είναι η αλληλεγγύη. Η τεχνολογία 5G μας δίνει την ευκαιρία να επιδειχθεί κάποια αλληλεγγύη. Και γιατί αυτό. Διότι δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να υπάρξει ρύθμιση ομοιόμορφη για όλα τα κρατημέλη όσον αφορά αυτήν την τεχνολογία και όλα τα σχετικά προϊόντα με θεσπίσει κάποιους κανόνες και κάποια πρότυπα πανευρωπαϊκής ισχύω. Είμαι πεπισμένος. Έτσι θα βελτιώσουμε τη συνοχή. Πολτσακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να μιλήσω για την πολιτική συνοχής που είναι κέρια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αναντικατάστατη ε, για πολλά κράτη-μέλη. Καταρχήν το νόημα της πολιτικής συνοχής. Ε, ο σκοπός ε, είναι να απαλείψει τις μειονεκτικές περιοχές, τις αδύναμες περιοχές. Και για τα νέα κράτη-μέλη αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουν ανταποκριθεί στα πρότυπα που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, τώρα η υποστήριξη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτά. Η πολιτική συνοχής δεν πρέπει να αποδυναμωθεί. Δυστυχώς όμως το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο ε, δεν την προωθεί όπως πρέπει και αυτό μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Ε, αν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι όπως το Brexit και λοιπά, να το καταλάβω. Αλλά αυτή την... πρόσπιση για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ενημερώσω τους συναδέλφους και την Κομισιόν ότι η Τσεχική Γερουσία δέχθηκε ένα νέο νομοσχέδιο, νομοσχέδιο του ποινικού κώδικα Ε, όπου οι ποινές έγιναν πιο αυστηρές προκειμένου περί βασανισμού ζώων. Και κατά τις συζητήσεις στο Κοινοβούλιο και στην κοινή γνώμη φάνηκε ότι το θέμα αυτό είναι πανευρωπαϊκό θέμα και οι χώρες δεν μπορούν να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα ζώα, τα οποία κατά δεκάδες χιλιάδες ε, μεταφέρονται κάτω από παράδεκτες συνθήκες από τα λεγόμενα νέα κράτη-μέλη στα λεγόμενα παλιά κράτη-μέλη. Πρόκειται κυρίως για κατοικίδια ζώα. Ε, είναι, μπορεί να φαίνεται ε, περιθωριακό το θέμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Συνεπάγεται και φοροδιαφυγή. Πρέπει η Κομισιόν να το πάρει στα σοβαρά και να το καταπιαστεί. Και καλό την Κομισιόν να... Το λόγο, για ένα λεπτό. Ε, Κύριε Πρόεδρε, αυτή η θητεία θα είναι η θητεία της ε, δίκαιης τεχνολογικής μετάβασης και της πράσινης συμφωνίας. Όμως θα πρέπει να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι. Εντάξει, καλά είναι τα λόγια, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο όσον αφορά την πρακτική πλευρά για την βιώσιμη ανάπτυξη, για την ε, δίκαιη μετάβαση. Αυτά τα ταμεία χρειάζονται πρικοδότηση. Άρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε επομένως τη δομή αυτών των ε, οργάνων ε, και, ε, και τις αρμοδιότητες τις σχετικές. Άρα χρειάζεται μια στροφή, ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι, ξέρουμε τις προκλήσεις, όμως χρειάζονται, χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια, περισσότερο χρήμα και κυρίως ένας καινούριο περιβαλλοντικός φόρος. Χάισελ, για ένα λεπτό. Ďakujem για να διασφαλίσουμε την δίκαιη μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία πρέπει να φροντίσουμε τη δίκαιη μετάβαση για όλους. Δεν θα πρέπει να πληρώσουν οι πιο ευάλωτοι και δύο φορές επειδή δεν θα λάβουν ε, από την Ένωση τίποτα και από την άλλη θα αυξηθούν οι τιμές ενέργειας, πρέπει να βεβαιωθούν ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Ε, έχουμε εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μηχανισμούς, ε, έχουμε το Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση για παράδειγμα, αλλά πρέπει να φροντίσουμε ώστε τα κονδύλια αυτού του ταμείου θα πάει εκεί που χρειάζονται περισσότερο, δηλαδή στις περιφέρειες που επηρεάζονται και πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση αυτή. Τι περιφέρειες που χρειάζονται περισσότερο τα κονδύλια αυτά. Να φροντίσουμε, να βοηθήσουμε ουσιαστικά τι περιφέρειες αυτέ και τι χώρε του. Ε, τα, σχέδια θα πρέπει να υποβάλλονται με τρόπο... Λόγο έχει κυρία για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης. Το Horizon άρχονται νέες δεξιότητες για διαφορετικούς κλάδους. Όσον αφορά την έρευνα πρέπει αυτές οι δεξιότητες να περάσουν μέσα από την παιδεία και τα κρατημέλη να μπορούν να κάνουν όσο μπορούν καλύτερη έρευνα για την καινοτομία. Ε, στον χώρο της δουλειάς να περάσουν και στην αγορά απασχόλησης αυτές οι δεξιότητες να συνεργαστούν οι εταιρείε που ε, κάνουν ε, έρευνα στην Μαδέρα που είναι εξώγος από κεντρή περιφέρεια θα πρέπει να γεφυρώσουμε το χάσμα με το παρελθόν να δώσουμε καινούργιες δυνατότητες και έτσι να γίνει μια πραγματική αλλαγή και να γίνουμε πρωτο, πρωτοπόροι σε αυτό. Πρόεδρε, 6 και 7 Φεβρουαρίου στο Σεν Μαρτέν της Γαλλίας είχαμε την 24η διάσκεψη των εξόχως ε, αποκέντρων ε, περιφερειών της Ευρώπης. Τι είναι, πρόκειται για μακρινές ε, περιοχές εκτός ε, της εθνικής ε, επικράτειας. Ε, Παρ' όλα αυτά όμως, στο πρωτογενές άρθρο, στο 149 άρθρο, κατονομάζονται με συγκεκριμένο τρόπο. Πρόκειται επομένως κάτι το οποίο στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτό που να πει συνοχή, συνοχή γεωγραφική, κοινωνική, θα πρέπει να καλυφθούν από το πολιτές δημοσιογικό πλαίσιο. Να μην υπάρχει εξίσωση προς τα κάτω. Το πρόβλημα τους είναι η γεωργία, η συνοχή και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Θα πρέπει επιμένως αυτές οι περιφέρειες να συνεχίσουν να απολαμβάνουν το 85% συγχρηματοδότησης. Ε, από πλευρά ενεργειακής έχουν ιδιομορφίε, είναι ευάλωτες. Επίσης ε, έχουν και θέμα με την μετανάστευση. Έτσι θα πρέπει να μείνουν ζωντανές αυτές οι περιοχές. Θα πρέπει να τιμήσουμε τις δεσμές μας προς αυτούς τους ανθρώπους. Το λόγο έχει ο κύριος Μπενέα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Να σκεφτούμε ότι δεν χρειαζόμαστε λύσεις μεταφορών ευφυής, αλλά και βιώσιμες και βιώσιμους δρόμους που θα ε, κατασκευάζονται λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον. Και ε, πρόκειται και για προστατευόμενες περιοχές. Υπάρχουν μεγάλες υποδομές, ε, σε εμά υπάρχει ένας μεγάλος αυτοκινητόδρομος για παράδειγμα και άλλα έργα στην βορειοανατολική περιοχή, στη Ρουμανία αυτή είναι μία από τις φτωχότερες περιοχές. Και επίσης πρόκειται και για προστατευμένες περιοχές. Ε, σίγουρα οι υποδομές δεν πρέπει να, τα έργα δηλαδή δεν πρέπει να εμποδιστούν. Ο αυτοκινητόδρομος της Μολδαβίας είναι πολύ σημαντικό έργο. Νομίζω ότι θα πρέπει να προτιμήσουμε το, ε, ένα άλλο έργο ε, στην Τρανσυλβανία και στη Μολδαβία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν αρκετού μήνε πήραμε την απόφαση ως Ευρωπαϊκή Ένωση για επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία λόγω των παράνομων επεμβάσεων τη στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και ενώ περιμένουμε ακόμη τα μέτρα, η Τουρκία συμφώνησε με το καθεστώς της Τρίπολης σε διαμοιρασμό τη θάλασσα μεταξύ του πράγμα που κρίθηκε ήδη από την ευρωπαϊκή ένωση ως εντελώς νομικά αβάσιμο και άκυρο. τις προάλλες η τουρκία ανακοίνωσε νέες παράνομες ενέργειες σε όλη την ανατολική μεσόγειο και διαρωτώ με αυτή είναι η αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής ένωσης να επιβάλλει μέτρα και κυρώσεις σε ένα τέτοιο αρπακτικό κράτος που είναι η τουρκία; αυτή είναι η αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής ένωσης να προασπιστεί τα δικά της συμφέροντα και το διεθνές δίκαιο. θεωρώ λοιπόν ότι όπως το έθεσε και ο κύριος μπορέλ το ζήτημα είναι θέμα απλώς εφαρμογής του διεθνούς δικαίου και η ευρωπαϊκή ένωση οφείλει να βρει τους τρόπους να προασπιστεί τα ίδια τα συμφέροντά της. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η απόφαση μπορεί να σώσει εκατομμύρια ανθρώπους. Υπάρχει στη Ρουμανία ένα ίδρυμα, ε, το Ινστιτούτο Κοζινό, που ε, ασχολείται με το νιό της γρήπης και την αντοχή ε, στα αντιβιωτικά πρέπει να προωθήσουμε τις προτεραιότητες των στρατηγικών μας στόχων. Υπάρχουν επίσης μέτρα που έλαβε το Ρουμανικό Κοινοβούλιο. Για να εφαρμοστούν όλα αυτά αποτελεσματικά πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκό σχέδιο, στρατηγικός στόχος ευρύτερος. Έτσι θα φροντίσουμε για φθηνότερα και αποτελεσματικότερα εμβόλια μεταξύ άλλων. Αυτό το Ίδρυμα ανήκει σε ε, ένα ονόμιλο από τα 7 που κάνουν εμβόλια κατά της γρήπης. Πρέπει να προωθήσουμε την ανοσία και πολλά άλλα. Ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης τώρα με τον κορονοϊό πρέπει να έχουμε έγκαιρες διαγνώσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο τομέας της υγείας... Για ένα λεπτό. Λέμε πολλά για τη νέα πράσινη συμφωνία ως στρατηγική για κλιματική ουδετερότητα, προς του περιβάλλοντος, βιοπικιλότητα και ευημερία η ΚΑΠ θα καλυφθεί και αυτή. Θα πρέπει να γίνει βιώσιμη από κάθε άποψη, να εξασφαλίσει την επιβίωση στην ε, Ήπεθρο για αγρότες και για όλο τον κόσμο στην ε, Ήπεθρο. Η βιωσιμότητα είναι το κλειδί για να πετύχει η Πράσινη Συμφωνία. Αλλά θα πρέπει οι γεωργοί για ίδια δουλειά να έχουν ίδια εισόδημα. Στη Λιθουανία ε, αυτά θέλει ο κόσμος, θέλει διατροφική ασφάλεια, ε, πλαισίωση της μεταχείρισης των ζώων, για να φτάσουμε στον επιθυμητό μέσο όρο. Η νέα πρώτη συμφωνία είναι ιστορική ευκαιρία. θέλουμε να σώσουμε τον πλανήτη και καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί δίκαιη εφαρμογή τη συμφωνία για όλου του γεωργού και επίση να έχουμε άμεσε πληρωμέ. Ευχαριστώ. μετά το Brexit ε, μπαίνουμε σε πολύ σημαντική εποχή. Χάνουμε ένα σημαντικό κράτος μέλος. Αλλά θα πρέπει να δούμε τη μελλοντική μας συνεργασία στο μέλλον προς το συμφέρον όλων ε, και προς το συμφέρον των τριών εκατομμυρίων Ευρωπαίων που ζουν εκεί. Ε, υπάρχουν διάφοροι, διάφορες μορφές επηρεασμού. Ε, θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προασπίσει τα συμφέροντα των ανθρώπων αυτών για να προχωρήσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα, να αναζωογονηθεί. Χρειαζόμαστε ε, νομικές εγγυήσει, ένα συγκεκριμένο καθεστώς δεν μπορούν να γίνουν διαφοροποίησεις πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε την ίση μεταχείριση πολύ σημαντικό αυτό για τους πολίτες και στη Ρουμανία Υπάρχει μια αναφορά 10.000 ε, ανθρώπων ε, που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικό και προς αυτή την κατεύθυνση ε, θα πρέπει να δούμε και την ηθαγένεια της Ένωσης. Ευχαριστώ. <clears throat> Κυρίες και κύριοι, στα Δυτικά Βαλκάνια υπάρχουν και άνθρωποι, όχι μόνο γεωπολιτικά συμφέροντα, ε, στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη είναι πολύ σημαντικές οι εκλογές στο Μόσταρ. Υπάρχουν εδώ πολιτικοί αποκλεισμοί. Από το 2008 δεν έχουν γίνει ε, ε, εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπάρχει ένας δήμαρχος ο οποίος είναι τελείως απονομιμοποιημένος. Οι κάτοικοι του Μόσταρ είπαν λοιπόν, προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, για αυτό το θέμα. Αυτό, το, αυτή η κατάσταση παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν να γίνουν αλλαγές. Το Μόσταρ είναι όμως μια ιδιαίτερη πόλη. Υπάρχουν ακόμα ε, οι πληγές των Βαλκανικών πολέμων. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βοηθήσει τους κατοίκους του Μόσταρ και να επιτρέψει στην πόλη αυτή να διοργανώσει τις εκλογές αυτές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό θα είναι ένα συγκεκριμένο βήμα προς τον εκδημοκρατισμό της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Και έτσι η Βοσνία και Ερζεγοβίνη θα μπορέσει να προσεγγίσει ευρωπαϊκές αξίες. Το λόγο έχει ο κύριος Στεφανούτα. Κύριε Πρόεδρε, Δεν εκπλήσει το γεγονός ότι ε, πολλές κυβερνητικές οργανώσεις ε, ενδιαφέρονται για τα δάση στη Ρουμανία, που είναι πολλά. Ε, είναι πολύ σημαντικό να διατηρούν το καθεστώς προστασίας. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να φροντίσουν το δάσος και το αγαπούν το δάσος αυτό. Γιατί τους δημιουργούμε προβλήματα το 1 τρίτον των ε, προστατευόμενων περιοχών Natura ε, έχουν πληγεί από πρόσφατα μέτρα και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις δεν διαθέτουν ε, το απαραίτητο προσωπικό ούτε τα απαραίτητα κονδύλια για να αμυνθούν. Τι νόημα έχει λοιπόν το Natura αν δεν επιτρέπουμε ε, στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, να βοηθηθούν από τους πολίτες. Τα δάση της Ρουμανίας είναι ευρωπαϊκά δάση και ο, ο αέρας... Το λόγο έχει ο κύριος Μπαουζάντιας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο οίκος της ελευθερίας. Την περασμένη εβδομάδα κάλεσα ο το ηγέτες της αντιπολίτευσης της Κούβας να εδώ και να μας εξηγήσουν ακριβώς τι γίνεται, τι περνάνε, τι κάνει ο Διέθ Κανέλ, ο δικτάτορας στην Κούβα. Όμως, όταν κάποιος έχει να κάνει με δικτατορίες, πρέπει να αντιμετωπίσει αυτούς. Και το καθεστώς ε, απαγόρευσε στους ε, πέντε να έρθουν εδώ. Δεν μπορούσαν να έρθουν Τρει ήρθαν γιατί μένουν στην εξορία, οπότε μπόρεσαν αυτοί οι τρεις να έρθουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως, πάρα αυτό, πάρα αυτά, ε, το πρόβλημα ήταν ότι ήρθαν κάποιοι εδώ ε, ε, οι οποίοι ήταν βαλτοί από το Κοινοβούλιο για να προπυλακίσουν αυτούς τους κουβανούς της αντιπολίτευσης. Και η Γκουε, υποδέμος δηλαδή της Ισπανίας, επέτρεψαν σε αυτούς τους ε, ε, εντελωμένους του καθεστώτος να έρθουν εδώ για τον προπυλακισμό. Ας ξέρουν οι δικτάτορες ότι όσο καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, διακόπτει. Ne gre več z manj. Veste, nisem dolgo v politiki, vendar dobro vem, da gre vsa politika skozi sredstva, eh, skozi denar namenjen financiranju. Ξέρω ότι πάντα οι πολιτικές συνδέονται με χρήματα. Ο προϋπολογισμός δεν ε, θα περιοριστεί ε, στην επόμενη ε, επταετία, αλλά θα θέσει τις βάσεις και για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε τα απαραίτητα έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης ε, στο επίπεδο της ε, πολιτικής ε, συνοχής δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αυτό όμως θα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να καλύψουμε όλες τις περιφέρειες που έχουν ανάγκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσει διότι αριθμό, τον αριθμό των έργων και την αλληλεγγύη. Ε, η συνοχή γι' αυτό χρειάζεται. Εμείς χρειαζόμαστε περισσότερα αν θέλουμε να πετύχουμε περισσότερα. Το λόγο έχει ο κύριος Ρουζέ. Για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Γουαδελούπη, η Γουιάννα, η Ρουινιόν, η Μαγιόρκη, ο Σαμαρτά, οι περιοχές Ρουίπ, όπως τις λέμε, δεν μπορούν να θυσιαστούν στο βωμό της μελλοντική γεωργικής πολιτικής. Το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να μειώσει κατά 3,9% τον προπολογισμό για τις επιλογές για αυτές τις περιοχές. Πρόκειται για απομακρυσμένες περιοχές οι οποίες φροντίζουν για το ζαχαροκάλαμο, τις μπανάνες, το ρούμι υπέρ των Ευρωπαίων καταναλωτών. Πρέπει να τις στηρίξουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν να μειώσουμε τα κονδύλια αυτά. Αφήστε που από αυτό εξαρτάται η ευημερία των ε, γεωργών μας. Πρόκειται για μια ειδική κατάσταση. Γι' αυτόν τον λόγο, μαζί με την Μαρίν Λεπέν και το κόμμα Rassemblement National, ζητούμε να αυξηθεί ο τρέχον προπολογισμό για τα κονδύλια αυτά. Ευχαριστώ πολύ. για ένα λεπτό. Monsieur le Président. Οι χώρες, όπως ξέρουμε, αναλαμβάνουν για έξι μήνε την Προεδρία με την υποστήριξη ιδιωτικών εταιριών. Σκανδαλώδες. Αυτό πλήττει την αντικειμενικότητα των κυβερνήσεων. Αυτό έκανε η Ρουμανία, είχε την υποστήριξη της Coca-Cola. Αυτή η αμερικανική πολυεθνική έδωσε 40 εκατομμύρια και απέκτησε το δικαίωμα να προσκαλεί τους δικούς τη προσκεκλημένους εκδηλώσεις της Ρουμανικής Προεδρίας. Ανακατεύονται λοιπόν ιδιωτικά με δημόσια συμφέροντα. Φέτο η Κροατία είπε να κάνει κάτι καλύτερο, απέτυχε, διότι την υποστηρίζει η ΙΝΑ, μια πετρελαϊκή εταιρεία. Θα λέγαμε ότι δεν πηγαίνουμε καλά. Έχει καμία σχέση με την πράσινη συμφωνία της Επιτροπής Φοντερ Λάιεν. Πρέπει λοιπόν να σημάνουμε συναγερμό και να απαγορεύσουμε τα sponsoring, τις χορηγίες των προεδριών. Μην δούμε σε λίγο την ε, BMW να υποστηρίζει τη Γερμανία και η Τραπέζα τη Γαλλία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τις ε, προηγούμενε μέρε είχαμε αυτή την επιστολή σα όλοι και εγώ και άλλοι 35 Ιταλοί υπογράψαμε ότι σήμερα στις 10 Δευτέρου με το που θα αρχίσει η Ολομέλεια θα, θα θυμηθούμε τις 30 περίπου και που κατέληξαν σε κάποια πηγάδια στην Ίστρια και 300.000 πρόσφυγες. Ήταν αυτό ένα μήνυμα για την μνήμη τους και θα πρέπει και σε αυτή την ε, ευκαιρία, με αυτή την επέτειο να θυμηθούμε ε, τις ευθύνες των Ιουγκοσλάβων παρτιζάνων του ε, Τίτο και κάποιων παρτιζάνων Ιταλών. γίναν οι Ιταλοί πρόσφυγες ή σκοτώθηκαν. Αλλά από ποιον και για ποιο λόγο θέλουν να φύγουν από ποιον. Αυτού του είδους η άρνηση θα πρέπει να καταπολεμηθεί με την ιστορική αλήθεια ε, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ειρήνη αν έχουμε χωρίσει τα θύματα σε πρώτη ή δεύτερη κατηγορία. Mr. Wallace. You didn't ask the floor. You are written here. President, I wasn't told about it. What's the topic? Για ποιο θέμα λέτε, λέει ο κ. Wallace. Μιλούμε για τις ΗΠΑ Πολιτείες και οι παρατυπίες ε, που έγιναν στην Αϊόβα. Θα μιλήσω η αδελφό μου. Αλλά μια που μου δίνεται ευκαιρία να χρησιμοποιήσω το λεπτό. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκλογική διαδικασία στην Ιλλανδία. Τα νέο τα Φέλ και Φιναγκέλ, τα δύο νεοφιλελεύθερα κόμματα προκάλεσαν μεγάλη αναταραχή. Ο κόσμος ε, αντέδρασε στην αδικία με την οποία διακυβερνάται η χώρα. Η ανάκαμψη, η υποτιθέμενη ανάκαμψη, έφυσε πίσω τις πολλούς στοχούς. Η κυβέρνηση δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τα σημαντικά προβλήματα που πλήττουν τον πληθυσμό. Έχουμε αστέγους, έχουμε ανθρώπους που δεν μπορούν να βρουν σπίτι και δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Διασώσαμε τις τράπεζες. Δεν στείλαμε δισεκατομμύρια προς τούτο. Και φορτώσαμε τα δισεκατομμύρια αυτά στους ώμους φτωχών ανθρώπων. Και τώρα τα σπίτια του κόσμου περνούν στα χέρια των τραπεζών ξανά και δεν κουνιέται φίλο. Έχουμε πολλά προβλήματα. Ελπίζω ότι στι ε, προσεχείς εκλογέ αυτήν την εβδομάδα κάτι θα κάνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και τώρα η κυρία Ντέιλι για το θέμα που προανέφερα. Thanks, Το Κοινοβούλιο είχαν ευκαιρία να δίνει μαθήματα σε άλλες χώρες ε, ή να μιλήσει για εμπλοκή σε εκλογικέ διαδικασίε κλπ. Ο Μπέρνι Σάντερ είναι ο πρώτος τις δημοσκοπήσεις αν και ξέρουμε ότι πολλοί δημοκρατικοί δεν τον πάνε τι έγινε λοιπόν το σύστημα στην ΑΙΟΒΑ το δημιούργησε μια εταιρεία την οποία χρηματοδοτήσει η αντίπαλη. Ο κ. Μπέλτερ λοιπόν ε, βγαίνει, ανακοινώνει τον εαυτό του ως νικητή. Ε, αυτά, αυτά συμβαίνουν στις ΗΠΑ Βασιλεύει η τηλεόραση. Νομίζω ότι θα έπρεπε να καταδικάσουμε αυτή την ε, υπόθεση, αλλά η η Αμερική μάλλον είναι πολύ μεγάλη και γι' αυτό σιωπούμε. Είναι μια μαύρη μέρα. Πρόκειται για ε, ένα περιστατικό το οποίο γελιοποιεί τη δημοκρατία. Δεν μπορούμε να μην το σχολιάσουμε. Το λόγο έχει ο κύριος Νικολάου Αλαβάνος για ένα λεπτό. Στις 18 Φλεβάρι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα απεργούν ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που διαλύει περαιτέρω την κοινωνική ασφάλιση με συνέπεια η πλειοψηφία των σημερινών εργαζομένων να πάρει λιγότερα από 450 ευρώ σύνταξη. κατοχυρώνονται οι μειώσεις της προηγούμενης κυβέρνησης του σύριζα διατηρούνται τα αυξημένα όρια συνταξιοδότησης και η εγγυημένη εθνική σύνταξη φτώχειας των 384 ευρώ. ανοίγεται ο δρόμος για να τζογάρονται τα αποθεματικά σε επενδυτικά προϊόντα υψηλού ρίσκου με την ιδιωτικοποίηση την εξατομίκευση τι περικοπέ υπάρχει ο κίνδυνο να χαθούν οι κόποι μια ολόκληρη ζωή. η υπονόμευση όμω τη κοινωνική ασφάλιση είναι στρατηγική σα επιλογή. οι αναφορέ σα, περί κοινωνικών δικαιωμάτων είναι μεγάλο ψέμα. ανάλογα αντεργατικά σχέδια προωθούνται σε γαλλία βέλγιο και αλλού όπου οι εργαζόμενοι απαντούν αγωνιστικά. με το βλέμμα στραμμένο στη νέα ύφεση που έρχεται διευκολύνετε του εργοδότε, μειώνοντα τι ασφαλιστικέ εισφορέ, ανοίγετε μια αγορά δισεκατομμυρίων για τα κέρδη των ασφαλιστικών μονοπωλίων του μοιράζετε ζεστό χρήμα με την πάλη του εργαζόμενοι και αυταπασχολούμενοι θα ανατρέψουν τα σχέδια ευρωπαϊκής ένωσης κυβερνήσεων απαιτώντας κοινωνική ασφάλιση με ευθύνη του κράτους με δωρεάν υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Ευχαριστώ. Ο κύριος για Ευχαριστώ. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για μία χώρα. Μία χώρα όχι μακρινή, μία χώρα της ανατολικής γειτονικής σχέσης. Ε, έχουμε 24 γλώσσες επίσημες εδώ, αλλά στο Κίεβο αυτό δεν ωφελεί. Ε, και υπάρχει ένας νόμος του 17 για την παιδεία και απαγορεύεται οι μειονότητες να χρησιμοποιούν στο σχολείο την μητρική τους γλώσσα. οι συνέπειε είναι πολύ σοβαρές. Η ρουμανική μειονότητα στην Ουκρανία αντιμετωπίζει μία πραγματικότητα πραγματικά σοβιετική. Είναι κάτι σαν ξένη γλώσσα για τους Ρουμάνους της Ουκρανίας, τα ρουμανικά. Ε, αυτό που λέμε μολδαβικά και ε, μιλούμε για 150.000 Ρουμάνους έχουν τη ρουμανική ηθαγένεια μιλούν ρουμανικά και... Ε, Δόθηκε η διαδικασία των ομιλιών του ενός λεπτού με βάση το άρθρο 172 του κανονισμού. Η επόμενη συνεδρίαση θα διεξαχθεί αύριο, Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου, από τις 9 έως τις 12.30 και από τις 15 έως τις 23. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συνεδρίαση έληξε. Ευχαριστούμε τους διερμηνείς.